Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε τη συνέδρια. Έχουμε για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της ε, ε, Ουγγρικής Προεδρίας τον κύριο Τωμά Φελεγγύη, που είναι μεταξύ, μεταξύ άλλων αρμόδιο και για την ε, περιφερειακή πολιτική. Τον ευχαριστούμε θερμά για την ε, παρουσία του εδώ Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, tisztelt elnök asszony! Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, καλημέρα σα, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εδώ παρόντε, ή ε, μέσω του ίντερνετ ε, ακροατές, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη συνεδρία, να σας ευχαριστώ για την υποδοχή και να σας αναφέρω τι έχουμε στο πρόγραμμά μας για το επόμενο διάστημα. Όπως είχαμε συμφωνήσει τον ε, Ιανουάριο, τουλάχιστον εγώ αυτό αντελήφθη κατόπιν των ε, συζητήσεων μας στη συνεδρία εκείνης. Όπως λοιπόν είχαμε συμφωνήσει, θα πραγματοποιούνταν μια άλλη συνεδρίαση για να σας ε, παρουσιάσω τα της προόδου στα πολιτικά ζητήματα και να σας εξηγήσω τι άλλα σχέδια έχουμε για το μέλλον. Προφανώς στην απαρχή αυτή της νέας ε, περίοδου που βρισκόμαστε καθίσατε σαφές ότι χρειάζεται επιπλέον ανάπτυξη της ε, πολιτικής συνοχής για να μπορέσει η Ευρώπη να αναλάβει το ρόλο που της ανήκει ως παγκόσμιος παράγων και γι' αυτό θα πρέπει να καταστεί πιο αποτελεσματική η πολιτική συνοχή από ό,τι μέχρι τώρα για να βοηθήσει τις χώρες να καλύψουν χαμένο έδαφος, να προχωρήσουν πιο γρήγορα, να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα. Με έναν μόνο τρόπο μπορεί η Ευρώπη να αποδειχθεί επιτυχής, δηλαδή μόνο αν λαμβάνει υπόψη με αποτελεσματικές στρατηγικές που θα εφαρμόζει τις ιδιαιτερότητες το εις κάθε περιφερειάς της. Αυτό πάντοτε πρέπει να το έχουμε υπόψη όταν χαράσουμε στρατηγική, όταν ε, ε, σχεδιάζουμε ή εφαρμόζουμε προγράμματα ή όταν ε, παρακολουθούμε τον τρόπο υλοποίησής τους. Έτσι λοιπόν τόσο η στρατηγική του 2020 όσο και η πολιτική συνοχής απαιτούν να λαμβάνονται πάντα υπόψη οι περιφερειακές εταιρότητες. Εμείς θέλουμε μια πρόοδο ουσιαστική ως Ουγγρική Προεδρία στο τομέα αυτών με την αναθεώρηση της, ε, της ατζέντα ε, για την περιφερειακή ε, ανάπτυξη που είναι κομμάτι της ατζέντα του 2020 σε συμφωνία με την Επιτροπή γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό θα συνεχίσουμε τη συνεργασία λαμβανωμένων υπόψη των πτυχών της, ε, των ιδιαιτεροτήτων των περιφερειών στην πολιτική συνοχή. ένα δε χαρακτηριστικό, μια ανάγκη της πολιτικής συνοχής είναι ότι πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση για, και να αντικοποιηθούν οι προτάσεις για το μέλλον της πολιτικής συνοχής και θέλουμε ε, να στηρίξουμε εμείς αυτή τη διαδικασία έτσι ώστε οι προτάσεις ε, που υπάρχουν και στο, στην έκθεση για τη συνοχή να υλοποιηθούν με απτά μέτρα τα οποία θα βρίσκουν σύμφωνα όλα τα κράτη-μέλη. Έτσι λοιπόν θέλουμε μια πολιτική η οποία θα εστιάζεται στους στόχους ε, της στρατηγικής του 2020 και την αλληλεγγύη μια πολιτική που θα είναι στραμμένη προς τα αποτελέσματα, που θα είναι οικονομική, θα ε, στο δυνατόν με λιγότερη γραφειοκρατία και θα ε, στο δυνατόν περισσότερους δικαιούχους. Επιτρέψτε μου λοιπόν ε, να σας παρουσιάσω κάποιες βασικές αρχές της ε, πολιτικής της Προεδρίας μας. Έχουμε προετοιμάσει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων ε, της 21 Φεβρουαρίου του 2011 με στόχο πρώτον να ανταποκριθούμε στα επιχειρήματα της εκθέσεως για την πολιτική συνοχής. Δεύτερον, να ορίσουμε συνοπτικά τους τομείς στους οποίους θα πρέπει να προχωρήσουμε σε συνενετικές ε, προτάσεις συμπεράσματα δηλαδή στα οποία καταγράφονται όλοι οι τομεί στου οποίου συμφωνούν τα κράτη-μέλη. Και είναι τα εξή. Οι εξή. Ε, συμφωνούν τα κράτη-μέλη ότι η πολιτική συνοχή είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για την πολιτική τη ενσωμάτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει συμβάλει τα μάλα έτσι ώστε να ε, απαλληφθούν ε, στο βαθμό του δυνατού οι διαφορέ μεταξύ των περιφερειών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη-μέλη δύο θα θέλανε να αποφύγουν την υπονόμευση των στόχων ε, της περιφερειακής ανάπτυξης και της στρατηγικής του 2020 ε, και έτσι όταν εφαρμόζονται οι στόχοι αυτοί, είτε πρόκειται για την περιφερειακή πολιτική είτε για τη στρατηγική του 2020, δεν θα έπρεπε να προξενούν προβλήματα στην εφαρμογή ημέν των ΔΕ, να υπονομεύουν ημέν των ΔΕ. Ε, θα πρέπει να λαμβάνουμε πάντα υπόψη την τοπική περιφερειακή ιδιαιτερότητα της ε, τοπικές ιδιαιτερότητες, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει η πολιτική της συνοχής να έχει και ε, προσέγγιση που θα επιτρέπει την ολοκλήρωση, την ενσωμάτωση δηλαδή. Στα συμπεράσματα επίσης καταγράφουν τα κράτη-μέλη την ανάγκη για μια διαφανή, σαφή, για ένα σαφές διαφανές ε, ρυθμιστικό πλαίσιο και υπογραμμίζουν ταυτόχρονα το γεγονός ότι θα πρέπει η υλοποίηση αυτού να είναι και πιο αποτελεσματική και πιο πολύ στραμμένη στα απτά αποτελέσματα. Στις 21 Φεβρουαρίου του 2011 έγινε λοιπόν όπως είπα μια πρώτη φορά συζήτηση στο Συμβούλιο των Υπουργών, ε, στο Συμβούλιο Υπουργενικών Υποθέσεων ε, για την πολιτική της συνοχής, δηλαδή σε πολιτικό επίπεδο συζήτηση για την πολιτική συνοχής. Όλοι υπεγράμμισαν ότι πρέπει αυτή η πολιτική να απλουστευθεί και πέραν μιας ε, ε, θεματολογικής προσέγγισης πιο συνοπτικής Είπαμε ότι θα πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση στραμμένη προς το αποτέλεσμα και προς την εξυπηρέτηση των αναγκών των περιφερειών, με ε, το δυνατόν πιο οικονομική βέβαια προσέγγιση και σχέση κόστου αποτελεσματικότητα. Ταυτόχρονα μεταξύ 29 Μαρτίου και 1 Απριλίου ε, ε, η Προεδρία μα οργάνωσε μια συνεδρίαση για τα κράτη-μέλη αλλά και για τα υποψήφια κράτη, ε, στην οποία συνεδρίαση είδαμε γενικούς διευθυντές αρμόδιους για την περιφερειακή ανάπτυξη, για την εδαφική μάλλον ανάπτυξη, οι οποίοι ε, υιοθέτησαν τα, τις προτάσεις με βάση τη στρατηγική του 2020. Η άλλη συνεδρίαση μεταξύ 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου συγκεκριμένα συζήτησε την εδαφική συνοχή, την ε, προσέγγιση ως προς τα αποτελέσματα με, με, με άξονα το με γνώμονα το αποτέλεσμα, ε, στην οποία μάλιστα συμμετείχε και η κυρία Χιούμπνερ, η πρόεδρό σα. Σημαντικό λοιπόν καθήκον, όπω βλέπετε, είναι και η έγκαιρη προετοιμασία του κανονιστικού πλαισίου των νομοθετημάτων δηλαδή, που χρειάζονται, αλλά και η εξασφάλιση κοινή θέση στα πιο σημαντικά ζητήματα. Μιλώντα από την εμπειρία που έχουμε συλλέξει, μπορώ να σα πω ότι θα χρειαστεί πάλι πολλή χρόνο μέχρι να καταλήξουμε σε κοινέ θέσει. Θα πρέπει να, χρειαστεί, ε, να εξασφαλιστεί αρκετό χρόνο και για να ε, ξεκινήσουν τα προγράμματα για την περίοδο μετά το 2014 και θα πρέπει για μια φορά να επικεντρωθούμε ιδιαίτερα στις εδαφικές πτυχές. Ε, στη διάσκεψη τη σχετική με το μέλλον της πολιτικής συνοχής, όλοι οι ε, συμμετέχοντες συμφώνησαν ως προς την ανάγκη για ευελιξία και τη σημασία το, της ε, αναγνώρισης των τοπικών ή περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες θεματικές προτεραιότητες ε, δεν θα πρέπει να συγχέονται με ε, τις κατηγορίες τις σχετικές με το, με το κόστος. Όλοι οι εκπρόσωποι συμφώνησαν ότι η προσέγγιση σχετική με τα αποτελέσματα, με γνώμη το αποτέλεσμα δηλαδή, ήταν σωστή. Θα έπρεπε όμως να υπάρξει ένα νέο σύστημα επαγωγής σε όρους και ε, υπογράμμισαν ιδιαίτερα την ανάγκη για κοινή ερμηνεία και την αναγκαιότητα να αποφευχθεί επιπλέον γραφειοκρατική επιβάρυνση. Υπόθηκε δηλαδή ότι μόνο ότι όλοι αυτοί οι νέοι όροι μπορούν να γίνουν δεκτοί μόνο εφόσον μπορεί ο συμμετέχον να ε, τους επηρεάσει και ότι θα πρέπει η προσέγγιση με βάση την ε, ε, ιδιοκτησία, ownership approach, να είναι αυτή που θα επιλεγεί εν τέλει. Εκφράστηκαν ανησυχίες επίσης ως προς τα ταμεία και τις ε, προτεραιότητες που θα οριστούν ε, ή τα κίνητρα. Οι συμμετέχοντες επίσης είπαν ότι δεν είναι καλή ιδέα τα αρνητικά ή τα αντικίνητρα, αλλά μόνο τα θετικά κίνητρα και ζήτησαν να εξασφαλιστεί η κρίσιμη εκείνη μάζα η οποία θα φέρει αποτελέσματα και αποτελεσματικότητα στην αξιοποίηση των ε, πόρων, δηλαδή να υπάρχει η ε, συνεργασία εκείνη που θα εξασφαλίσει την κρίσιμη μάζα. Επίσης μίλησαν για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση οι συμμετέχοντες και τη διατήρηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ως μέσου για την πολιτική συνοχής. Στα υπόλοιπα θέματα που έχουμε, θα ήθελα να σας αναφέρω κάποια ζητήματα τα οποία επίσης έχουν στη σε επίπεδο Συμβουλίου, ε, θεματικές ενότητες, ε, κίνητρα, προτεραιότητες, στις οποίες θα θέλαμε να ε, επικεντρωθούμε για τις επόμενες εβδομάδες. Θα θέλαμε το ταχύτερο δυνατό να έχουμε σχέδιο κανόνων για να επικεντρωθούμε στα πιο σημαντικά ζητήματα το ταχύτερο δυνατό. Και στην προσέγγιση για το έγγραφο του 2020 θα έχουμε την θεώρηση εκείνη που θα μας επιτρέπει να συνδυάσουμε την πολιτική συνοχή με την στρατηγική 2020. Στρατηγικός σχεδιασμός λοιπόν, μηχανισμοί εφαρμογής, ολοκληρωμένη προσέγγιση, ε, ανατολισμοί ήταν τα κύρια θέματα που θα έχουμε στην ημερήσια διάταξη των ε, ομάδων εργασίας του Συμβουλίου για την πολιτική συνοχή και θα θέλαμε να ακούσουμε τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς των κρατών μελών, αλλά βέβαια και από το και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβουμε πληροφορίες οι οποίες θα μας επιτρέψουν να κερδίσουμε χρόνο από τις διαπραγματεύσεις για τις ε, νομοθετικές προτάσεις. Και θα θέλαμε επίσης να συνοψίσουμε τα, τις ερωτήσεις και απαντήσεις ε, από την Επιτροπή σε ένα μόνο έγγραφο. Όλες οι θέσεις λοιπόν και οι προτάσεις που συλλέγουμε θα συμπληθούν σε ένα έγγραφο το οποίο θα εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της άτυπης συνεδρίας των Υπουργών του Γκούντουλ τις αρχές Μαΐου εφέτος για να διατυπωθούν τα συμπεράσματα της Προεδρίας με βάση αυτό. Αυτή είναι η πρόταση της ε, Ουγγρικής Προεδρίας ε, για την προετοιμασία της ε, ε, μελλοντικής πολιτική συνοχής, την οποία μετά θα συνεχίσει η Πολωνική Προεδρία. Ελπίζουμε, καθώ συμφωνούμε στις, ως προς τις αρχές, ότι θα φτάσουμε πιο κοντά ακόμη στην επιτεύξη των στόχων μας και ελπίζουμε ότι με όλη αυτή την προσπάθεια θα καταστήσουμε την, την πολιτική συνοχής πιο αποτελεσματική, μετρήσιμη, την εφαρμογή της πιο ε, απλή, τις διοικητικές διαδικασίες λιγότερο περίπλοκε. Και θέλω επίση να επισημάνω ότι παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή τι δικέ σα εργασίε και ευχαριστούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξη που έχει προσφέρει στην Ουγγρική Προεδρία στον τομέα τη πολιτική συνοχή. Μελετήσαμε την έκθεση του κυρίου Πίπερ και θα ήθελα να υπογραμμίσω το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής καλύπτει τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα της Ουγγρικής Προεδρίας σε ένα σημείο πολύ σημαντικό για μας, για την Προεδρία, ότι δηλαδή η πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ουσιαστικά εν μέρει εφαρμόζει την, ε, τους στόχους στρατηγικής του 2020 αφενός αφετέρου δε η πολιτική συνοχή θα πρέπει κατά κύριο λόγο να επικεντρώνεται στα όσα ορίζει η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε ευπρόσδεκτη αυτή την ε, τοποθέτηση. Θεωρούμε ευπρόσδεκτο το γεγονός ότι ο ε, εισηγητής υπογραμμής τη σημασία της δαφικής συνοχής και των μακροπεριφερειακών στρατηγικών ε, που αποτελούν επίσης κεντρικά σημεία της δικής μας των δικών μας επιλογών του προγράμματος Προεδρίας μας δηλαδή και κάτι ακόμη για την έκθεση του κυρίου Βλάσσα ο οποίος υπογραμμίζει την ολοκληρωμένη στρατηγική, τον ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό για την περιφερειακή πολιτική, εντοπίζοντας συγκεκριμένες περιοχές των αστικών κέντρων ή συγκεκριμένα αστικά κέντρα, που αποδεικνύουν με τον τρόπο αυτό την πολυπικιλότητα αυτής της πολιτικής. Θα ήθελα να επισημάνω λοιπόν ότι στις επόμενους, επόμενες εβδομάδες ή μήνες ε, περιμένουμε ακόμη την συμμετοχή σας σε αυτές τις προσπάθειές μας, όπως έχετε πράξει και στο παρελθόν φυσικά. Σας καλούμε και θα σας προσκαλέσουμε και σε μελλοντικέ εκδηλώσεις μας, ελπίζοντας ότι θα έχετε πάντα την ευκαιρία να συμμετέχετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Υπουργέ. Θα ήθελα να αρχίσει τώρα η συζήτηση. Μάρκους, θα ήθελες να αρχίσεις. Ja, danke, Frau. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τον Υπουργό Ήταν πολύ η τοποθέτηση του για το μέλλον της ε, διαρθρωτική πολιτικής και τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει η Ουγγρική Προεδρία να την συνοδεύσει, να την παρακολουθήσει. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο συγκεκριμένε πτυχέ. Αυτό το οποίο αναφέρατε ω ε, υπαγωγή σε όρου, conditionality. Και δεύτερον, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επωνομαζόμενη ενδιάμεση κατηγορία δηλαδή τις περιφέρειες που βρίσκονται στο επίπεδο 75-90% επί του ΑΕΠ, για την υπαγωγή. Είπατε ότι μπορείτε να δείξετε κατανόηση σε περίπτωση όπου έχουμε ε, δράσεις στις οποίες μπορούμε να επηρεάσουμε ως κράτος ε, Θα ήθελα να επισημάνω όμως ότι έχουμε μία ε, μείωση κατά 11% των ε, αναθέσεων ε, σε, δημόσιες, ε, σε δημόσιους διαγωνισμούς που μερικές φορές πέφτει και στο 9%. Είναι πάρα πολύ χαμηλό αυτό το ποσοστό. Το ίδιο ισχύει και σε σχέση με το δίκαιο του ανταγωνισμού Εάν ε, σκεφτούμε ότι ε, αναμειγνώνται όλο και περισσότερο δημόσιες επιχειρήσεις σε ιδιωτικές υποθέσεις, ιδιωτικά έργα, και γι' αυτό νομίζω ότι θα ήταν ε, καλό η Επιτροπή, και απευθύνομαι προς την Επιτροπή τώρα, να κάνει τη δουλειά της όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Ανταγωνισμού, να το προσδιορίσει κατά όρους λογικούς, ορθολογικούς, έτσι ώστε να είναι και σύμφωνα με τα όσα ισχύουν και στα κράτη-μέλη και Μόνο τότε μπορούμε να έχουμε την ε, πλήρη εκροή των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αυτό το λέω ξεκάθαρα. Και επίσης θα ήθελα να ρωτήσω σε ποιο βαθμό μπορείτε να δεχθείτε επιπλέον ε, προτάσεις στον τομέα αυτών για πρόοδο ε, ή όχι. Και κάτι άλλο για την ενδιάμεση κατηγορία. όπου η Επιτροπή λέει ότι θα μπορούσε στις περιοχές αυτές, 22 περίπου στην, ε, ε, της Ευρώπης, να δώσει ένα νέο καθεστώς υποστήριξης. Για τη Γερμανία Φερρυπίν θα ήταν το Λούνεμπουργκ, στην περιοχή δηλαδή του Αμβούργου με 80 περίπου 85% επί του ΑΕΠ και που μάκρο για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν περιοχή ε, στήριξη, την περιφέρεια στήριξη, εφόσον περάσει βέβαια αυτή η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που όμω είναι μια ευημερούσα περιφέρεια, για να μην πω πλούσια. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα στην Ευρώπη όπου διρωτόμαστε εάν έχει νόημα αυτή η δημιουργία μιας ενδιάμεσης κατηγορίας. Έστω είμαστε και στο τέλος αξιολόγηση, αλλά θα ήθελα να δω τι ε, προτάσεις έχει η ε, Προεδρία. Πώς κρίνει αυτή την πρόταση για μια ενδιάμεση ε, κατηγορία περιφέρειας. Ευχαριστώ, κύριε Φλάτσουκ. Ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό και θα μου επιτρέψει ο κύριος ε, Υπουργός να επαναλάβω μερικά πράγματα που κατά την απόψή μου είναι σημαντικά. Και νομίζω ότι αν θα βελτιωθούν τότε ακόμα περισσότερο και καλύτερα θα επηρεάσουν τα, τα, τα κονδύλια αυτά. Λοιπόν, Κατά την άποψή μου έχουμε δύο έννοιες ε, πολύ σημαντικές. Εδώ γνωρίζετε ότι εμείς τι προτείνουμε διάφορα κονδύλια να συνδυαστούν ακριβώς την ώρα της χρηματοδότησης ε, προγραμμάτων και θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση και διαφορετικά να χρησιμοποιήσουμε άλλα μέσα χρηματοδοτικά όπως το Jessica και θα πρέπει να συνεργαστούμε καλύτερα στο πλαίσιο αυτό. Το Jessica χρειάζεται να εμπλουτιστεί για να είναι ένα εργαλείο περισσότερο ανταγωνιστικό μπροστά σε άλλα προϊόντα των ε, χρηματαγορών και νομίζω ότι τα πράγματα όμως είναι αρκετά μπερδεμένα, δεν θα πρέπει να χειροτερεύσουν και να χειρότερα από ό,τι σε διάφορες τράπεζες ακόμα. Ακόμα ένα σχόλιο σχετικά με τα ιδιωτικά κονδύλια για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων. Αυτά που ονομάζονται ε, τα PPP και θα πρέπει να διευκρινίσουμε τις συνθήκες που θα πρέπει να ισχύουν για αυτά τα ιδιωτικά κονδύλια. Και εδώ χρειάζεται να δούμε τα πράγματα να μην είναι τόσο περίπλοκα τη στιγμή της χρονοποίησής τους αυτά τα σδίδε. Ευχαριστώ. Ναι, έχετε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ακριβώ επειδή κάνουμε απολογισμό της προηγούμενης πολιτικής ε, συνοχή ε, και σκεφτόμαστε να πάμε τη μελλοντική, αυτό που θεωρούμε είναι ότι αυτή η πολιτική όπω υπάρχει σήμερα ε, είναι, ήταν σημαντική ιστορικά που προσπάθησε να καλύψει ένα κενό από τι φτωχότερε περιοχέ, όπω τη Ισπανία, α πούμε και τώρα οι χώρες τη πρώην Ανατολική Ευρώπης. Αυτές αφορά κυρίως το θέμα και θα πρέπει να έχουμε απτά αποτελέσματα όσον αφορά την κάλυψη αυτής της απόστασης. Και εκεί ακριβώς δικαιολογείται η πολιτική αυτή και ε, ε, είναι επιβαλλόμενο να ισχύσει και να εφαρμοστεί. Θα πρέπει να δούμε πώς θα καταλήξουμε σε μια συνοχή, σε μια ρύθμιση ε, περιφερειακή. Κατά την άποψή μας η χρηματοδοτική αυτή η ρύθμιση χρειάζεται, συμβαίνει και επίσης εδαφική. Χρειάζεται η οικονομία της Ευρώπης να κατανεμηθεί όπως πρέπει αρμονικά, γεωγραφικά και όχι κατά προτίμηση στις περισσότερο ελκυστικές περιοχές γιατί θα έχουμε σε δύο γενιές αργότερα δηλαδή ε, θα μπουκώσουν, το πούμε έτσι, αυτές οι περιοχές και αλήθετα θα ερημώσουν άλλες περιοχές. Χρειάζεται λοιπόν αυτό το μέσο αυτής της ρύθμισης γεωγραφικής αυτή η πολιτική συνοχή ε, και γι' αυτό και η ομάδα μου ε, θα ήθελα να υποστηρίξει την ιδέα αυτή που προώθησε η Επιτροπή για ενδιάμεσες κατηγορίες ε, περιοχές και έτσι να έχουμε μια προοδοποιωτική ανάμεσα στην προηγούμενη πολιτική ώστε για ιστορικούς λόγους ω περιοχές αρκετά συχνά είχαν καθυστερήσει ιδιαίτερα να μπορέσουν να καλύψουν αυτό κενό και να είναι στραμμένη προς το μέλλον αυτή η πολιτική συνοχή με περισσότερο ομοιομορφή Ευρώπη, ομοιογένεια και να έχουμε τα κατάλληλα μέσα, τα οικονομικά, τα εργαλεία για να το πετύχουμε. Αυτές οι ενδιάμεσες περιοχές προς αυτό στρέφονται λοιπόν και γι' αυτό ακριβώ επιθυμούμε έτσι και να ληφθούν υπόψη και μάλιστα οριστικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είπατε ε, κάνατε προτάσεις τις οποίες μπορώ να δεχθώ, συμφωνώ μαζί σας, και για τη στρατηγική 2020 και την πολιτική συνοχής οι τοποθετήσει σας ε, βρίσκουν σύμφωνοι. Χαίρομαι ιδιαίτερως που κατέχει την Προεδρία η Ουγγαρία αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρουμε ότι δίνει ιδιαίτερη σημασία στην πολιτική συνοχή. Θα ακολουθήσει η Πολωνία. Πρόκειται δηλαδή για δύο κράτη, τα οποία, όπως και, ε, τα, τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά στην πατρίδα μου, τη Σλοβακία, και όχι μόνο γεωγραφικά. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι ε, θα μπορέσουμε να βρούμε όταν έρθει η ώρα λύσεις συμβαστικές σε επίπεδο Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και θα πρέπει να έχουμε και δυσκολίες όταν έρθει η ώρα για τον προϋπολογισμό ή για τον προσδορισμό των προτεραιοτήτων μας. Θα ήθελα να δω δηλαδή συγκεκριμένα η Ουγγρική Προεδρία τι θέση έχει, τι θέσεις μάλλον θα υποστηρίξει όταν έρθει η ώρα να συζητήσουμε το προσοχές δημοσιονομικό πλαίσιο. Γιατί συχνά ακούμε να γίνεται λόγος ε, για τη διάρκεια του. Θα είναι πενταετές, θα είναι επταετές. Έχετε να μου δώσετε μια απάντηση τώρα. Ο κύριος Ποστινάρου. First. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Φελεγγύη, καταρχάς ε, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει και μία νέα έννοια. Στην έκθεση Γκαρίγκα αναφέρεται αυτό το use it or lose it, δηλαδή χρησιμοποίησέ το ή απλώς το χάνεις. Τι ακριβώς όμως ε, σημαίνει αυτό, τι είναι δεσμευτικό για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεύτερον, αυτό το νέο συμβόλαιο για την ανάπτυξη, ε, τι ακριβώς θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει, τι θα είναι δεσμευτικό για τα κράτη-μέλη και τι θα είναι δεσμευτικό για τις περιφέρειες. Και τέλος, ποιο θα είναι το μήνυμα για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο σε σχέση με τους ε, υπεργολάβους. Γιατί ένας από, τις, ένας από τους λόγους της δραματικής αύξησης ε, οποιασδήποτε, οποιαδήποτε τμήματος υποδομής ε, είναι ακριβώς το ότι υπάρχει μια τεράστια λυσίδα αναδόχων ε, που αυξάνει εκθετικά τις τιμές. Τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε για να ε, προστατεύσουμε ε, και τα κονδόλια της χρηματοδότησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Κυρία ε, Τέλη, κύριε Υπουργέ, δεν αναφερθήκατε σε ένα θέμα πολύ σημαντικό για την πολιτική συνοχή, που είναι οι δείκτες. Υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή να τεθεί αυτό το ζήτημα ποιοι είναι οι υπόλοιποι δείκτες ε, σε σχέση με το ΑΠΕΠ που μπορούν να προσμετρήσουν την ευημερία των πολιτών μας. Αυτά τα κριτήρια, αυτοί οι δείκτες πρέπει οπωσδήποτε να ενσωματωθούν στα νέα προγράμματα της ε, μέλουσας πολιτικής συνοχής. Εγώ ε, προέρχομαι από τη Μητροπολιτική περιοχή του Παρουσιού, πολύ πλούσια σε ΑΕΠ, αλλά με μεγάλες κοινωνικές ανισότητες Υπάρχει, υπάρχουν προβλήματα φτώχειας, ανεργίας, πολλά προβλήματα. Και υπάρχουν επίσης και κριτήρια περιβαλλοντικά. Σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία διπλή πρόκληση. Ένα, μία πρόκληση ε, ε, κοινωνικού ε, αλλά και ένα πρόβλημα περιβαλλοντικό. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή πρέπει να φύγει σε λίγο ο ε, Υπουργό, θα του δώσουμε 10 λεπτά για να απαντήσει στις ερωτήσεις. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και όλους σας για τα ερωτήματα και τα σχόλια. Καταρχάς, από τα σχόλια σας κρατάω το εξής, ότι η πολιτική συνοχής είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κάτι ακόμη. Ότι αυτό δημιουργεί πραγματικά πολλές ανησυχίες και ερωτήματα. Και αυτό είναι και καλό και κακό. Θέλουμε όλα αυτά τα ζητήματα να τα ενσωματώσουμε στον τρόπο σκέψης μας για όλες αυτές τις διαδικασίες στις οποίες θα πρέπει να βασίζεται η μέλουσα πολιτική συνοχής. Και νομίζω ότι θα προσπαθήσω να ομαδοποιήσω κάπως τις ερωτήσεις. Υπήρξαν ερωτήσεις που δεν ήταν απολύτως σαφές ε, για μένα. Δεν κατάλαβα ακριβώς δηλαδή τι με ρωτήσατε. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπε η κυρία Σμέλκοβα για το δημοσιονομικό πλαίσιο και τις ε, οικονομικές συνθήκες. Ειδικότερα δεδομένων των συνθήκων που υφίσταται αυτή τη στιγμή. Θα είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για το μέλλον της ε, πολιτικής συνοχής. Η Ουγγρική Προεδρία εξ αρχής υποστήριξε την προσέγγιση βάσει της οποίας η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής θα έπρεπε να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική προτεραιότητα για την Ουγγρική Προεδρία. εκτός από την οικονομική συνοχή και η εδαφική συνοχή είναι μια ε, τρίτη διάσταση της, ε, της πολιτικής ε, συνοχής που συμπληρώνει τα άλλα δύο στοιχεία. Θα πρέπει λοιπόν η χρηματοδότηση να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο. Αυτή είναι μια κατηγορηματική θέση της Ουγγρικής Προεδρίας. Από τις συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων και υπουργών έβγαλε το συμπέρασμα ότι αυτή είναι άποψη της πλειονότητας των κρατών μελών όμως. Υπάρχουν βέβαια και αποκλίνουσες απόψεις. Για παράδειγμα, αναφερθήκατε για παράδειγμα στο σε ποιο βαθμό θα έπρεπε να δώσουμε προτεραιότητα στις περιοχές που έχουν καθυστερήσει και πρέπει να προλάβουν τις υπόλοιπες. Από τη στιγμή που θέλουμε μια ενσωματωμένη προσέγγιση και από τη στιγμή που θέλουμε να συνδυάσουμε τις ε, διάφορες πτυχές της ανάπτυξης που σε διαφορετική περίπτωση θα είναι κατακαιρματισμένες σε διάφορους ε, τομείς πολιτικής. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο πολιτικής, ε, χωρίς το οποίο η στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση 2020 δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί. Συνεπώς, οι πόροι πρέπει να οργανωθούν αναλόγως. Και υπάρχει και ένα ερώτημα σε σχέση με τη χρήση της χρηματοδότησης, κατά πόσο είναι στοχευμένη η χρήση ή αν ε, είμαστε προσανατολισμένοι στο αποτέλεσμα στους δείκτες. Είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητήσαμε τον Ιανουάριο, το συζητήσαμε Και τότε και σας είχα πει ότι η Ουγγρική Προεδρία υποστηρίζει την ε, ενίσχυση των δικτών και θα ήθελα να επανεπισημάνω τη θέση μας αυτή. Όπως είπα άλλωστε και στα εισαγωγικά μου σχόλια, ότι θα θέλαμε να υπάρχουν οι δείκτες και να υπάρχουν και συγκεκριμένοι όροι βάση... που θα μπορούσαν να είναι αποδεκτές, ε, αποδεκτή βέβαια από όλα τα κράτη-μέλη. Η πολιτική συνοχής δεν είναι μία ε, μια πολιτική ε, την οποία απλώς, ε, στην, στην οποία εμείς απλώς υποχρεώνουμε τα κράτη-μέλη. Πρέπει να γίνει ένας διάλογος. Η ιδέα αυτή είτε ε, το εδαφικό στοιχείο είτε το στοιχείο της, των πιο καθυστερημένων περιοχών είναι ένα ζήτημα που έχει άμεση σχέση και με το θέμα της ανταγωνιστικότητας. Νομίζω ότι αυτό το δίλημα πρέπει να επιληθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε πολιτικό επίπεδο και νομίζω ότι θα έπρεπε όλες οι πτυχές να ειδωθούν και από αυτή τη σκοπιά. Αυτή ήταν η θέση μας ήδη από τον Ιανουάριο. Κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε από τις συνεδριάσεις που είχαμε κατά τις τελευταίες εβδομάδες. Πρέπει να είμαστε συνεπείς και πρέπει να τονίσουμε αυτό το στοιχείο των πιο ε, καθυστερημένων περιοχών και να δούμε που μπορούμε να σκίσουμε να έχουμε και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από απόψε ως εδαφική συνοχής. Η αλήθεια είναι, επανέρχομαι στο θέμα των δικτών τώρα, Κατά τις τελευταίες εβδομάδες μετά από συνεδριά σε επίπεδο και πολιτικό αλλά και εμπειρογνωμόνων, δεν έχω ακούσει μια περιεκτική πρόταση. Υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν συστάσεις, αλλά δεν υπάρχει καμία συστηματική ε, πρόταση. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν μια τέτοια έννοια να συμπεριληφθεί στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αυτή τη στιγμή ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι βέβαιος ότι κάπου θα αναπτυχθεί η έννοια αυτή. Αλλά αν ψηφίζαμε σήμερα, οι παρόντες θα ψήφιζαν υπέρ μιας τέτοιας προσέγγισης. Πρέπει όμως η ιδέα αυτή να εκφραστεί με ένα λειτουργικό τρόπο για να μπορέσει να λειτουργήσει πράγματι στην πράξη. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να συζητηθούν και οι νέες δημοσιονομικές προοπτικές. Όταν λοιπόν θα γίνει η συζήτηση αυτή, θα έπρεπε τα κριτήρια να τα έχουμε ήδη στη διάθεσή μας, γιατί τότε η πολιτική συνοχή θα έχει μια πραγματική ευκαιρία να λάβει χρηματοδότηση σε κατάλληλο επίπεδο. Σε σχέση τώρα με τα σχόλια του Μάρκους, δεν κατάλαβα πολύ καλά την ερώτηση την πολύ συγκεκριμένη που έθεσε. Ίσως εγώ δεν κατάλαβα καλά, συγγνώμη. Αν έχετε την καλοσύνη να την επαναλάβετε μόνο για να προσπαθήσω να την καταλάβω καλύτερα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η μία ερώτηση. Ίσως ε, γι' αυτό δεν με καταλάβατε, λέει ο η Μια ερώτηση λοιπόν είχε να κάνει με την υπαγωγή σε όρους, conditionality, δηλαδή το γεγονός ότι η Ευρώπη ορίζει για τα κράτη-μέλη όρους, προϋποθέσεις με βάση τους οποίους, τις οποίες και μόνο θα προχωρήσει στην ε, λήψη αποφάσεων, είτε πρόκειται για τον ε, ανταγωνισμό, είτε πρόκειται για τις ε, προμήθειες, γιατί εκεί πέρα έχουμε την πτέρνα και εντοπίζονται οι καταχρήσεις, τα προβλήματα. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται να υπάρξει κάποια εξέλιξη με αυτόν ή αρκεί. Και η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με την ενδιάμεση εκείνη κατηγορία των περιφερειών εκείνων που έχουν ξεπεράσει το 75% επί του ΑΕΠ και μπορεί να έχουν μια συμπληρωματική στήριξη, αλλά όχι μόνο αυτές οι περιοχές, γιατί εκεί υπάρχει διαφορά τώρα. Όχι μόνο αυτές, όλες οι περιφέρειες οι οποίες πια αναγνωρίζεται ότι ανήκουν στο 75 έως 90%. Όχι μόνο αυτές που παλιά ήταν κάτω από το 75. Ε, αυτές δηλαδή οι οποίες ήδη πια είναι ευημερούσες περιφέρειες. Δεν είχαν προβλήματα ποτέ. ποτέ. Ε, ανέφερα ένα παράδειγμα νωρίτερα αλλά εν και άλλες, και άλλες περιφέρειες που δεν θα ήταν αιτιολογημένο ίσω. Ποια είναι η γνώμη σα για αυτή τη νέα ε, κατηγορία που θα σήμαινε υπαγωγή 22 περιφερειών τη Ευρώπη σε αυτήν. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κατάλαβα τώρα. Συγγνώμη που σας έκανα να, να επαναλάβετε την ερώτηση. Για το πρώτο σας ερώτημα, η απάντησή μου είναι ναι. η υπαγωγή σε όρους θα πρέπει να ενισχυθεί και εμείς θα την υποστηρίξουμε. Βέβαια, θα υπάρχουν και συγκεκριμένοι όροι. Δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο χωρίς την συμμετοχή των κρατών μελών. Οι κανόνες θα είναι σαφείς και θα είναι σαφές το πλαίσιο. Και εγώ λοιπόν υποστηρίζω την ιδέα αυτή, γιατί είναι απαραίτητη προκειμένου η πολιτική συνοχή να καταστεί αποδοτική και αξιόπιστη. Για το δεύτερο ερώτημα που θέσατε, τα τελευταία δυόμιση με τρία χρόνια διερχόμεθα κρίση, κάτι που δείχνει ότι ούτε στην Ευρώπη, αλλά ούτε και πουθενά αλλού, υπάρχουν ε, περιφέρειες ε, που δεν χρειάζονται ε, την υποστήριξη του είδους αυτού που μπορεί να παρέχει η πολιτική συνοχή. Δηλαδή, για παράδειγμα, το πρόβλημα της περιοχής του Παρισιού. Νομίζω ότι είναι ένα παρόμοιο πρόβλημα και γι' αυτό συμφωνώ εγώ με τη δική σας προσέγγιση. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Εκ μέρου όλων θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να σας πω ότι εκτιμώ όλος ιδιαίτερο συνεργασία με την Ουγγρική Προεδρία και ειδικότερα τη διαθεσιμότητά σας για τη συμμετοχή ε, των ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλες τις συνεδριάσεις που είχε προβλέψει η ε, Ουγγρική Προεδρία. Για μας είναι πραγματικά άνευ προηγουμένου, τουλάχιστον ε, η δική μου εμπειρία είναι αυτή. Τέτοιου είδου συμμετοχή δηλαδή σε ζητήματα πολιτική συνοχή πραγματικά δείχνει πόσο πολλή δουλειά έγινε στο πλαίσιο τη διακυβερνητική ε, συνεργασία ε, για να υπάρξει ένα τέτοιο πλαίσιο συμπερασμάτων. Θα σα ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ και ελπίζουμε κατά το τέλος της Προεδρίας σας να σας ξαναδούμε. Ευχαριστώ πολύ και θα ξανάρθω. Και εμείς ευχαριστούμε και είστε πάντοτε ευπρόσδεκτος. Μια και ο Μάρκος είναι εδώ, μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, ε, που είναι η δεύτερη ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση του Μάρκου Πίπερ για την μελλοντική πολιτική συνοχή είναι εδώ και ο Μισελ Ντελεμπάρ που εκπροσωπεί την Επιτροπή Περιφερειών, όπως επίσης ε, και έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής και Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής, τον κύριο Τσεντρώνε. Και θα ήθελα να δώσω καταρχάς το λόγο στον Μάρκους για τις παρατηρήσεις του. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκριση στο εγγραφείο εργασία μου. 36 ερωτήσεις είχα θέσει και όντως οι συνάδελφοι έκαναν τον κόπο, μάλιστα κάποιοι να απαντήσουν και στις 36. Πολλές λοιπόν ενδιαφέρουσες ιδέες είδα, τις οποίες προσπαθώ να ε, λάβω υπόψη στην έκθεσή μου, στο βαθμό του δυνατού. Η έκθεση ακολουθεί μια βασική φιλοσοφία, θα το πω έτσι, ότι δηλαδή η πολιτική συνοχή, η πολιτική διαρθρωτική, διαρθρωτικού ταμείου, δεν είναι αυτός δεν την θεωρούμε αυτοσκοπό ή αυτοδύναμη ιδέα, αλλά ένα εργαλείο για να ε, εφαρμοστούν σωστά άλλες σημαντικές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά κύριο λόγο δηλαδή η στοχοθέτηση του 2020 στον τομέα της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της δημογραφίας, της έρευνας, της καινοτομίας και άλλων αντίστοιχων επιλογών. Πιστεύουμε λοιπόν, τουλάχιστον εγώ στην έκθεσή μου, ότι θα πρέπει να διαφυλαχθεί το επίπεδο των, ε, της πρικοδότησης, τα κονδύλια δηλαδή στήριξης, όπως αναφέρονται, όπως έχουν οριστεί ήδη και πιστεύω επίσης ότι πέραν αυτής της βασικής τοποθέτησης ότι δηλαδή τα ερωτικά ταμεία αποτελούν ε, εργαλείο για το 2020 ότι μπορούν να αποτελήσουν, ότι αποτελούν και το νοτιαίο μυελό τη φιλοσοφία δηλαδή της πολιτικής συνοχής. Κατανομή και ευθύνη, κατανομή κονδυλίων και ευθύνη. Αυτό σημαίνει ότι μαζί με τα κρατημέλη, μαζί με τις περιφέρειες, θέλουμε από κοινού να εφαρμόσουμε τα ε, προγράμματα αυτά και όχι κατά κεντρικά οργανωμένη ε, και τομεακή ε, παρέμβαση, δηλαδή περιβάλλον, ενέργεια κτλ. Θέλουμε να είναι η κατανομή σε επίπεδο κρατών μελών. Βλέπουμε μέχρι στιγμής ότι είναι επιτυχής η περιφερειακή μας πολιτική. Υπάρχουν ακόμη ε, αποκλήσεις ανισότητες αλλά τις έχουμε περιορίσει σημαντικά. Έχουμε στόχο ανταγωνιστικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον οποίο έχουμε συμβάλει τα μάλα. Έχουμε πρόοδο και στην ε, κοινωνική ενσωμάτωση και στην οικολογία που έχουν βοηθήσει οι ίδιες περιφέρειες να εξασφαλιστούν. Όμως εξασφαλίστηκε γιατί, διότι εμείς σε μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης επιλέξαμε να έχουμε μία οριζόντια δυνατότητα στήριξης ε, για αυτή την περίοδο, δηλαδή όχι μόνο μία ε, παράθεση θα έλεγα περιφερειών όπου η μία ήταν ε, περιφέρεια στήριξης και άλλη μη, δικαιούχος η μη, αλλά και μια οριζόντια στήριξη από κοινού να προωθήσουμε κάποιες, κάποιους τομείς. Και έτσι έχουμε Κλάστρο, όπως λέμε, δηλαδή θύλακες ε, αναζωογόνησης σε περιφέρειες που φερειπήρ υπήρχαν μικρομέσες επιχειρήσεις που δεν τα πήγαν πολύ καλά. Ξεσφαλίσαμε συνεργασία με πανεπιστήμια που τα πηγαίνανε, είχαν καλή έρευνα, τεχνολογία και έτσι μπορέσαμε να προωθήσουμε διαπεριφερειακά αυτή την πρόοδο. Είναι μια προσέγγιση αυτή την οποία, ε, η οποία φαίνεται ότι έχει αποδειχθεί στην, κατά την άποψή μα επιτυχημένη. Φαίνεται όμω ότι η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα πάει να καταστρέψει ακριβώ αυτή την προσέγγιση. Δηλαδή, μόνο μία προσέγγιση μέσα στην ίδια περιφέρεια θα επιτρέπεται συνεργασία ενό πανεπιστημίου με μια μικρομεσαία επιχείρηση, όχι διαπεριφερειακά. Δεν θα επιτρέπεται δηλαδή η σύνδεση του δυναμικού διαφορετικών περιφερειών. Άρα, αυτό που έχω να πω είναι έπαινο για τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα, έπαινο για την φιλοσοφία που την επιλογή, τη φιλοσοφική, την ιδεολογική που οδήγησε στα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα, αλλά και τώρα περνάω στις επικρίσεις μου, βλέπουμε ότι η προσθέμενη αξία και η αποτελεσματικότητα αυτής της πολιτικής πρέπει να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο. Για μένα η καλύτερη περιφερειακή πολιτική είναι η εσωτερική αγορά. Εφόσον λειτουργεί η εσωτερική αγορά, εφόσον ε, εντα πραγματικοποιούνται οι επαφέ μεταξύ των επιχειρήσεων, φερειπίν εξαγωγέ, ε, ε, ενισχύονται και η δημιουργία θέσεων εργασία μέσα στι ίδιε περιφέρειε. Αλλά η εσωτερική αγορά μπορεί να λειτουργήσει μόνο εάν λειτουργεί αποτελεσματικά και η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όπου εντοπίζεται το έλλειμμα και ω προ την χορήγηση των κονδυλίων ενίσχυση και ω προ την ανάθεση των ε, έργων και ως προς ε, τις θυμές και γι' αυτό υποστηρίζω ιδιαίτερο την προσέγγιση Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπαγάγει περισσότερο τα κονδύλια στο μέλλον ε, σε όρους, το ζήτημα δηλαδή που συστήσαμε μόλις τώρα, και να εξετάζει εάν λειτουργούν αποτελεσματικά οι δημόσιες προμήθειες στα κράτη-μέλη, εάν υπάρχει και αν αυτό δεν συμβαίνει, αν δηλαδή δεν λειτουργούν αυτά τα έργα κατά τρόπο αντικειμενικό και ούτερο, να μην χορηγούνται οι ε, ενισχύσεις από τα κοινοτικά κονδύλια. Άρα πρέπει να έχουμε και σαφείς δείκτες με βάση του οποίου θα καταμετρούμε την πρόοδο από την οποία θα εξαρτάται η διάθεση των κονδυλίων, η ακροή των κονδυλίων, αλλά πιστεύω ότι αυτόχρονα θα πρέπει και να επικεντρωθούμε στα σημεία εκείνα στα οποία έχει κατά κύριο λόγο ε, αρμοδιότητες Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τομεί ευθύνη Ευρωπαϊκή Ένωση, έρευνα, διαπεριφερειακή περιβαλλοντική προστασία, οικολογική προστασία, ε, μεταφορέ, ναι, αλλά όταν βλέπω ότι υπάρχουν δείκτες, όπως τώρα από τους πρώτους καταλόγους που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, δείκτες λοιπόν οι οποίοι έχουν να κάνουν με την διάθεση κονδυλίων με βάση τον αριθμό των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς ή τον αριθμό των παιδιών που εγκαταλείπουν προώρα το σχολείο τους, Αυτά ως δείκτες για μένα σημαίνουν κίνδυνο να εξευρωπαϊστεί η κοινωνική πολιτική, η πολιτική της εκπαίδευσης, της παιδείας και αυτό σημαίνει τι, ότι με τα λίγα χρήματα που έχουμε στην πολιτική συνοχή δεν θα μπορούσαμε ποτέ να κάνουμε ουσιαστικό έργο. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα, εκεί όπου κατά κύριο λόγο υπάρχει αρμοδιότητα εθνική ή και περιφερειακή, σχολείο Φερρυπίν, να μεριμνούμε έτσι ώστε να έχουμε πρότυπα ως έργα, μοντέλα δηλαδή, τα οποία θα μπορούν να μεταφερθούν ενδεχομένως σε κάποιες άλλες περιφέρειες και να εφαρμοστούν, αλλά όχι δείκτες όπως παιδιά έχει κάθε παιδικό σταθμό ή συνολικά όλη η παιδική σταθμή μιας χώρας, μιας περιφέρειας. Γιατί εκεί νομίζω ότι χάνουμε το μέτρο και μπαίνουμε στα χορύφια των κρατών μελών. Και θα πρέπει να τηρηθεί με ε, θρησκευτική ευλάβεια η αρχή της επικουρικότητας στον τομέα αυτών. Κάτι ακόμη που πιστεύω θα, ήθελ, θα έπρεπε να μπει στην ε, πολιτική συνοχή η ε, έμφαση βεβαίως στις πιο αδύναμες περιφέρειες, στις άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες είναι πολύ σημαντική. Όμως πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει και ο οριζόντιος στόχος της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας να διαφυλαχθεί και να ενισχυθεί. Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε κοινέ ε, προτεραιότητες ε, ή πρωτοβουλίες όπως δημογραφικού τύπου ή μάλλον με δημογραφικά κριτήρια αλλά όχι μόνο μια κατηγορία η οποία να σημαίνει τελικά ότι μια περιφέρεια μπορεί να μπει σε μια νέα κατηγορία και να μην ξαναβγεί ποτέ από εκεί. Γιατί ακούγεται ότι μπορεί να υπάρξει ένα τέτοιο μοντέλο, δηλαδή μια νέα κατηγορία ε, ενίσχυσης, περιφερειών ενίσχυσης. Ε, αυτό όμω, αγαπητοί συνάδελφοι, θα είναι μεγάλο σφάλμα. Δεν θα βγουν ποτέ από αυτήν την κατηγορία οι εν λόγω περιφέρειε. Θα πρέπει να δούμε αυτέ οι περιφέρειε γιατί δεν είναι πια οι πιο φτωχέ περιοχέ τη Ευρώπη, γιατί όταν είναι οι Έλληνε, οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι σε μια καλύτερη κατάσταση από τι φτωχότερε περιοχέ τη Ευρώπη, θα πρέπει να του εντάξουμε σε μια άλλη περιφέρεια στήριξη, σε μια άλλη κατηγορία μάλλον περιφερειών στήριξη. Δεν θα έπρεπε να τους αφήσουμε να προχωρήσουν μόνοι τους. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα σήμαινε και το τέλος ή την αρχή του τέλους αξιοπιστίας της, περιοχή, της ε, πολιτικής μας συνοχής. Θα πρέπει να στηρίξουμε τους πιο ασθενείς, τους πιο αδύναμους. Αυτό σημαίνει η Ευρώπη. Ο ενδιάμεσος στόχος, η ενδιάμεση κατηγορία στόχου για μένα δεν έχει καμία θέση σε μια πολιτική συνοχή. Και επίσης θα ήθελα ως προς το περιεχόμενο της έκθεσης να πω ακόμη δύο λόγια για το ε, θέμα των υποδομών, σε ποιο βαθμό θα επιστερχόμαστε πλέον σε υποδομές. Νομίζω ότι θα πρέπει να ε, και πρέπει να ε, υποστηρίξουμε υποδομές στην ενέργεια εκεί όπου η αγορά δεν αρκεί να τη στηρίξουμε με ευρωπαϊκά κονδύλια και ιδιαίτερα στις παραμεθόριες περιοχές να μπορέσουμε να βοηθήσουμε για δικτύωση διασυνοριακή ή υπερσυνοριακή ε, γιατί είδαμε και στην έκθεση αλλά και στη δική μου στο στόχο 3 την ε, ενίσχυση κατά 7%, μάλλον αύξηση στο 7% από το 2,5%, νομίζω ότι αυτό θα αποτελούσε ένα πραγματικό, μια πραγματική απόδειξη της προσθέμενης αξίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, αγαπητοί φίλοι. Αν μπορούσαμε δηλαδή στι παραμεθόρειες περιοχές να πείσουμε τον πολίτη ότι μπορεί να στηρίζεται στην βελτίωση των διασυνοριακών δικτύων, να την δει απτά, στην καθημερινή του ζωή, νομίζω ότι ε, θα ήταν σημαντική επιτυχία και αυτό μπορούμε να το κάνουμε σε απόλυτη ανόηση με τι περιφέρειε. Είναι κάτι το ορατό, είναι κάτι το οποίο στη τελευταία ανάλυση μπορούν να προσφέρουν στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε οι περιφέρειε. Και εν προκειμένου ε, πιστεύω ότι η διαγώνια χρηματοδότηση του προγράμματος ε, πλαισίου για την έρευνα και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι νομίζω πολύ σημαντική. Δηλαδή αν έχουμε να υποστηρίξουμε σε ένα ε, εργοστάσιο την απασχόληση ατόμων με αναπηρίες φερρυπίν στο πλαίσιο του Κοινωνικού Ταμείου, ταυτόχρονα θα μπορούσαμε να ε, περιμένουμε οι δομές οι οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί από δικά μας κονδύλια και να αποκτήσουν μία διάρκεια, να μην εξαφανιστούν δηλαδή μόλις τελειώσει η χρηματοδότηση. Αυτές νομίζω ότι θα πρέπει να είναι οι επιλογές μας. Ε, στηρίζω όπως εξήγησα νωρίτερα τις ε, επιλογές της Επιτροπής. Προσπάθησα για συγκεκριμένα σχέδια να προτείνω ε, κάποιες ιδέες για σχέδια. Παρακαλώ κοιτάξτε αν θέλετε στα σημεία 1 και 2 των προτάσεών μου. Και ε, όπως είπα, γνώμονος θα πρέπει να είναι εάν έχουμε ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία ή όχι με βάση αυτά που χρηματοδοτούμε. Ε, για, τα, για τα οικονομικά τώρα. Θα έλεγα ότι θα ήταν καλό να σπρώξουμε τις περιφέρειες σε ανάληψη περισσότερων ευθυνών, δηλαδή να περιορίσουμε την ικανότητά τους να απορροφούν κονδύλια από δωρεές αλλά να τους βοηθήσουμε, να τις βοηθήσουμε να βρούνε κονδύλια από άλλου τύπου χρηματοδότηση, δάνεια κτλ. Το 90% της χρηματοδότησης επί του κόστους ενός έργου ε, θα πρέπει να αφορά ε, όχι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα αλλά το προϊόν της, το, της απόφασης για τη συγχρηματοδότηση κατά την άποψή μου. Επίσης θα πρέπει να κοιτάξουμε περισσότερο το θέμα της πιστοποίησης των ελεγκτικών αρχών, μία ελεγκτική αρχή ανακράτος κατά την άποψή μου, η οποία όμως θα πρέπει να περάσει από μια διαδικασία πιστοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο Πλήρω 100% και μόνο όταν έχει μπει η τελική σφραγίδα της πιστοποίηση, θα μπορεί αυτή η αρχή να αναλάβει το έργο και να αναγνωριστεί ω ελέγχου αρχή. Εάν κάποιο κράτος όμως αρνείται, τότε θα πρέπει να πιέσουμε για περισσότερη πίεση ελεγκτική προς το κράτος αυτό ή προς τα κράτη αυτά. Δηλαδή πιστεύω ότι θα πρέπει εκείνος ο οποίος βλέπουμε ότι συνεργάζεται καλά να έχει μια ελάφρυνση από την πίεση την ελεγκτική, αλλά εκείνο ο οποίο δεν κάνει σωστά τη δουλειά του να πιέζεται περισσότερο και να ελέγχουμε πιο αυστηρά το πού χρησιμοποιούνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Για την ε, πολιτική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε, και θα ήθελα να το υπογραμμίσω εδώ, ε, απέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ε, ε, σαφέστερη, εντονότερη εμπλοκή της Επιτροπής Περιφερειακών ε, Θεμάτων στην ε, πολιτική της γειτονίας και όπως λέει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε κράτη να εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση απροετοίμαστα και αναφέρομαι, έχω υπόψη μάλλον εδώ τα παραδείγματα της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας όπου θα έπρεπε πιστεύω να είχαμε φροντίσει νωρίτερα τα προενταξιακά μέσα να χρησιμοποιηθούν περισσότερο και στη διαφορετική πολιτική πράγματα τα οποία όμως τις ξέφυγαν της περιφερειακής μας επιτροπής όλος διόλου καθόλου. Έχοντας λοιπόν δει τι ε, έχουμε μπροστά μας ως ε, διεύρυνση, δηλαδή Κροατία και Τουρκία, θα πρέπει να αποφύγουμε την διάπραξη του ίδιου σφάλματος, θα πρέπει να φροντίσουμε την ε, υποψηφιότητα της Τουρκίας να την οξολογήσουμε και, και με βάση τις τη διαρθρωτική μας πολιτική και τη δυνατότητα απορρόφησης διαρθρωτικά της χώρας αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναλόγως να την κρίνουμε. Και όπως είπα πάντα με επίκαιρα στοιχεία. Αυτά όσον αφορά την πρότασή μου. Ευχαριστώ θερμά όλους τους συναδέλφους οι οποίοι συνεργάστηκαν στην προσπάθεια αυτή. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποια σημεία που χρειάζονται ακόμη συζήτηση, ίσως και εντατική συζήτηση. Πιστεύω όμως ότι αυτή η νέα κατεύθυνση, ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής, και θα προέρχεται αλλά και θα πρέπει να παραμείνει στις περιφέρειες. Χαίρομαι λοιπόν για τη συζήτηση και ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ Μάρκους Πίπερ για αυτήν την εμπνευστική ε, ε, ε, παρουσίασή σου. Κάθε φορά που μας παρουσιάζεις μία έκθεση υπάρχει και κάτι διαφορετικό. Επειδή δεν θέλω πάλι τους τελευταίους να τους πιέσω, θα ήθελα να πω ότι πρέπει να είμαστε σύντομοι. Είναι πολλοί αυτοί που θέλουν να λάβουν το λόγο και δεν θα τα καταφέρουμε αν δεν είναι όλοι σύντομοι. Βέβαια δεν θα περιορίσω τον Μισελ Ντελμπάρ και τον Καμέλο Τσεντρόνε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Μισελ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη γενεοδορία σας, ε, κυρία Πρόεδρε. Πριν από 10 μέρες ε, η Επιτροπή Περιφερειών παρουσίασε, ε, κυρίες και κύριοι, ε, ενέκρινε ε, με πολύ μεγάλη πλειοψηφία την έκθεση την οποία παρουσίασα εγώ. Μόνο τρεις ψήφοι κατά και διάβασα την έκθεση του κυρίου Πίπερ. Αν, αν μου επιτρέψετε θα επανέλθω σε πολύ συγκεκριμένα ε, σημεία θα προσπαθήσω να τηρήσω τα χρονικά μου περιθώρια. Υπάρχει ένα, ένας βαθμός σύγκλησης αρκετά μεγάλος και υπάρχουν επίσης και κάποιες ε, αποκλήσεις. Πρώτη από αυτέ, είναι ότι και εμεί η Επιτροπή Περιφερειών θέλουμε να είναι προσβάσιμη για όλε τι περιφέρειες Ευρωπαϊκή Ένωση ε, που θέλουν να συμμετέχουν ε, σε οικονομική ανάπτυξη, στην οικονομική ανάπτυξη ο, η πολιτική που έχει τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα είναι, αυτές που είναι αυτή που είναι η πιο ορατή από όλες τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ήθελα πραγματικά να εκφράσω την, ευχα... ικανοποίησή μου ε, για την συνεργασία σε πολλά επίπεδα, για την εδαφική συνοχή και θα θέλαμε να πούμε ότι σε σχέση με το 7% που ανέφερε ο εισηγητής, ε, σε αυτό συμφωνώ απολύτως. Όσον αφορά την ανάλυση του κοινωνικού ε, ε, ταμείου, επίσης συμφωνούμε για τη συμμετοχή του περιφερειακού επίπεδου, όμως διαφωνούμε με τις μονοθεματικές προσεγγίσεις, διότι υπάρχουν και οι άκρος απόκεντρες περιφέρειες. Τώρα, η πολιτική συνοχή και η σχέση τους με την ε, διαρθρωτική μεταρρύθμιση για να υπάρχει επιλεξιμότητα μακροοικονομική χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα με τα διαρθρωτικά ε, ταμεία που την καλύπτουν, ενώ οι εθνικές κυβερνήσεις δεν σέβονται το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, αυτό κατά τη γνώμη μου θα ήταν ε, πραγματικά μία κύρωση ε, άνευ στο περιφερειακό επίπεδο. Ε, δεν άκουσα μια συγκεκριμένη θέση όσον αφορά ε, τις επιδόσεις, κύριε Σιγητά. Εμείς διαφωνούμε ε, σε περίπτωση που ενός τέτοιου είδους ε, αποθεματικό ε, χρησιμοποιηθεί για περιοχές πλούσιες που έχουν ήδη πάρα πολλούς πόρους. Είμαστε υπέρ λοιπόν με μιας ευελιξίας η οποία θα μπορούσε να ισχύει σε κάποιες περιπτώσεις. Έχουμε λοιπόν και κάποιες διαφωνίες. Το πρώτο θέμα είναι το θέμα της εναρμόνης πολιτικής συνοχής με τη στρατηγική για το 2020. Πιστεύουμε στην Επιτροπή Περιφερειών ότι η πολιτική συνοχής δεν μπορεί να υποβαθμιστεί σε μία, ένα απλό εργαλείο της στρατηγικής 2020 μπορεί να συνεισφέρει, αλλά πρέπει να μπορεί να επιτύχει και άλλους στόχους και συγκεκριμένα την μείωση των κοινωνικών, εδαφικών και οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των, περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν αφορά μόνο τη στρατηγική του 2020. Ε, επίσης διαφωνούμε για ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό για μας, των ενδιάμεσων περιφερειών. Ε, σε μεγάλη πλειοψηφία η Επιτροπή Περιφερειών υπάρχουν περιοχές ανάμεσα στο 75% και 85% του κοινοτικού ΑΕΠ. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να τις μεταχειριζόμαστε με τον ίδιο τρόπο ε, με τις ε, ε, περιφέρειες που υπερβαίνουν τα ποσοστά αυτά. Είναι λοιπόν νομίζω λάθος χρήση αυτής της, αυτής της ιδέας των ενδιάμεσων περιφερειών. Θα θέλαμε όσον αφορά το ΑΕΠ να υπάρξει μια ευρύτερη προσέγγιση. Δεν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο το ΑΕΠ ω κριτήριο. Πρέπει και άλλες πτυχέ να λάβουμε υπόψη. Θα θέλαμε για παράδειγμα ε, να εμβαθύνουμε ακόμη περισσότερε εργασίε εργασίες και μεθοπρόθεσμη αναθεώρηση της περίοδου προγραμματισμού να λάβει υπόψη και άλλα κριτήρια ε, και όχι μόνο το ΑΕΠ. Το θέμα τώρα της εκπνοής επόμενη προγραμματικής περίοδου για μας ε, επίσης δημιούργησε κάποια προβλήματα. Ε, είμαστε μάλλον υπέρ του 5 συν 5, γιατί αυτό θα έδινε τη δυνατότητα μια, ε, μιας χρήσιμης αναθεώρησης. Αυτά κυρία Πρόεδρε, έκανα τις περισσότερες από τις παρατηρήσεις μου στο λιγότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω από τον Καρμέλο Τσεντρώνε να παρουσιάσει τα σχόλιά του. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή Πίπερ, τον οποίο συνάντησα ήδη και απάντησα σε 20 από τις ερωτήσεις του που μου είχε υποβάλει και βρήκα και αρκετά πράγματα στην έκθεσή του. Συμμερίζομαι σε μεγάλο μέρος τα όσα υποστηρίζει και σε όσα υπόθηκαν σήμερα το πρωί. Δεν θα επανέλθω σε αυτά. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στην προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή να προσθέσει αυτή την αξία σε αυτά και να προσπαθήσει ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παίξει ακόμα περισσότερο ε, δυνατό ρόλο στα σχέδια αυτά και ειδικότερα στο να είναι κάτι το υποχρεωτικό η εκτίμηση των τελικών αποτελεσμάτων και είναι σημαντικό, θεμελιώδες αυτό θα έπρεπε να επιμείνουμε ας πούμε στο θέμα του συντονισμού των κονδυλίων και αυτό τα λέτε προς, προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά τέλος πάντων ε, είναι σημαντικό το θέμα για μια ενιαία αρχή για να πετύχει κανείς το στόχο που έχει θέσει όπως εσείς και ακόμα κάτι για την απλούστευση. Αυτή η απλούστευση νομίζω ότι αποτελεί το πρώτο, το σημαντικότερο πρόβλημα όχι μόνο για λόγους χρόνου. Χρειάζεται και στην αρχική στιγμή να κάνουμε μια εκτίμηση όλων των διαδικασιών σε κάθε σχέδιο, να έχουμε τη σωστή πορεία, να το δούμε, να το εξετάσουμε και όσον αφορά την εκτίμηση από διοικητικής πλευράς, ε, βλέπουμε ότι ο καθένας επιβάλλει τη μέθοδό του. Αυτό που υπενθύμησε προηγουμένως ο συνάδελφος, αυτό του 2020, θα πρέπει και εκεί κάπως να ξεχωρίσουμε τα πράγματα. Πραξενεύω που δεν το κάνει εδώ, δεν το κάνουμε εδώ. Πέρα από αυτό, να δούμε τη στρατηγική χρηματοδότηση. Όλα αυτά δεν εξαρτώνται μόνο από την πολιτική συνοχή. Επίση, συμμερίζουμε τη θέση τη Επιτροπή Περιφερειών για τι ενδιάμεσε περιφέρειε, όπω επίση και την εκτίμηση του ΑΕΠ. Χρειάζονται επίσης και άλλες παράμετροι για να δούμε ποιες είναι οι συνθήκες που ισχύουν σε μια περιοχή και όχι μόνο το παραδοσιακό ΑΕΠ και εδώ δεν θα ήθελα να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Λοιπόν, μιλάτε για την εταιρική σχέση και πολύ σωστά. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι αυτό το συνδέεται μόνο ανάμεσα στην ιδιωτικό τομέα και στα δημόσιο περιφέρεια, επιτροπή, όλα αυτά μεταξύ τους. Αυτό είναι ένα αίτημα πώς μπορεί να γίνει στα πλαίσια της αυτονομίας του Κοινοβουλίου να μπορέσει να προβλέψει αυτή την κοινωνική, οικονομική, εταιρική σχέση εκείνων που συμμετέχουν και πριν και μετά στην αρχή και στο τέλος να δούμε όλη τη διαδικασία, όλη την πορεία σε κάθε επίπεδο και αυτό για να είναι ορατή όσο γίνεται καλύτερα και διάφανη αυτή η πολιτική θα μπορούσαμε να θετήσουμε αυτό που έκανε και η ΚΑΠ την Κοινωνική πολιτική, να δούμε όλες τις χρηματοδοτήσεις, ποιος ε, ε, παίρνει αυτά τα χρήματα κλπ. Έτσι να έχουμε όσο γίνεται περισσότερη διαφάνεια από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ λέει Πρόεδρος. Και τώρα το, ο σκιώδης εισογητής, ο κύριος Γιώργος Σταυρακάκης έχει το λόγο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή και την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει. Έχουμε στα χέρια μας ένα κείμενο που μας θυμίζει ποιος είναι ο πραγματικός στόχος της πολιτικής συνοχής και πού θα πρέπει να εστιάζει. Στηρίζω επιφύλακτα τις πιο πολλές από τις προτάσεις του εισηγητή. Είναι μια σειρά προτάσεων για λόγους οικονομίας χρόνου. Δεν θα τις αναφέρω ε, ξεχωριστά. Όμως, υπάρχουν κάποια σημεία του σχεδίου έκθεσης τα οποία δεν μπορώ να συμφωνήσω. Πρώτον, είναι η πρόταση για ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση στο, Ταμείο Κοινωνικό Ταμείο, στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Όπω όλοι γνωρίζουμε και τα δύο αυτά ταμεία έχουν εντελώ διαφορετικού στόχου και διαφορετικά κριτήρια παρέμβαση. Δεύτερον, ισχύει το ίδιο και για την πρόταση του εισηγητή για την συγχώνευση του Ταμείου Συνοχή με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Υπάρχουν επίσης κάποια άλλα σημεία για τα οποία θα ήθελα να ζητήσω από τον εισηγητή να μας δώσει κάποιες περαιτέρω διευκρινήσεις. Πρώτον, σχετικά με την πρόταση για σταδιακή μείωση της παροχής ενίσχυσης στις περιοχές που έλαβαν τη μέγιστη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του στόχου σύγκληση. Θα υποστηρίζετε κύριε Πίπερ ότι μια τέτοια σταδιακή μείωση θα πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένα και σαφώς καθορισμένα κριτήρια που έχουν να κάνουν με τις σημερινές ανάγκες και το επίπεδο ανάπτυξης αυτών των περιοχών. Και δεύτερον, μία ερώτηση σχετικά με την παράγραφο 51 και την καθιέρωση αυτόματα εφαρμόσιμων κανόνων για εντατικότερο έλεγχο σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος παραβιάζει σε σημαντικό βαθμό τα κριτήρια σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν η πρόταση του εισηγητή στοχεύει απλώς στη διενέργεια αυστηρότερων ελέγχων ως προς τη διαχείριση των πόρων σε τέτοιες περιπτώσεις, τότε είμαι θετικός. Αν ωστόσο η πρόταση αναφέρεται έμεσα και στην αυτόματη επιβολή κυρώσεων, τότε μιλάμε για σύνδεστο των στόχων της πολιτικής συνοχής με μακροοικονομικές προϋποθέσεις, κάτι τέτοιο το οποίο λυπάμαι δεν μπορώ να στηρίξω. Ευχαριστώ. Uh, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον Πίπερ, τον Μάρκους, για την εργασία του αυτή. Ε, είναι υπέροχο το στυλ, το ύφος με το οποίο συντάσσει ε, παρουσιάζει τα πράγματα με ιδιαίτερη σαφήνεια και αυτό είναι κάτι το πολύ θετικό. Επίσης χαίρομαι που δείχνει καθαρά τον σημαντικό ρόλο της πολιτικής συνοχής στα πλαίσια της στρατηγικής του 2020 και αυτό το προτείνει σαν ένα μέσο για να προωθηθεί η στρατηγική αυτή. Και επίσης είναι σημαντικό να έχουμε σημαντική επαρκή χρηματοδότηση. Συμφωνώ σε πολλά θέματα με τον εισηγητή από αυτά που αναφέρει, όπως την ίσχυση του στόχου 2. Νομίζω ότι είναι κάτι το πολύ θετικό όταν μιλάμε για αυτά τα κλάστερς καινοτομία και μπορούμε να αναφέρουμε επίσης και τη συνεργασία στα πλαίσια του προγράμματος πλαισίου, με ποιο τρόπο προωθείται αυτή και πολλά πράγματα, πολλούς στόχους που μας βρίσκουν σύμφωνους όσον αφορά τα ξεχωριστά κονδύλια και τα μία αυτό συμφωνώ με την θέση του εισηγητή, την τοποθέτησή του. Επίσης ιδιαίτερα με ικανοποιεί ότι το έγγραφο λαμβάνει υπόψη τις διάφορους στόχους, υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες που ισχύουν σε κάθε περιφέρεια και πρέπει αυτή την διαφορά να τη λαμβάνουμε υπόψη. Και επίσης για τις μακροπεριφέρειες θα νομίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους μηχανισμούς χρηματοδότησης που διαθέτουμε ήδη αντί να αρχίσουμε τώρα να ε, το υποστηρίζουμε αυτή μέσω του προπολογισμού να γίνει αυτή η χρηματοδότηση. Θα πρέπει να υποφεληθούμε όσο γίνεται περισσότερο από τους υπάρχοντες μηχανισμούς και για την ενδιάμεση κατηγορία περιφερειών σίγουρα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ένα μόνιμα στοιχείο εδώ βέβαια αυτό περιλαμβάνει και διάφορους κινδύνους για την προσεχή χρηματοδότηση. Εγώ προς την κατεύθυνση αυτή δεν συμφωνώ και τόσο με τον εισηγητή. Έχω μια τοποθέτηση δικιά μου κάπως πιο ουδέτερη γιατί νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερη συζήτηση, περισσότερο διάλογο για να δούμε ποιο είναι το καλύτερο στην περίπτωση αυτή. Και ακόμα για τα διάφορα ταμεία. Εντάξει, καλό θα είναι να επιφεληθούμε από αυτά που διαθέτουμε ήδη. Θα έπρεπε ο εισηγητής να μας πει κάτι περισσότερα πράγματα και πιο συγκεκριμένα. Τι γίνεται με τα ταμεία, μήπως θέλει κάποια βασική, ριζική μεταρρύθμιση και για το σφαιρικό αυτό χαρακτήρα. Σιγά σιγά εξ, ε, διάφορες χρηματοδοτήσεις εξαφανίζονται. Ίσως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο το κοινωνικό ταμείο γιατί τα κριτήρια και οι στόχοι ε, μέσα των οποίων όλα αυτά κατανέμονται δεν είναι και τόσο σαφή και συγκεκριμένα. Κάπως θολά είναι. Γι' αυτό ακριβώς μήπως θα μπορούσε να μου πει ο συγκητής την άποψή του. Επαναλαμβάνομαι ότι τα πράγματα θα πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια της περιφερειακής πολιτικής, της πολιτικής συνοχής. Θα πρέπει δεν να αποδίδουμε τους κατάλληλους, τις κατάλληλες προτεραιότητες και αυτό το υποστηρίζω. Και όσον αφορά την απλούστευση της περιφερειακής πολιτικής και της ε, ε, απάτες πώς θα μειωθούν. Ε, συμφωνώ, συμφωνώ ότι υπάρχουν ε, ορισμένες προϋποθέσεις και πρέπει να δούμε πώς συνδέονται οι προσπάθειες με τα αποτελέσματα. Χρειάζεται πάντως να συνεχίσουμε πάνω σε αυτό το δρόμο και ακόμα κάτι. Εάν έχουμε ένα αυτόματο σύστημα κυρώσεων, δεν ξέρω, αλλά εντάξει, καλό, θετικό κατά την απόψή μου θα πρέπει, καταλαβαίνω τι είναι κάτω από αυτά. Χρειάζεται όμως να το προσέξουμε ιδιαίτερα γιατί να το εξαρτήσουμε αυτό από τα υπόλοιπα. Ναι, ναι, τελειώσατε, εντάξει, καταλαβαίνω, με συγχωρείτε. Και πολύ γρήγορα τα λέγατε. Θα ήθελα επίσης να σας ζητήσω να μιλάτε λίγο πιο αργά, για να σας παρακολουθούν και οι διερμηνείς. Ο κύριος Σίμων. Αξιότιμη κύριε Σιχτά, ευχαριστώ πολύ για την ε, έκθεση. Έχω παρατηρήσει στο 33 καταρχάς, εκεί που γίνεται λόγος για τη συμμετοχή των ε, κρατών μελών και των ε, περιφερειών. Υπάρχει μια αντίστοιχη παρατήρηση δική μου σήμερα στην έκθεση Φλάσακ, δηλαδή θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο και να ζητήσουμε ρητά τη συμπερίληψη της περιφερειακής διάστασης και συγχρηματοδότηση θα πρέπει να γίνεται εφόσον πρόκειται να περάσει η συγχρηματοδότηση αυτή μέσω ενό τρίτου, θα πρέπει να το ρωτάμε εάν πράγματι θέλει το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε. Νομίζω ότι έτσι θα έχουμε καλύτερο ποσοστό απορρόφησης, δηλαδή με καλύτερη συμμετοχή της περιφερειακής, της, της ε, περιφερειακής διάστασης εάν συμμετέχει και αυτή στην ανάπτυξη κατάρτιση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Επίσης πιο πάνω στο σημείο 9 των τοποθετήσεων των θέσεών σας εκεί όπου γίνεται λόγος για τα επιχειρησιακά προγράμματα της ε, τα μεγάλα αστικά κέντρα, μετροπολιτικά κέντρα, μετροπολιτικές περιφέρειες μάλλον και την ευθύνη στην υλοποίηση των προγραμμάτων για τη Γερμανία, την κοινή μας πατρίδα. Θα πρέπει να πω όμως ότι οι μετροπολιτικές περιφέρειες είναι ακριβώς εκείνες οι οποίες δυνάμει της νομοθεσίας έχουν και την δημοκρατική νομιμοποίηση για την επεξεργασία αυτών των προγραμμάτων το Ανόβερο Φερρυπίν, Μητροπολιτική Περιφέρεια ή ε, Νέκαρ. Είναι ακριβώς περιπτώσεις όπου λειτουργικές ε, συνεργασίες επιτρέπουν ακριβώς την εξασφάλιση αυτής της νομιμοποίησης, δημοκρατικής νομιμοποίησης και την ανάπτυξη των προτάσεων από αυτές τις Μητροπολιτικές περιφέρειες που ε, αναπτύσσονται, θα, επεκτείνονται θα έλεγα σε περισσότερες από μία εθνικές περιφέρειες. Ρήνος Νέκαρ είναι τρεις περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωσης που μόνες τους δεν μπορούσαν να επιτρέψουν, να, να διεκδικήσουν μάλλον μια ε, ομοιόμορφη πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά μπορούν μαζί να διεκδικήσουν κοινά προγράμματα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να διευρύνουμε το, το φάσμα, τουλάχιστον να επιτρέψουμε τη διεύρυνση του φάσματος. Κύριε ευχαριστώ για την εργασία σας. Να επανέλθω σε δύο στοιχεία που θεωρώ εγώ τουλάχιστον σημαντικά αλλά και εντελώς αντιφατικά μεταξύ τους. Για να δούμε τη γράφω 19. Το ΑΕΠ θα πρέπει να παραμείνει το πρώτο και κύριο κριτήριο. Τι λέτε μετά τα εθνικά όργανα έχουν περιθώρια λιγμών και θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν και άλλους δείκτες. Αυτοί οι άλλοι δείκτες ποιοι είναι. Εδώ ε, βλέπουμε να εμφανίζεται μια αντίφαση. Εμείς ε, σε μετροπολογία θα προτείνουμε ποιοι θα είναι αυτοί οι ενδείκτες γιατί χρειάζεται ο τρόπος σκέψης μας να είναι διαφορετικός εκτός από με μόνο το στόχο την αύξηση του ΑΕΠ ε, σχετικά με την επίπεδο ποιοτικά των ε, πολιτών. Σχετικά λοιπόν με αυτές τις ενδιάμεσες περιφέρειες, ε, η Ευρωπαϊκή μέσω της εκθεσίας σας θα πρέπει να δείξει ότι είναι υπέρ της δημιουργίας της κατηγορίας αυτής της ενδιάμεσης ε, και θα πρέπει να δούμε και την πρωτοβουλία της Επιτροπής που υποστηρίζει και η έκθεση της Επιτρής Περιφερειών του κ. Ντελεμπάρ και θα πρέπει να το υποστηρίξουμε αυτό. Έτσι, ναι, πραγματικά και στο Συμβούλιο, ώστε τα κράτη-μέλη να τα πείσουμε όσα τουλάχιστον διστάζουν ακόμα ότι αυτό το phasing in και το phasing out, αυτό το μπέρδεμα που κάνουν τον μπαλώματα εδώ και εκεί δεν είναι θετικά μακροβάσμα. Θα πρέπει να δούμε και, το ε, μεταβαλλόμενο και τις μεταβολές που επιφέρονται. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτές σε ενδιάμεση κατηγορία και θα πρέπει να υπερασπιστούμε την ιδέα αυτή. Αυτή είναι η άποψή μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο Ελίωρο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για την δουλειά του. Νομίζω όμως ότι σε επίπεδο εργασιών μας είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε την έννοια της πολιτικής συνοχής και είναι επίσης σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανέλθει σε σχέση με το τι ακριβώς είναι η πολιτική συνοχής ε, και αυτό το λέω στο πλαίσιο των προθέσεων αναδιάρθρωσης. Δεν πρέπει να υπάρχει σύγχυση μεταξύ της Στρατηγικής Ευρωπαϊκή Ένωση 2020 και της Πολιτικής Συνοχής. Η στρατηγική για το 2020 ορίστηκε ως ε, πολιτική μακροοικονομική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επαφίεται στα κράτη-μέλη να την εφαρμόσουν. Αν τώρα ε, θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτήσει τη μία ή την άλλη πτυχή της στρατηγικής αυτής, πρέπει να δημιουργήσει νέους πόρους, αλλά όχι να ε, χρησιμοποιήσει κονδύλια τα οποία έχουν ε, δοθεί για την πολιτική συνοχή. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι η πολιτική συνοχή δεν γίνεται να είναι η πολιτική εφαρμογή στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020. Πρέπει η πολιτική συνοχή να συμμετέχει, όπως είπε και ο εισηγητής, ε, στην αύξηση απασχόλησης, στη μείωση της καθυστέρησης ανάπτυξη ορισμένων περιφερειών, την ενίσχυση των ε, πληθυσμών που είναι σε μειονεκτική θέση, όπως επίσης και αύξηση πλούτου για όσους μειονεκτούν. Κατά την άποψή μου λοιπόν δεν υπάρχουν άλλοι κεντρικοί στόχοι Τώρα για τους υπόλοιπους στόχους που θέλουμε να επιτύχουμε πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναφερθεί στις πόλεις που πρέπει να προχωρήσουν, να τους δώσει τη δυνατότητα να επενδύσουν στις ε, ε, νέες πηγές ενέργειας, ε, στην οικολογία, ε, σε προσεγγίσεις πιο φιλικές προς το περιβάλλον ε, και θέλω να ρωτήσω, μήπως πρέπει επιτέλους να βάλουμε όρους στις επιδοτήσεις της άμεσης προς επιχειρήσεις βάσει της απασχόλησης, της αποκέντρωσης, της μείωσης των θέσεων εργασίας, μήπως πρέπει να τεθούν τέτοιου είδους όροι. Απλώς θέτω το ερώτημα. Και για να είμαι και σύντομος δεν θα επιμείνω στο πρόβλημα της προστιθέμενης αξίας νομίζω ότι και ε, για το θέμα αυτό ε, μην εξειδανικεύουμε και την προστιθέμενη αξία. Πρέπει να την καταλάβουν ε, οι πολίτες μας ως προστιθέμενη αξία που τους δίνει τη δυνατότητα να προοδεύσουν και σε οικονομικό επίπεδο αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οικοδομήθηκε γύρω από ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης ε, ε, ε, ενιαίας αγοράς η οποία βάσει της ανταγωνιστικότητας δεν θα έπρεπε να αποκλεί τους ε, τους ε, πιο ευάλωτους ε, έξιμων. Πρέπει να προβλέψουμε την ενσωμάτωση όλων ώστε να είναι μια δίκαιη αγορά. Η πολιτική συνοχή είναι η μόνη ευρωπαϊκή πολιτική που μπορεί να βοηθήσει την επίτευξη του στόχου αυτού και δεν βασίζεται μόνο στην ανταγωνιστικότητα, την πάση φυσία ανταγωνιστικότητα. Επίσης, δεν πρέπει να καταστήσουμε κενές περιεχομένου τους στόχους της πολιτικής συνοχής, ακόμη και αν νέοι πολιτικοί στόχοι ή οικονομικοί στόχοι πρέπει να επιτευχθούν. Δεν πρέπει αυτό να ε, αποδυναμώνει τις βασικές ιδρυτικές αξίες που είχαμε κάποτε, δηλαδή αρμονική και ε, ίση εξέλιξη και ανάπτυξη για όλες τις ε, περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Euh, Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βόαν. Ευχαριστώ πολύ. Η γνωμοδότηση Επιτροπής Προπολογισμών ε, υποθέτω ότι ε, την γνωρίζει ο κύριος Πίπερ και βλέπετε ότι συμφωνούμε σε πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, ε, μπορούμε να συμφωνήσουμε τη μείωση του αριθμού των σφαλμάτων, διευκόλυνση των διαδικασιών, ε, ε, καλύτερη διαχείριση και επίσης είμαι υπέρ ενός ενιαίου συστήματος ελέγχου που βέβαια πρέπει να πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για παράδειγμα στην Ουαλία έχουμε ένα τέτοιο είδους σύστημα που μας δίνει τη δυνατότητα πολύ μεγαλύτερου ελέγχου όσον αφορά ε, τους λογαριασμούς και ενδεχομένως να πρέπει αυτό να επεκταθεί και στις περιφέρειες. Ένα ζήτημα που θα ήθελα να θέσω είναι αυτή η αυτόματη διακοπή των πληρωμών όταν ε, εμφανίζονται ατασταλίες ε, συστηματική διακοπή, λέει η Επιτροπή Προπολογισμών, γιατί αυτό ακριβώ αναφερόταν στην έκθεση για την απαλλαγή και νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια διαδικασία συγκεκριμένη που θα πρέπει να ακολουθείτε πριν ε, γίνουν οι πληρωμέ. Το άλλο θέμα είναι η επιλεξιμότητα, δηλαδή η σύνδεση των κυρώσεων με ε, τα μακροοικονομικά ε, στοιχεία, δηλαδή πληρωμές ε, διαρθρωτικών κονδυλίων στις χώρες που δεν τηρούν το Σύμφωνο Σταθερότητα και ανάπτυξη. Αυτό νομίζω όμως ότι πραγματικά επιβάλλει κυρώσεις στα κράτη-μέλη τελικά και στις συγκεκριμένες περιφέρειες και θα ήταν λάθος να γίνει κάτι τέτοιο. Ο κύριος Ντελεμπάρ το ανέφερε και στην παρουσίασή του. Θα θέλω να πω ότι η έκθεσή του μας βρίσκει σύμφωνους ε, ε, πολλά, τα, πολλά από αυτά που αναφέρονται ε, είναι σωστά. Ίσως θα έπρεπε οι όροι να έχουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο να είναι κάπως πιο στοχευμένοι. Εμείς συμφωνούμε με το αποθεματικό επιδόσεων για λόγους ευελιξίας και όπως ε, είπε και η Επιτροπή Περιφερειών είναι κάτι που μπορεί να διερευνηθεί περαιτέρω. Κάτι ακόμη όσον αφορά τη συνολική διάρθρωση. Νομίζω ότι είναι μια τεράστια συζήτηση για μας. Ε, εγώ συμφωνώ με το επίπεδο ε, του στόχου 1, 2 και 3 ώστε όλες οι περιφέρειες να μπορούν να κάνουν αιτήσει, να είναι επιλέξιμες για διαρθρωτικά κονδύλια. Μία από τις ιδέες που εξετάζεται είναι οι περιφέρειες που πηγαίνουν στο στόχο 2 για παράδειγμα να παίρνουν τα κονδύλια μαζί τους. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να διερευνηθεί περαιτέρω. Κάτι ακόμη που θα ήθελα να αναφέρω, οι αστικές περιοχές Ποιο είναι ακριβώ ο ορισμός και ποιο θα το ορίσει αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι περιφέρειε, τα κράτη-μέλη. Μέχρι τώρα είχαμε την εντύπωση ότι ο Επίτροπος μας είπε ότι το ορισμό στα κράτη-μέλη. Όμως ε, η απάντηση που μας έδωσε την τελευταία φορά που έθεσε εγώ το ερώτημα σε σχέση με τον ορισμό των αστικών περιοχών ε, ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να ε, επεξεργαστεί έναν αναρμονισμένο ορισμό των αστικών περιοχών. Δύσκολο αυτό και ενδεχομένως και να αποτελέσει, να δημιουργήσει σφάλματα γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο ορισμένα κράτη-μέλη να αποδεχθούν ένα κεντρικά ε, ε επιβαλόμενο στόχο της αστικής περιοχής και σωστά πρέπει και αυτό να το δούμε. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ, Σάνκελ. Κύριε Σκέλη. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα καταρχά να συγχαρώ τον Μάρκου, ε, εξαιρετική η δουλειά του. Όπω είπατε και εσεί, είναι προκλητική ή μη τι άλλο. Ή μη τι άλλο μα ε, δίνει πολύ τροφή για σκέψη. Και βέβαια τη λεπτομερή συζήτηση, το διάλογο που έχουμε τώρα. Θα ήθελα να συμφωνήσω προκαταβολικά ότι η πολιτική τη συνοχή δεν είναι αυτό ο σκοπό. Ναι. Θα πρέπει να εγγράφεται μέσα στου στόχου τη στρατηγική 2020 να τους εξυπηρετεί κατά κάποιον τρόπο, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κριθεί από το πώς σε νέα χρόνια θα έχουν υλοποιηθεί αυτοί οι στόχοι. Ε, αυτό πρέπει να είναι ο κύριος γνωμονάς των προσπαθειών μας και στην κοινοτομία και στα διευρωπαϊκά δίκτυα ε, και στην ενέργεια, σε όλα τα σημαντικά αυτά θέματα που μπορεί να προσφέρει προς θεμένη αξία η Ευρώπη. Επίσης συμφωνώ ότι μια προσέγγιση με γνώμονα το αποτέλεσμα έχει ζωτική σημασία και για τις αναλύσεις, για τις αιτήσει για τις αναλύσεις, για την αξιολόγηση, τον έλεγχο. Όσο, λιγότερη, όσο περισσότερη ε, εστίαση δίνουμε στο αποτέλεσμα και λιγότερη στην ε, γραφειοκρατία, τόσο το καλύτερο. Και έτσι νομίζω ότι μπορούμε τον στόχο της μείωσης της γραφειοκρατίας να τον εγγράψουμε σε αυτή την κατηγορία. Επίσης θα συμφωνήσω ως προς ε, την ε, Ε, θέση σχετική με το EGF που βλέπουμε πολύ συχνά στις ε, συνεδριάσεις μας και τις προφορίες που έρχονται από καιρού σε καιρό να μας ζητήσουν ε, είτε για την Πολωνία είτε για τη Σλοβενία η μία χώρα ακολουθεί την άλλη συνέχεια ως προς το EGF βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ρόλο στη συγκεκριμένη περίπτωση να διαδραματίσει επίσης ρόλο έχουν να διαδραματίσουν οι όμορες περιφέρειες με βάση προτάσεις του εισηγητή και νομίζω ότι η παράγραφος παριθμών 6 εκεί όπου λέει ότι υπογραμμίζει πως ε, η κοινότητα μπορεί να επιβιώσει στο πλαίσιο του, οικονομικού, του παγκόσμιου ανταγωνισμού μόνο εφόσον η πολιτική για τη συνοχή αξιοποίηση, το δυναμικό ανάπτυξη όλων των περιφερειών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 είναι πολύ σημαντικό. Για το ΑΕΠ βλέπω ότι δίνει υπερβολική έμφαση ο Μάρκο όπως και στην έκθεση της να επισημάνουμε ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη και τις επιπτώσεις αυτών στις υποπεριφέρειες της Ευρώπης και εν τέλει θα ήθελα να υπογραμμίζω, μάλλον να προσθέσω ακόμη ένα-δύο πράγματι, έφαση θα ήθελα να δω περισσότερες προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να τις βοηθήσουμε δηλαδή να αξιοποιήσουν, να έχουν πρόσβαση στις τα ταμεία, σε όλο το φάσμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γιατί διαρκώς λέμε πόσο σημαντικές είναι αυτές Διαρκώ υπογραμμίζουμε ότι αν μια μικρομεσα... κάθε μικρομεσαία προσλάμβανε έναν υπάλληλο, θα είχαμε λύσει το πρόβλημα τη ανεργία στην Ευρώπη. Άρα θα ήθελα περισσότερη έμφαση εδώ. Και επίση για το διαχρονικό τομέα, θα ήθελα να επισημάνω ότι οι πολίτε δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτή η πολιτική. Και αυτό διότι δεν δίνουμε αρκετή σημασία στην ορατότητα τη πολιτική στα κράτη-μέλη και τον τρόπο που μπορεί να έχουν πρόσβαση στα κονδύλια τα κράτη-μέλη. Και πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα από την πατρίδα μου υπάρχει μια κρατική υπηρεσία φως η οποία χρηματοδοτείται απευθεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει ιδέα κανεί για το τι είναι αυτή η εταιρεία, τι κάνει η υπηρεσία, ε, η εταιρεία του δημοσίου καλύτερα, τι κάνει, τι χρήματα παίρνει, πού τα χρησιμοποιεί. Θα ήθελα λοιπόν να απαιτηθεί οπουδήποτε υπάρχει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στον τίτλο του προγράμματο ή του έργου, να υπάρχει ή του έργου, να υπάρχει ο, η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η EU δηλαδή. Ευχαριστώ. παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Συγχαρητήρια στον Μάρκους για την εργασία του άριστης ποιότητας. Πολλά σημεία της έκθεσης ε, τα συμμερίζουμε. Ναι, μη χαμογελάς Μάρκο, αλήθεια λέω. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την πράγμα 50 λυπάμαι που είναι μόνο 50 εδώ, αλλά που λέω ότι ο προπολογισμό για το μετά το 2013 θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ο ίδιο με την σημερινή περίοδου. Η πολιτική συνοχή σε που δεν είδε θα πρέπει να υποφέρει από μια μείωση προπολογισμού. Ο Μάρκο Πίπερ είμαι σίγουρο ότι αυτό θα την περισπιστεί ιδιαίτερα γιατί είναι σημαντικό ουσιαστικό σημείο. Πέρα τώρα από αυτό το βασικό για τον προπολογισμό, συμφωνώ και με πολλά άλλα σημεία με τον εισηγητή. Ε, τη διαπίστωσή του τη συμμερίζομαι ότι η πολιτική συνοχή θα πρέπει να υποφεληθεί από τη δυνατότητα ανάπτυξη όλων των περιφερειών για να πετύχουμε του στόχου τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Επίση, συμφωνώ με τι προτάσει του για τη συγκέντρωση όσον αφορά τις πηγές της χρηματοδότηση εντάξει, και το εμπιστευτικό χαρακτήρα των βοηθειών και λυπάμαι που θα πρέπει να, να βοηθηθούν για οικονομικές, πολιτικές και ε, οικονομικές, κοινωνικές ε, μεταρρυθμίσεις. Τα πρώτα που σου είπα σε θουσίασαν, αλλά δεν μπορούσα να συνεχιστεί αυτό Μάρκος. Τέλος πάντων. Εδώ επίσης με την πράφο 9 για το επιχειρησιακό πρόγραμμα για γεωγραφικές μονάδες λειτουργικές πραγματικά. Αμφιβάλλει για για την προσθέμενη αξία αυτών των επιχειρησιακών προγραμμάτων εισηγητή. Και εγώ είμαι αντίθετο με εκείνον ε, μέσω ενό οδικού χάρτη ειδικού. Αυτέ ε, θα προχωρηθούν ε, και να πω ένα τυχαίο παράδειγμα. Η στρατηγική για την ε, Ατλαντικό, εκεί στην περιοχή αυτή, όπως ξεκίνησε από την Επιτροπή μας, επιχειρησιακό πρόγραμμα Ατλαντικός, που είναι ο καλύτερος δυνατό τρόπος για να δούμε τις στρατηγικές, τις προτεραιότητες αυτής της στρατηγικής. Και τα περιοχή προγράμματα έχουν το θετικό ότι είναι και νομικό μέσο, το οποίο έχει ήδη δοκιμαστεί και που το γνωρίζουν εκείνοι που το χρησιμοποιούν. τα υπόλοιπα για τη συνεργασία είναι οι λειτουργικές γεωγραφικές μονάδες δεν είναι τόσο ικανοποιητικέ γιατί πολλές φορές ε, είναι κάτι το αδρανές είτε υπάρχει κάτι το νέο σαν δομή που δεν το επιθυμούμε. Τώρα εμείς ε, θέλουμε να δούμε τα τρία όχι, όχι νέα θεσμικά όργανα, όχι νέος προϋπολογισμός, ε, όχι νέα νομοθεσία. Εντάξει συμφωνούμε πάνω σε αυτά τα τρία, ναι. Και τώρα τα επιχειρησιακά προγράμματα, το να καταφύγουμε σε αυτά είναι η καλύτερη λύση όσον αφορά τη σταθερότητα, την αποτελεσματικότητα, την επάρκεια, την νομιμότητα. Και είμαι στη διάθεση του εισηγητή για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για τα σημεία αυτά, τα διάφορα και σίγουρα η Επιτροπή μα θα πετύχει μια συμβαστική λύση που να μπορείτε δεχτούν όλοι πάνω σε αυτά τα θέματα που μα απασχολούν στην έκθεση μαζί μέσα και την ενδιάμεση κατηγορία ή τουλάχιστον, τουλάχιστον να δούμε μια κάποια οργάνωση ώστε οι υποφέρουσες ε, ε περιοχές από το κατόφλι του 90, το 75% να μπορούν να προτιμηθούν στα πλαίσια του στόχου 2. Αυτά και σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Ε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ζητήσω από τους μιλητές που θα πάρουν το λόγο να ε, ε, σεβαστούν τα δύο λεπτά γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να μιλήσουν οι τελευταίοι ομιλητές. Κυρία Κρέλ. Ναι, τώρα είναι σειρά μου. Θα ήθελα να ευχαριστώ ρητά τον εισηγητή. Είναι πράγματι πολύ καλή βάση συζήτηση αυτή η έκθεση, αφού έχω μόνο δύο, χρόνο, δύο λεπτά χρόνο, θα περιοριστώ σε τρία σημεία. Θέλω να σα υποστηρίξω ρητά στην μακροσκελή συζήτηση που κάναμε εδώ μέσα στην Επιτροπή ω προ το βασικό δίκτυο για το ΑΕΠ που θα πρέπει να προσδοριστεί. Ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη για την προσοχή περίοδο στήριξη. Ωστόσο, θα ήθελα σε περιφερειακό επίπεδο να επισημάνω ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν οι ιδιαίτεροι δείκτες, αλλά αυτή τη στιγμή μόνο με βάση το ΕΠ μπορούμε να δουλέψουμε. Τώρα, εάν θελήσουμε να καταργήσουμε το EGF, το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση δηλαδή, θα πρέπει να δούμε τι συνέπειες θα έχει αυτό. Εικονικό χρήμα θα προσθεθεί στο πραγματικό χρήμα αυτό θα είναι το αποτέλεσμα και αυτό ήταν το επιδιωκόμενο. Δεν νομίζω ότι είναι θα βγει τίποτα καλό από αυτό. Και επίσης θα συμφωνήσω προς τις αμφιβολίες που εκφράζεται. Αλλά βλέπω ότι όντως έχει η Επιτροπή ε, προσπαθήσει να προχωρήσει προς την κατάργηση, τη σταδιακή μάλλον έξοδο ορισμένων περιφερειών από την στήριξη. Αυτό είναι μια λύση την οποία δεν νομίζω ότι πρέπει να καταδικάσουμε. Ε, θα πρέπει να δούμε βέβαια αν η Επιτροπή όντως σκοπεύει να καταργεί σταδιακά αυτή την υπαγωγή, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε επι, ε, επαόριστον ή διαβίου ε, ιστοδιενικές καλύτερα υπαγωγή των περιφερειών αυτών ε, στην στήριξη. Ε, αν πούμε τώρα ότι πρόκειται για κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες που έχει προκαλέσει η κρίση, είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά πάντως θέλουμε να δούμε πώς θα βγουν από, την, από, την, από τους στόχους αυτές οι περιφέρειες. Ευχαριστώ. Κορνέλια. Jetzt. Zunächst erst einmal Berichterstatter. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστώ τον εισηγητή. Υπάρχει μια σειρά από πράγματα που ε, μας βρίσκουν σύμφωνους. Ε, για τα νέα θεματικά ταμεία, Φερρυπίν, για την ε, διασταυρούμενη χρηματοδότηση έρευνα και κοινωνικό ταμείο θα πρέπει να καταστεί πιο εύκολη, είναι δυνατότητα που θα πρέπει να μας θέσει να προσφέρουμε που βλέπουμε κάποια σημεία που χρειάζεται περισσότερη συζήτηση. Ε, ζητάτε την ενίσχυση του στόχου 2, περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση. Ε, θα ήθελα να ξέρω ακριβώς τι εννοείτε με αυτό. Θέλετε μια καλύτερη πρικοδότηση, θέλετε πιο αποτελεσματική λειτουργία αυτού του στόχου. Γιατί αυτό μπορώ να το δεχθώ, αλλά αν σημαίνει ότι πρέπει να ενισχυθεί και να διευρυνθεί ο στόχο, δεν θα συμφωνήσω. Ε, για το στόχο 3 όμως τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά γιατί λέτε ότι υπάρχει αύξηση στο 7%. Μπορεί να είναι κάπως ελκυστική αυτή η ιδέα γιατί και εγώ ε, προέρχομαι από μια περιοχή που έχει πολλές σχέσεις με την Πολωνία και την Τσεχία. Βλέπω ότι υπάρχει ε, κάποια βάση σε αυτή την ιδέα. Αλλά πώς καταλήγουμε στον υπολογισμό του 7%, πώς καταλήγεται εκεί και από πού θα βγουν τα χρήματα. Θεμεί το ερώτημα νομίζω. Επίσης, ε, εμείς είμαστε υπέρ των μεταβατικών διατάξεων μάλλον παρά των ενδιάμεσων κατηγοριών. Άρα θα πρέπει να ε, επισημανθεί με κάποιο τρόπο ότι αυτή η ενδιάμεση χρηματοδότηση δεν θα είναι και ε, αιώνια. κατάσταση. Καθιστάται λοιπόν σαφέ ότι υπάρχουν κάποιε περιφέρειε οι οποίε βγαίνουν σιγά σιγά από τη στήριξη. Καλό θα είναι ότι αυτή η περιπτώση να είναι η, η λύση, όχι η ενδιάμεση κατηγορία, αλλά οι μεταβατικέ διατάξει. Επίση η αρχή τη υπαγωγή σε προποθέσει, conditionality. Η πολλαπλή υπαγωγή σε προποθέσει. Ε, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να απορρίπτεται αυτή η ιδέα της ε, υπαγωγής σε όρους, αλλά θα πρέπει να είναι ουσιαστική αυτή. Στο 37 το αναφέρεται. Επίσης ε, στο 51 υποβολή πρόταση για την καθιέρωση αυστηρότερων αυτόματων εφαρμογών κανόνων για το και εκεί συμφωνώ απολύτως. Το βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό. Στο 60 βλέπουμε ότι θα ήταν ε, βεβαίως ε, δύσκολο όταν υπάρχουν περιπτώσεις υπέρβασης ικανότητας απορρόφησης κοινότητας για την πολιτική συνοχής ε, να συνεχίσει η πολιτική στον τρέχουσα υπολογισμό των δημοσιονομικών συνεπειών. Αυτά όλα πρέπει να τα ξαναδούμε λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, Ερμήνια. Ευχαριστώ. Θα ήθελα όπως και οι υπόλοιποι να εκφράσω την εκτίμησή μου για την εργασία του κυρίου Πίπερ και συμμερίζομαι κυρίως την προσπάθεια του να διατηρηθεί η πολιτική συνοχής με την προσοχή τη περισσότερη στις ασθενέστερες περιοχές και τις πιο απομακρυσμένες και ακολουθώντα βέβαια ε, στρατηγική 2020 που κατά την άποψή μου θα πρέπει να αποτελεί μέρος της πολιτικής συνοχής και με μια προσπάθεια και αυτό το κατορθώνει με την πρόταση που διατυπώνει μια προσπάθεια ακριβώς απλούστευσης συγκέντρωσης ταυτόχρονα και μεγαλύτερης διαφάνειας επίσης σε όλη τη γραφετική οργάνωση της πολιτικής συνοχής. Διάφορα σημεία όμως με βρίσκουν αντίθετη ή τουλάχιστον αμφιβολίες μου προκαλούν, μου δημιουργούν. Θα τα πω στον συνάδελφο Πίπερ για να μου πει και εκείνο την άποψή του. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, το ΑΕΠ σαν κύριο κριτήριο καταλαβαίνω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να βρίσκουν τα εθνικά τους κριτήρια, εθνικούς δείκτες. Θα πρέπει όμως να καταλάβουμε πώς τους βρίσκουν αυτούς τους δείκτες και να διευκρινίσουμε ότι αυτή η προσθήκη εθνικών δείκτων δεν θα δημιουργήσει μια μεταφορά από τον ένα στόχο στον άλλο, ένα παρόμοιο πέρασμα. Και μετά υπάρχει και μια κάποια αντίθεση ε, ίσως και ε, λίγο που να μοιάζει ανάμεσα στους στόχους. Ο πρώτος στόχος λέει ότι θα πρέπει να διατηρηθεί ο πρώτος στόχος στο σύνολό του και ενισχυμένο. Δεν χρησιμοποιεί το όρος ενισχυμένο, αλλά αυτό εννοείται. Το ίδιο για τους στόχους 2 και 3 στα πλαίσια μιας πολιτικής που θα πρέπει να υπερασπιστούμε γιατί υφίσταται επιθέσεις και υπάρχει φόβος για περικοπές. Ε, δεν μπορούμε όμως να φανταστούμε ότι θα ε, ενισχύσουμε και τους τρεις στόχους, λοιπόν θα πρέπει ο καθένας στόχος να υποστηριχθεί σύμφωνα με τη σημασία του και να μην ε, αυτό για την διάμεση κατηγορία το σημεριζομαι, μάλλον καλύτερα να βρούμε το phasing out, την μη συμπερίληψη ακριβώς. Ακόμα κάτι το σημαντικό είναι οι προϋποθέσεις, εντάξει, υποπροϋποθέσεις σωστό αυτό ότι θα πρέπει να προβλέψουμε αυτό το προϋποθέσεις αλλά χρειάζεται να διευκρινίσουμε για κάτι άλλο. Αυτές οι προϋποθέσεις θα πρέπει να αναφερθούν λεπτομεριακά εκ των προτέρων πριν από τον όλο προγραμματισμό για να αποφύγουμε στη συνέχεια να δημιουργηθούν προβλήματα σύμφωνα με τα προγράμματα τα οποία έχουν ήδη εφαρμοστεί. Κάτι τελευταίο να πω ότι κάπως μπερδεμένη με όχι αντίθετη τόσο, αλλά μπερδεμένη σχετικά με το σημείο 51 για τις κυρώσεις. Δεν είναι σαφής η διατύπωση. Ο κ. Πίπερ τι θέλει να πει με αυτό. Ζητάει μια ρύθμιση διαφορετική με κυρώσεις μόνο για τις ε, περιφέρειες που δεν σέβονται είτε προβλέπει έτσι ε, σταδιακές κυρώσεις για να ε, πετύχουμε και την αποτελεσματικότητα την οποία ψάχνουμε να πετύχουμε ακριβώς. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω επίσης τον εισηγητή μας ε, και να του υποβάλω ορισμένες ερωτήσεις για να με ευκρινίσει πράγματα. Όταν μιλάει για το ρόλο αυτό των, ε, αυτών των ταμείων, αυτών των κονδυλίων από στα πλαίσια του κοινωνικού ταμείου αυτό το γενικό τι, που αναφέρεται στην ε, συνδυασμό των δύο και τη συνοχής και του περιφερειακού γίνεται αυτό να συνδυαστούν αυτά δύο ποσά, να συγχωνευτούν. Και ακόμα κάτι που ρώτησαν επίσης και μερικοί προηγουμένως όταν ακριβώς αναφέρεται αυτό το ποσοστό, το 7% στο 24% για τον στόχο τον περιφερειακό της συνοχής, γιατί αυτό το ποσοστό και όχι ένα διαφορετικό. Όταν μιλάμε επίσης για συγχρηματοδότηση, λέμε το το ποσό στο 75% ποσοστού σε σχέση με το σημείο 41. Αυτό το 75% και γιατί όχι, ας πούμε από το 75% μέχρι το 80% αυτό το περιθώριο όπως μέχρι τώρα και ακόμα ένα σημείο όταν μιλάμε για στους, τους αναγνωρισμένους δρόμους, τους ευρωπαϊκούς, ε, ταξινομημένους, αναγνωρισμένους, ε, τι είναι αυτοί στο οποίο αναφέρεται ο εισηγητής. Και στο 14 όταν μιλά για την ενέργεια που βασίζεται σε αποτελεσματική ε, μέθοδο εναποθήκευσης της περιφέρειας. Τι γίνεται εδώ, έχουμε τη συγκεκριμένη γερμανική περίπτωση, μήπως θα μπορούσε να μας εξηγήσει τι σημαίνουν όλα αυτά. Επίσης, η στρατηγική του 2020 είναι βέβαια κάτι το πολύ σημαντικό, αλλά σύμφων, σίγουρα η στρατηγική συνοχή βοηθάει το 2020, αλλά είναι και κάτι παραπάνω, πολύ περισσότερο από το 2020 τη στρατηγική αυτή. Και τι θίγεται με τις περιοχές phasing out, τι θα γίνει με τις περιοχές αυτές αν δεν έχουμε έχουμε μια ενδιάμεση κατηγορία όπως την Ισπανία, τότε θα είχαμε πόλεις που θα συγκλίνουν προς τα εκεί. Τι θα κάνουμε με αυτές τις περιφέρειες. Αυτό θα είναι κάτι μεταβατικό, Τι ακριβώς θα είναι. Μήπως θα μπορούσαμε να αναφερθούμε περισσότερες λεπτομέρειες πάνω σε αυτό το σημείο. je... Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ δεν συμφωνώ με την άποψη του γιατί έχουμε σοβαρέ διαφωνίε σε σχέση με του στόχου τη πολιτική συνοχή, αλλά θα αρκεστώ στο αναφερθώ στα βασικά σημεία. Πρώτον, θα ήθελα να πω ότι διαφωνώ καθέτο ε, με κάθε μορφή επιλεξιμότητα που σημαίνει ότι θα υπήρχαν οικονομικέ ηρώσει για τι τοπικέ αρχέ. Ε, θα ήταν άδικο για τις τοπικές αρχές ε, για λόγους, για παράδειγμα, μη εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης παρά το γεγονός ότι αυτό δεν ε, είναι δική τους αρμοδιότητα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα έπρεπε να επιμείνουμε στο γεγονός ότι η αρχή της θεματικής συγκέντρωσης δεν θα έπρεπε να γίνει όπως με το earmarking σήμερα ένα πρόβλημα αποτελεσματικότητας πολιτικής συνοχής. Πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και ρεαλιστές για να μπορέσουμε να, να είμαστε επιτυχείς. Όσον αφορά τον, τις, τους δείκτες πρέπει να είναι η καρδιά του προβλήματος για την επόμενη πολιτική συνοχή, γιατί έχει να κάνει και με το θέμα της επιλεξιμότητας, αλλά και με το θέμα της ε, αναθεώρησης. Το να πάμε πέρα από το ΑΕΠ ε, είναι ένα, θα ήταν ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο ε, προς την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Θα ήθελα επίσης να πω ότι διαφωνώ καθέτος με τα επιχειρήματα του εισηγητή σε σχέση με τις ενδιάμεσες περιφέρειες. Θα πρέπει να υπενθυμίσω τη δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε συγκεκριμένες περιφέρειες βάσει του 149 και 349 της συνθήκης της Λισαβόνας για την ε, συμβολή των χωρών αυτών, για τη συμμετοχή τη των χωρών αυτών, των περιφερειών αυτών σε, στην κοινοτική αγορά. και αναφέρομαι κυρίως ε, στις άκρος περιφερειακές, ε, στις άκρος ε, απόκεντρες περιφέρειες και τα σχετικά κονδύλια. Όσον αφορά τώρα την, τα, από, τις, τα αποκεντρωμένα στοιχεία, αυτό θα δώσει τη δυνατότητα ε, βιώσιμων ε, ε, αναπτυξιακών προγραμμάτων που θα είναι επωφελής όχι μόνο για τις άκρως περιφερειακές, για τις άκρως απόκεντρες περιφέρειες, αλλά για όλους. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, για τη γενική αυτή έκθεση, θέλω να πω κύριε Πίπερ, ότι απέχει λιγότερο θα έλεγα από αυτό που περίμενα από τις θέσεις μας. Και άρα νομίζω μπορούμε να συζητήσουμε. Υπάρχουν κάποια θέματα στα οποία δίνεται ιδιαίτερη ιδιαίτερη έμφαση ως προς την ε, προβολή στον προγραμματισμό των περιφερειών, τις μακροπεριφέρειες, το στόχο 3, τις ε, άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες, θεματολογίες οι οποίες καταστρέφουν το οικοδόμα της συνοχής και την οριζόντια προσέγγιση κάθε σε κάθε περιφέρεια, όλα αυτά τα βρίσκω θετικά. Υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία χρειάζεται συζήτηση περαιτέρω διότι υπάρχουν επιχειρήματα που μπορούν να προβληθούν για να πείσουμε τους μεν και τους δε και η Επιτροπή των Περιφερειών έχει επιχειρήματα. Ο κύριος Στελοπά μας είπε ότι υπάρχει ζήτημα αξιοπιστής αλλά και ευελιξίας, γιατί όχι. Και έχοντας συστήσει με τον Επίτροπο Χάν, βλέπω ότι αυτή η ιδέα είναι λίγο πολύ ιδέα ευελιξίας για να μην είμαστε στην κατάσταση του 2008 με μια ανάγκη για ανάκαμψη και διάθεση κονδυλίων για την ενεργειακή, για την προμήθεια σε ενέργεια. Ιδιαίτερα να περάσουμε σε περίοδο προγραμματισμού 5 συν 5 ετών. Πιο μακροπρόθεσμα δηλαδή. Άρα θα πρέπει να έχουμε στο δυνατόν πιο εις ανάλυση. Για τι ε, ενδιάμεσε περιφέρειες θα ήθελα να αναφερθώ. επίση. για να πω ότι δεν θέλουμε ομοιομορφία, θέλουμε μια σταδιακή έξοδο. Βεβαίω το 75% είναι πολύ πιο εύστοχη επιλογή από την 90%. Και η μείωση σταδιακή των ενισχύσεων δεν είναι μόνο οικονομικού χαρακτήρα, αλλά και του πεδίου εφαρμογής πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης. Σιγά σιγά αυτή θα περιστέλλεται. Εάν όμως έχουμε μια περιφέρεια από αυτές η οποία αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αναδιάρθρωσης μιας ε, βιομηχανίας, ε, ενό εργοστασίου και χρειάζεται να στηριχθεί ο κόσμο που θα βγει στην ανεργία, εκεί πέρα θα πρέπει να δώσουμε έμφαση. Δηλαδή αυτό επιτρέπει ω σύστημα ε, περιφέρεια η οποία σήμερα αντιμετωπίζει μια κρίση. Απρόβλεπτη πιστεύω μέχρι πρόσφατα, όπως φέρει επίσης στην Ιρλανδία, να βοηθηθεί για να βγει αν όχι αλόβητη, γιατί δεν είναι δυνατό αυτό για όλε τι περιφέρειες τη Ιρλανδία ή με τι άλλο, αλλά πάντω με, τη στήριξη τη Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη να πέσει στα μαλακά ή να μην πέσει από τόσο ψηλά και πάντως να σηκωθεί τα πόδια της πιο, πιο γρήγορα. Αυτό θα είναι ένα εργαλείο για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Ευχαριστώ κυρία Σρότερ. Ας συνεχίσω λοιπόν και εγώ σε αυτήν την ιδέα. Ας μην επαναλάβω τα όσα είπε ο Φρανσουά εξ ονόματος ομάδας μας. Ήδη και χθε τα συζητήσαμε. Έχει νόημα νομίζω να τα σκεφτούμε πιο προσεκτικά αυτά τα πράγματα και να καταστήσουμε σαφές ότι αυτή η ενδιάμεση κατηγορία έχει χαρακτήρα μεταβατικό. Μεν, αλλά ταυτόχρονα και για λόγου δικαιοσύνη, θα πρέπει όλες τι περιφέρειες να την χάνουν τις ιδίες μεταχείρισης, και στο phasing in και στο phasing out. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν περιφέρειες οι οποίες έχουν αντιμετωπίσει σοβαρέ ε, ζημιές. και γι' αυτό θέλουμε να είναι σαφέ ότι χάρη στην ευρωπαϊκή στήριξη θα μπορέσουν πιο γρήγορα να βγουν από την κρίση. Αυτό σημαίνει phasing in και phasing out. Θα ήθελα πάντω να πω ότι είναι πολύ καλή διάρθρωση της έκθεσης, της μας βοηθάει στη δουλειά μας, είναι ευανάγνωστη. Βέβαια έχω και, την, ε, το επιπλέον πλεονέκτημα εγώ τη ε, γερμανικής. Μπορώ να διαβάσω δηλαδή το πρωτότυπο κείμενο. Και εκεί μπορώ και να κάνω τις παρατηρήσεις μου βλέποντας αν συμφωνώ απολύτω με τη διατύπωση ή όχι. Όλα αυτά λοιπόν ως προς τη δομή κτλ. Ως προς το περιεχόμενο θα το έλεγα κάπως old fashioned, δηλαδή είναι στραμμένο προς τα πίσω, προς το παρελθόν. Κοιτάει τι υπήρχε μέχρι τώρα, αλλά αυτά που υπάρχουν μέχρι τώρα δεν μπορούν να διαφυλαχθούν, δεν μπορούν να διατηρηθούν, γιατί έχουμε διαφορετικές καταστάσεις. Έχουμε κρίσεις, έχουμε κρίση περιβαλλοντική, ε, κλιματική μάλλον, έχουμε κρίση ε, οικονομική, έχουμε στρατηγική του 2020 που ακόμη δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή, άρα όλα αυτά πρέπει να αποτελέσουν τα στοιχεία με βάση τα οποία θα διατυπωθεί το κείμενο και ως εκ τούτου θα κάνουμε τις σχετικές τροπολογίες. Θα ήθελα μια σύγχρονη πολιτική για, τις, ε, για τη διαρθρωτική πολιτική στην Ευρώπη και στοχευμένη πολιτική. Άρα θα πρέπει και να ομολογήσουμε την πικρή αλήθεια ότι ο στόχος 2, παλαιότερος, δηλαδή απασχόληση ανταγωνιστικότητα, ίσως να χρειαστεί να του βρούμε και κάποιο πιο συμπαθητικό όνομα. Εν πάση περιπτώσει όμως, με βάση την ορολογία της Επιτροπής, ε, θα πρέπει αυτός ο ρόλος ε, της ε, γέφυρας που παίζει αυτός ο στόχος να ξαναεφευρεθεί, να ξαναδιατυπωθεί για να μην λησμονούμε τις προτεραιότητες της Ευρώπης του 2020. Κάνει μια πολύ κομψή πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή λέει ότι υπάρχουν προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτέ αυτές οι περιφέρειες στόχου 2 που έχουν τον ρόλο της γέφυρας χρηματοδοτούνται επειδή εξυπηρετούν τις προτεραιότητες του 2020. Ναι, αλλά αυτό θα πρέπει να ισχύει και για τους μεγαλύτερους και για εκείνους που ακόμη έχουν προβλήματα και πρέπει να τα λύσουν. Είναι πολύ καλή η ιδέα αυτή. Πρέπει να την προωθήσουμε, πρέπει να επεξεργαστούμε περισσότερο και να μην περιοριστούμε μόνο στην τρέχουσα περίοδο στήριξη, αλλά να προβάλλουμε τα πιο προοδευτικά στοιχεία τη πρόταση τη Επιτροπής, πράγμα το οποίο δυστυχώ δεν βλέπω στην έκθεση τόσο όσο θα το ήθελα τουλάχιστον. Θα ήθελα να αντικατοπτρίζει περισσότερο τι προτάσει που έχουμε δει από το έγγραφο τη Επιτροπή, να τι καταγράφει και να λέει «Καλό αυτό, σύγχρονη προσέγγιση, μοντέρνα ιδέα ή αυτό και εκείνο δεν μα αρέσουν και θέλουμε να τα τροποποιήσουμε. Ασφαλώ θα χρειαστεί να κάνουμε πολλέ τροπολογίε, τουλάχιστον εμεί από την ομάδα μα, που έχω αναλάβει εγώ το συντονισμό, ξέρω ότι θα είναι πολλέ οι τροπολογίε και περιμένω βέβαια τι τις συζητήσει τι συμβαστικέ. Ευχαριστώ. Thank you, Elizabeth. No, no, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σασίερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στον συνάδελφο Πίπερ για την εργασία του, για την έκθεση που υπέβαλε. Επίσης της Έρικας, με τα λόγια της Έρικας συμφωνώ. Έγινε μια σαφή σύνταξη πάντως του κειμένου. Είτε κανείς συμφωνεί είτε όχι αλλά είναι ιδιαίτερα σαφής και συγκεκριμένη όλα με επιχειρήματα το ένα το άλλο, είτε συμφωνούμε λοιπόν είτε όχι. Δεν υπάρχει μεσαίος δρόμος, κανείς δεν κρύβεται πίσω από δέντρα και δεντράκια, είναι σαφή συγκεκριμένη η άποψή του. Με το πέντε συμφωνώ που μιλάει ο Μάρκος για ε, μειονεκτικές περιοχές, ε, ιδιαίτερα απόμακρε και άλλες με δυσκολίες και αντιμετωπίζουμε πάντω και κάποιες δυσκολίες εκεί που λέει ότι ίσως θα μπορούσε να υπάρξει μια συγχώνευση των δύο ε, ποσών των δύο ταμείων και θα πρέπει να δούμε και να σας αναφέρω και εγώ την ανησυχία που με διακατέχει για περιφέρειες που περνάνε από τον ένα στόχο στον άλλο από τη σύγκληση προς την, ε, την... Ε, τη στην απασχόληση και ανταγωνιστικότητα. Αυτό είναι πάνω από ένα ποσοστό του ε... κοινωνικού μεσοόρου και βλέπουμε ότι οι κοινωνικές ενισχύσεις μειώνται τρομερά, κάτι που δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα. Και αυτά είναι ακόμα πιο άσχημα γιατί, εντάξει αυτή είναι η απόψή μου, Υπάρχει ένα παράδεξο εδώ στην πολιτική συνοχή. Υπάρχουν περιοχέ που επεφελούνται ιδιαίτερα από τα ποσά αυτά, από τα κονδύλια αυτά και βοηθούνται και σημειώνουν πρόοδου. Και από τη στιγμή που πετυχαίνουν αυτέ τι πρόοδου, τι κάνουν, του τους περικόπτουν τα κονδύλια. Άλλε που δεν είναι αποτελεσματικέ, δεν ξέρουν να εργαστούν σωστά, δεν μπορούν να εργαστούν σωστά. Και αυτέ εντάξει επιβραβεύονται και θα παίρνουν τα στόχο του, μάλλον θα παίρνουν τα λεφτουδάκια του παραμένοντα τον ίδιο στόχο και όποιος ε, δεν εργάζεται καλά αυτός επιβραβεύεται έτσι και δυστυχώς ε, ε, είδαμε στην έκθεση της Επιτροπής Περιφερειών του 2010 που προέβλεπε μεταβατικές περιόδους εδώ στην πέμπτη έκθεση αναφέρεται η δημιουργία μιας νέας κατηγορίας ώστε να είναι εύκολη η μετάβαση ανάμεσα δύο κατηγορίες και να υπάρχει μια αντιμετώπιση καλύτερη ανάλογα με το ποσοστό ανάπτυξη. Ο Μάρκο Πίπερ στην εκθεσή του δυστυχώ θεωρεί ότι η κατηγορία αυτή η ενδιάμεση είναι ενάντια στην πολιτική συνοχή και γι' αυτό ακριβώ απορρίπτει την ενδιάμεση περιοχή. Στη Μαδέρα μέχρι το 2010 πήρε ένα δισεκατομμύριο ευρώ και είχαμε το 41% παλιότερα του ΑΕΠ και το 2009 πήγαμε στο 105 του κοινοτικού μεσουόρου. Από το 41 πήγε στο 105. Αυτό είναι πολύ απτό αποτέλεσμα. Ήταν πραγματική αυτή η ανάπτυξη ανάμεσα στο 2007 και στο 2000... Ε, τι γίνεται, ε, ε, τότε θα παίρνει από το 2013 και μετά μόνο 700, χάνει το 30% και πάνω. Εάν δεν υπάρχει αυτό το phasing, το phasing out, εάν διατηρηθεί αυτό που ισχύει σήμερα, αν δεν υπάρξει αυτή η διάμεση κατηγορία, ποιες λύσεις διαθέτουμε εμείς για να αποφύγουμε αυτή την αρνητική επίπτωση στο πέρασμα από τη μία κατηγορία στην άλλη, από τη στιγμή που θα περικοπούν απότομα κονδύλια και δεν θα τα λαμβάνουν πια αυτές οι περιφέρειες που πέτυχαν πολλά πράγματα. Ευχαριστώ. Thank you. Teresa Sanchez-Schmidt. Ε, Σμιτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Μάρκους ε, για τη διάσταση που έδωσε στην ε, έκθεση του. Συμπεριέλαβε τις βασικότερες πτυχές της πολιτικής συνοχής. Χρειαζόμαστε μια πολιτική συνοχή ευρωπαϊκή που μειώνει τις ανισότητες, που είναι ολοκληρωμένη, που είναι απλή, που είναι ορατή, που ενισχύει την συνεργασία σε τοπικό επίπεδο. Θα ήθελα να επιμείνω στο 6. Χαίρομαι ιδιαίτερα που καταλαβαίνει τη σημασία της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας του στόχου 3 και είναι υπέρ της αύξησης ε, ε, της χρηματοδότησης όπως την έχουμε άλλωστε ψηφίσει ε, Επίσης θα ήθελα εντάχει να αναφερθώ και στη σημασία των επενδύσεων στα μεγάλα διασυνοριακά προγράμματα όπως για παράδειγμα τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Ε, βέβαια, ας μην απορροφήσουν όλα τα κεφάλαια ε, των τα διασυνοριακά γιατί έχουμε και άλλους στόχους να επιτύχουμε σε αυτό το πλαίσιο. Επίσης, ε, ε, η πολιτική συνοχή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και ε, με την πολιτική συνοχή στο σύνολό της ε, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να, να μας απασχολεί όλους για το μέλλον της πολιτικής συνοχής ώστε να είναι πιο δίκαιη, να βοηθήσει περισσότερο τις περιοχές που έχουν περισσότερα προβλήματα γιατί δεν έχει νόημα μία περιοχή να είναι επιλέξιμη για περισσότερη χρηματοδότηση αν δεν έχουμε σκοπό να πετύχουμε την ισότητα, μεγαλύτερη ισότητα των περιφερειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ε, υπάρχει μια ενδιάμεση κατηγορία η οποία θα λάμβανε καλύτερα υπόψη τις περιοχές που καθυστέρησαν στην ανάπτυξή τους και έχουν διαρθρωτικά προβλήματα. Ε, το phasing out κατά τη γνώμη μου είναι δύσκολο γιατί υπάρχει περίπτωση να μειώνεται η χρηματοδότηση κάθε χρόνο, δεν θα υπάρχει δημοσιονομική σταθερότητα και θα με δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα στον πολυετή προγραμματισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ η Ελίσσα Ρόλερ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Επιτροπή καλωσορίζει βέβαια το σχέδιο εκθέσεως του κυρίου Πίπερ Ιδιαίτερα υποστηρίζουμε, καλωσορίζουμε τις γενικές αρχές και προσανατολισμούς προς το μέλλον της πολιτικής συνοχής που περιγράφονται ε, με βάση βέβαια και την πρόταση για την πέμπτη έκθεση συνοχής, ε, θεμενή αξία της πολιτικής συνοχής πάνω απ' όλα. Και θα ήθελα πολύ σύντομα να αναφερθώ στην ενδιάμεση περιφέρεια, στην ενδιάμεση κατηγορία περιφέρειας που από ό,τι βλέπω απασχολεί σε μεγάλο βαθμό τη συζήτηση σήμερα. Δεν πρέπει λοιπόν να διευκρινίσω τους λόγους για τους οποίους θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να συμπεριληφθεί αυτή η κατηγορία στα συμπεράσματα της πέμπτης έκθεσης συνοχής. Πιστεύει η Επιτροπή ότι χρειάζεται ένας μηχανισμός δίκαιος και πιο διαφανής για τις συγκεκριμένε αυτές περιοχές, περιφέρειες, διότι διαπιστώνονται κάποιες, ε, κάποια προβλήματα στις περιφέρειες αυτές που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν δυσλειτουργίες, όπως σε παραδείγματι περιφέρειες με αντίστοιχα επίπεδα ανάπτυξης που όμως τη χάνουν διαφορετική αντιμετώπιση στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, διαφορετική ένταση ενισχύσεων, διαφορετικοί στόχοι, διαφορετικοί κανόνες περί υπαγωγής, προϋποθέσεις δηλαδή για το πεδίο παρέμβαση ε, των κονδυλίων και όσο και το θεωρούμε ότι ένα σύστημα πιο απλό και πιο δίκαιο, πιο ισοδίκαιο θα μας βοηθήσει και θα επιτρέψει τις περιφέρειες, τις περιφέρειες που για λόγους διαφορετικούς, ιστορικούς ή άλλους ε, έχουν καταλήξει σε δύο διαφορετικούς στόχους να τύχουν μιας πιο δίκης και απλής στη διατυπώση της μεταχείρισης. Αυτά ως εξήγηση των λόγων για τους οποίους θεωρούμε ότι αυτή η, ενδιάμεση κατηγορία η νέα ενδιάμεση κατηγορία περιφερειών είναι σύμφωνη σε μεγάλο βαθμό των βασικών αρχών της πολιτικής μας, της αλληλεγγύης, της μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ όλων των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γιατί θεωρούμε ότι ένα σύστημα με περιφέρειες που θα έχουν αντίστοιχο επίπεδο ανάπτυξης ε, δεν θα πρέπει να επιτρέπει διαφορετική μεταχείριση. Ευχαριστώ πολύ. Μάρκους, θα ήθελες να πεις δύο λόγια για να καταλήξουμε. Έχω πέντε λεπτά τουλάχιστον. Όχι. Ε, απλώς τρως χρόνο από τους άλλους, από το άλλο θέμα, ροκανίζεις. Πολλές προτάσεις, πρόεδρε, πολλές ιδέες. Ενδιάμεση κατηγορία, λοιπόν. Έχουμε πρόσφατα την, ε, τους εορτασμούς ε, των ε, συνθήκων φιλίας μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Και δεν ήθελα να πω και εγώ ότι ιδιαίτερα υποστηρίζω τις δημοκρατικές διαδικασίες. Εάν λοιπόν η κρατούσα γνώμη εδώ είναι ότι πρέπει να υπάρξει αυτή η ενδιάμεση κατηγορία, ασφαλώς θα βρούμε μια συμβαστική λύση. Για την κυρία Κρέιλ. Να τύχουν μεταχείριση αντίστοιχες, αντίστοιχες με αυτές των περιφερειών phasing out, έστω, αλλά τότε μόνο άπαξ θα δοθεί αυτή η δυνατότητα. Δεν θα μπορούσε δηλαδή να είναι δι, στο διγυναικές η μεταχείριση αυτή. Ίσως με μια οριζόντια προσέγγιση του στόχου 2 ή άλλες ιδέες, γιατί υπάρχει υλικό, μπορούμε να αναπτύξουμε περισσότερο. Στόχος 3, 7%. Με ρωτήσατε από πού βγαίνουν τα λεφτά. Θα ήθελα να πω ότι ναι, χαιρόμαστε πολύ καλά όταν κάποια και πολύ καλά όταν κάποια περιφέρεια αναπτύσσεται, όταν στην επόμενη περίοδο στήριξης χρειάζεται λιγότερα κονδύλια. Φυσικά, ζήτω. Και θα προσπαθήσουμε ενδεχομένω να βρούμε λύσεις για το τι θα κάνουμε τα χρήματα αυτά. Αλλά όχι να τα χώσουμε κάπου ντε και καλά, να τα χρησιμοποιήσουμε εκεί που έχουν πράγματι νόημα. Και αν έχει νόημα αυτή η ενδιάμεση περιφέρεια, ε, κατηγορία περιφερειών, εάν πράγματι βλέπουμε ότι βοηθά την περιφερειακή πολιτική της Ευρώπης, ας το δούμε. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν αρκετά χρήματα με το 7% που θα πρέπει να είμαστε θέσει να χρηματοδοτήσουμε. Πρόσθετο ε, κριτήριο για το ΑΕΠ. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο η συζήτηση είναι ανοιχτή ακόμη. Ζητώ συγγνώμη στους συναδέλφους, δεν θα αναφέρω ονόματα επιμέρους και τις παρατηρήσεις του καθενός για να δώσω απάντηση χωριστά. Μόνο, μόνο εξαίρεση τον κύριο Ντελμπάχ και την Επιτροπή των Περιφερειών. Γιατί δεν έχω χρόνο βέβαια. Βλέπω μια έκθεση της Επιτροπής των Περιφερειών όπου δεν ζητάτε ενδιάμεσο στόχο στο παρελθόν. Έτσι. Τώρα, στη γνωμοδότηση για τη δική μου έκθεση, λέτε προτείνει να εξεταστεί η δυνατότητα ίδρυσης μιας νέας ενδιάμεσης κατηγορίας. Δηλαδή, είναι διαφορετική η στάση σας τώρα. Βλέπω ότι αυτή η πρόταση αλλάζει με βάση και τις τροπολογίες που κατατέθηκαν στη γνωμοδότησή σας. Άρα υπάρχουν εξελίξεις. Αντίστοιχα και η δική μας συζήτηση δεν έχει κλείσει ακόμα. Όπως και η Επιτροπή των Περιφερειών ε, φαντάζομαι ότι δεν έχει μία ενιαία και πάγια θέση στην υπόθεση αυτή, διαπιστώνω ότι και σε δικό μας επίπεδο υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις. Αυτά για τον ενδιάμεσο στόχο. Δεν θα πω περισσότερα προς το παρόν. Μετά, κάποιοι συναδελφοί ρώτησαν για τις μακροπεριφέρειες. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δεν θα συμφωνήσω με τον κύριο Σζίμων ότι δηλαδή η μακροπεριφέρεια αποτελεί την νομοποίηση δημοκρατική νομοποίηση μιας μετροπολιτικής περιφέρειας για συμμετοχή της σε ένα πρόγραμμα δεν νομίζω ότι είναι αυτό ο μόνο όρο. Ε, Στην τελευταία ανάλυση, αν κοιτάξουμε την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τη Γερμανία, ε, ολόκληρη είναι οργανωμένη, κατανεμημένη σε μητροπολιτικέ περιφέρειες. Θα ήταν λοιπόν η διάκριση αυτή με βάση τη μακροπεριφέρεια, μάλλον ει βάρος των υπόλοιπων ε, μικροπολιτικών περιφερειών. Θα πρέπει να υπάρχει κάποια πιο ρεαλιστική δυνατότητα διάκριση. Κύριο Ζημών επίσης μίλησε για συγχρηματοδότηση, εταιρικέ σχέσεις για την ανάπτυξη. Ναι, και τη συμμετοχή των ε, τοπικών αρχών. Είπατε. Ναι, δεν έχω καμιά αντίρρηση. Πολύ ευχαριστώ να το δούμε μέσα από τις τροπολογίες. Θα πιστώ από αυτά που θα μου προτείνετε. Για τον κύριο Αλφόνζη, κάποιες ιδέες που άκουσα με ανησυχούν διότι εάν λέτε εσείς αυτά που λέτε και εγώ αυτά που λέω, τότε μάλλον δεν έχουμε συνοηθεί. Και οι απειλές της κυρία Σρόιντερ επίσης με ανησυχούν ότι θα μου καταθέσει εκατοντάδες τροπολογιών. Κυρία Σρούντερ. μπορεί να ανήκω σε συντηρητικό κόμμα, μπορεί να μην είμαι και τόσο μοντέρνος πια ως προς τη στρατηγική της πολιτικής συνοχής. Συγχωρέστε με. Συμπαθάτε με. Το λέω σαν ε, αστείο βέβαια. Φυσικά, είχαμε στο παρελθόν μια στρατηγική στην ομάδα μου να απορρίπτουμε στη κάθε τροπολογία των πρασίνων. Δεν θα το κάνουμε τώρα, σα διαβεβαιώ, το είπα μόνο σαν αστείο. Ξέρω ότι έχετε πάντα καλές προτάσεις, ενδιαφέρουσε ιδέες. Και είμαι βεβαία, ε, βέβαια, ότι θα βρούμε καλές συμβαστικέ λύσει. Α σταματήσω λοιπόν εδώ και ευχαριστώ θερμά του συναδέλφου για τη μέχρι τώρα και για τη μελλοντική συνεργασία. Ευχαριστώ Μάρκους και βέβαια πάνω απ' όλα με ικανοποιείται ότι είχαμε καλή συζήτηση, ουσιαστική συζήτηση. Προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών θα ήθελα να σας υπενθυμίσω. Η πρόταση που έχει διατυπωθεί είναι 19η Απριλίου, Τρίτη, τη επόμενη εβδομάδα, 12 το μεσημέρι. 19 Απριλίου. Κλείνω το θέμα αυτό για να περάσουμε στο επόμενο της ημερησία μας διάταξης που είναι η ενσωμάτωση της διάσταση του φύλου στην πολιτική συνοχή. Και υπενθυμίζω όλους τους παρισταμένους, παρακαλώ, παρακαλώ, συνάδελφοι, βοηθοί, συνεργάτες, όποιος αποχωρεί, παρακαλώ, ησύχως. Παρακαλώ και τις συνομιλίες σας έξω από την αίθουσα παρακαλώ να τις ξεκινάτε. Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε εμεί. Έχουμε λοιπόν τη συμπερίληψη τη διάσταση του φίλου στην πολιτική συνοχή Ευρωπαϊκή Ένωση και παρακαλώ ε, ενημερώνω του αδέλφου που μένουν στην αίθουσα ότι έχει φτάσει η ώρα σχεδόν που θα συζητήσουμε το προσεχές νομοθετικό πλαίσιο για την πολιτική αυτή και άρα πρέπει να συζητήσουμε τώρα με τους εμπειρογνώμονες τις βέλτιστες πρακτικές για την πολιτική της συνοχής. Σας έχουμε διανύμει τα, τις σημειώσεις της ε, Elizabeth με το σημείο εστίασης πολιτικής για την ενσωμάτωση των φύλων, της διάστασης του φύλου καλύτερα, στην ε, πολιτική συνοχή και παρακαλώ τώρα τους εμπειρογνωμονές μας να μας παρουσιάσουν τις θέσεις τους. Έχουμε την Μπρίτ Μαρίζε Σέντεμπερκ Τόλστερσον, επικεφαλής του ε, σχεδίου WINET, συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής. Έχουμε την κυρία Εύα Ρουμίνσκα Ζήμνη, από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, πρώην επικεφαλής του προγράμματος του ΟΗΕ για το φύλλο και την ε, οικονομία από την Οικονομική Επιτροπή των ΗΠΑ για την Ευρώπη και την κυρία Αν Σάρλοτ Κάλερστη και Ευρωπαϊκή Κοινότητα για την Ευρωπαϊκή Εφαρμογή της διάθεσης του Φύλου. Καλό λοιπόν πρώτα την Μπριτ Μαρίζε. Σόντερμπερκ Τόστερσον παρακαλώ όλοι οι υπόλοιποι που συνομιλείτε μέσα στην αίθουσα ησυχία. Ε, Μπρίτ Μαρία, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και εσάς και την Επιτροπή σας βέβαια για την πρόσκληση. να σας παρουσιάσουμε το σχέδιό μας και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε η προοπτική των δύο φίλων να ενσωματωθεί σε μια μελλοντική πολιτική για την, για την συνοχή και τη στρατηγική του 2020. Είχαμε ήδη την ευκαιρία να συστήσουμε ε, προτάσεις περί την Βαλτική, για την περιοχή της Βαλτικής δηλαδή και την συμμετοχή των γυναικών σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ε, το έργο αυτό, Winnet 8, του Interreg 4C, Capitalization, ε, ξεκίνησε το 2008 και ολοκληρώνει το 2011. Έχουμε χώρες από τον βορρά, τον νότο, την Ανατολή και τη δύση της Ευρώπης και συντονισμό πόρων, συμμετοχή γυναικών από όλες τις χώρες, νέο εισερχόμενα μέλη. Έχουμε την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, όπως βλέπετε την Πολωνία, με δύο περιφέρειες, σε επίπεδο διορθωτικών ταμείων, Φινλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία και Σουηδία που αποτελεί και τον ε, επικεφαλής του έργου μια κοινότητα συγκεκριμένα στην κεντρική Σουηδία. Έχουμε και την Σκοτία. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με κέντρα, ε, όχι μάλλον έχουμε κάνει λάθος στην ε, Διαφάνεια λέει η ομιλήτρια. Όχι, όχι, καλά, τότε να συνεχίσω. Στόχοι μας λοιπόν, στόχοι του Winnet 8, είναι η ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας των γυναικών σε χώρους όπου επικρατούν οι άντρες, οι τομείς και αντιμετώπιση της διάκρισης των φύλων στην απασχόληση, η ανταλλαγή εμπειριών και πολιτικό, από πολιτείες και μεταφορά βέλθων πρακτικών ε, στην ομάδα του Winnet 8, η ενίσχυση των κέντρων στήριξης των γυναικών, ή γυναικείων πόρων όπως λέγονται στις διάφορες περιφέρειες ε, εταίρους. Στην επόμενη διαφάνεια. Αποστολή και λόγος ύπαρξης του Winnet 8 είναι η ενίσχυση του αριθμού των γυναικών που συμμετέχουν στον οικονομικό βίο σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η ανάπτυξη νέων μόνιμων θέσεων εργασία με την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των γυναικών και η ενίσχυση της ε, παραγωγικότητας, της αύξησης παραγωγικότητας ε, σε αγαθά και υπηρεσίες, η ενίσχυση της επιρροής που μπορούν να ασκήσουν οι γυναίκες στην αγορά εργασία, τα πιο, ισοδύναμη, πιο ισότιμη κατανομή ε, και δραστηριότητες σε περιφερειακό τοπικό επίπεδο με διαφορετικά προφίλ. Στην επόμενη διαφάνεια, εάν κοιτάξουμε την ποικιλία των πρωτοβουλειών που έχουν αναπτυχθεί, Βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορές σε επίπεδο είτε κράτους μέλους, είτε περιφέρειας, είτε κοινότητας, είτε και κράτους ακόμη. Δηλαδή μπορεί κανείς να αναπτύξει δραστηριότητα σε πανεπιστήμιο, σε σχολείο, να ενθαρρύνει την επιστημονική γνώση, μηχανολογική τεχνολογία, καινοτομία, ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση στο να κατευθυνούν οι γυναίκες προς τις μη παραδοσιακές επιλογές, ε, διευκόλυνση για ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, ε, κατάρτιση και υποστήριξη με μαθήματα, ιδιαίτερα σε γυναίκες διαφόρων μειονοτικών ομάδων και βέβαια προσφορά είτε ε, πραγματικών είτε εικονικών υπηρεσιών και ευκαιριών. Στην επόμενη διαφάνεια, οι λειτουργίες και η προσέγγιση είναι η πρόσδοση ικανότητας στις γυναίκες ε, απευθείας η δικτύωση σε διάφορα επίπεδα των κοινωνικών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και μέσα σε κράτη-μέλη σε επίπεδο εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό αλλά και ευρωπαϊκό όπως είπα. όπου κρίνουμε πολύ σημαντικό να υπάρχει ο συνδυασμός της ενσωμάτωσης του φύλου μέσα στις κύριες δράσεις μετά έχουμε ένα πρακτικό παράδειγμα από την Ελλάδα, στην επόμενη όπου είχαμε συνεργασία πάνω σε ένα μοντέλο για πολλά χρόνια για την ανάπτυξη ενός κέντρου γυναικείων πόρων με θέμα ιδιαίτερα την απασχόληση και ε, επιχειρηματική δραστηριότητα των γυναικών, την στήριξη γυναικών, ε, ενίσχυση των ε, δεξιοτήτων τους, επαγγελματικών δεξιοτήτων, δυνατότητα επανένταξη στην αγορά εργασίας, συνδυασμό αυτών των υπηρεσιών με άλλου δυναμικού ε, σχέδια, προγράμματα έργα στο τοπικό, εθνικό, περιφερειακό επίπεδο, συμμετοχή γυναικών 143 τον αριθμό που βρήκαν θέση στην εργασία, 63 που ίδρυσαν δική τους επιχείρηση, 7 που ίδρυσαν στην ε, αγροτική εταιρεία, επιχείρηση μάλλον με υποστήριξη και 21 που είχαν ε, υποστήριξη σε επιχειρηματικά, ε, με επιχειρησιακά σχέδια. Μετά έχουμε το παράδειγμα της Σουηδίας με το κέντρο γυναικείων πόρων Περιφερειακό Κέντρο Γυναικείων Πόρων που ξεκίνησε τις δραστηριότητες το 1995 αν και οι βέλτιστες πρακτικές ορίζεται ορίζουν ε, ότι υπάρχει κρατική χρηματοδότηση αυτών των κέντρων γυναικείων πόρων για τις ε, ειδικά σε εθνικό επίπεδο χρηματοδότηση αλλά και τοπικό ή εθνικό για την ανάπτυξη του δυναμικού για το 2002 και συγκεκριμένα η Σουηδική Υπηρεσία Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, δηλαδή κρατική επιχείρηση, κρατική εταιρεία ε, στηρίζει αυτό το πρόγραμμα. Σε αυτή την προγραμματική περίοδο λοιπόν 2010-2012 η κυβέρνηση της Σουηδίας ε, χορηγεί 3,3 εκατομμύρια ευρώ για κάθε χρόνο στη συγχρηματοδότηση και με το Ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακή Ανάπτυξης και με άλλα προγράμματα ευρωπαϊκά. Καθήκον αυτού του κέντρου γυναικείων πόρων είναι στην περιφερειακή ανάπτυξη για την ε, οικονομική ανάπτυξη, η επιχειρηματική δραστηριότητα και η καινοτομία, η είσοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας σε όσο δυνατόν ευρύτερο φάσμα θέσεων εργασίας στο να αντιμετωπιστεί αυτός ο διαχωρισμός των φύλων, προσβασιμότητα, υποδομές, μεταφορές, τηλεεργασία, δι ασυνοριακή και υπερσυνοριακή συνεργασία, επιχειρηματική δραστηριότητα, καιροτομία, περιφερειακή ανάπτυξη. Στο Winnet 8 λοιπόν έχουμε σε συστασή την πρόταση για μια πλήρη συζήτηση στρογγύλης σε ευρωπαϊκό επίπεδο πριν από τον προσδιορισμό 14 16 Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα των τελικών ε, συστάσεων και του προγράμματος δράσεως για την προσεχή προγραμματική επίπεδο στο πλαίσιο του προγράμμα, περιφερειακού προγράμματος ε, δράσης. Αλλά πάντως έχουμε να προτείνουμε μια πλατφόρμα δράσης μέσα από τη στρατηγική του 2020 να προβάλλουμε την διάσταση των φύλων, τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, την ε, κοινωνία της πληροφορίας, την καινοτομία, την ε, συμμετοχή στη γνώση, την συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σε κάθε επίπεδο στην Ευρώπη και στο διαπεριφερειακό πρόγραμμα δημιουργία συγκεκριμένων δικτών αποτελεσμάτων και μέτρων για την ισότητα των φύλων με ειδικού που θα μπορούσαν να προσφέρουν μέσω των γνώσεών τους των ειδικών συγκεκριμένε προτάσεις ε, για δράση και τελική πρόταση όταν τα κράτη-μέλη θεσπίζουν μια πλατφόρμα, είναι η θέσπιση μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας ε, για την ισότητα των φύλων. Η προαγωγή, όπως είπα, της αγοράς εργασίας επιχειρηματικότητας, ε, μια ουσιαστική αλλαγή δηλαδή, και βέβαια η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Αυτός είναι ο τελικός στόχος τελευταία ανάλυση. Ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Και έτσι κλείνω σημειώνοντας ότι ο αποκλεισμός των γυναικών από την αγορά εργασίας, η, η διακριτική αντιμετώπιση τους, ε, κοστίζει πολλά δισεκατομμύρια στην Ευρώπη. Η ενσωματωσία των φίλων η συμμετοχή των γυναικών σε κάθε τομέα της ε, επαγγελματική δραστηριότητας και τώρα στον επιχειρηματικό έχουν πράγματι τεράστια σημασία για την ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Κυρία Καζίμνα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Επιτροπή που οργάνωσε αυτήν την ε, ακρόαση και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα τη ε, ενσωμάτωσης διάσταση του φύλου για το μέλλον τη πολιτική συνοχή. Επομένω. είναι πολύ έγκαιρο το ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μοιραστώ κάποιε από τι εμπειρίε και τι συστάσει μου βάσει, από, βάσει της ε, προηγούμενης μου εμπειρίας σε διακυβερνητικό επίπεδο, διαπραγματεύσεις με Άλλε χώρε ε, και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό στην πολιτική συνοχή ε, σε σχέση με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου. Όταν βλέπουμε τα αποτελέσματα, το θέμα αυτό ε, επικεντρώνεται κυρίως στο κοινωνικό χάσμα, όπω για παράδειγμα τον αποκλεισμό, τον κοινωνικό, όμως ε, όλοι, όλοι οι στόχοι μας ε, δεν αφορούν καθόλου τη διάσταση του φύλου. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότερες γυναίκες είναι εντελώς αποκλεισμένες από τις ε, πρωτοβουλίες της, της, πολιτική, της κοινωνικής συνοχής που αφορούν για παράδειγμα την αύξηση, την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα Επομένως, ε, μένουν και εκτός χρηματοδότησης και θα επανέλθω σε αυτό. Αν ε, διαβάσει κανείς ε, την πέμπτη έκθεση για τη συνοχή και την εδαφική συνοχή, είναι σαφές ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο, κεφάλαιο η πρωτοβουλία και η ε, ανταγωνιστικότητα δεν έχουν καμία ε, γυναικεία διάσταση. Ακόμη και στον τομέα του ανθρώπινου κεφαλαίου δεν ε, έχει συμπεριληφθεί αυτή η διάσταση. Πράγματι υπάρχει αναγνώριση του, του, του ρόλου των γυναικών στην απασχόληση και στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά όταν αξιολογείται ο αντίκτυπος ε, σε σχέση με την ισότητα των ευκαιριών είναι σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, πολιτών δηλαδή, Κάτι το οποίο πάλι είναι περίεργο, γιατί έχει έναν αντίκτυπο στις οικονομικές επιδόσεις. Ε, δεν είναι μόνο ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, ο ρόλος των και γιατί συμβαίνει αυτό. Πρώτον, γιατί υπάρχει μία ιδέα ότι τα οικονομικά είναι μία ε, ε από άποψη φύλου ουδέτερη επιστήμη και πηγαίνει παλιά πίσω στον Άνταμ Σμιθ και στους άλλους μεγάλους ε, ε, ε οικονομολόγους πριν από 200 χρόνια οι γυναίκες ήταν ε, στην κουζίνα ε, και οι άντρες ε, ήταν στην παραγωγική, παραγωγική σφαίρα και είχαν πολύ σημαντικές θέσεις απασχόλησης. Οι οικονομολόγοι και οι μεγάλοι επιστήμονες δεν παρατηρούν το γεγονός ότι η διάσταση του φύλου είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό τμήμα της οικονομικής επιστήμης αυτής καθεαυτής. Γι' αυτό κάθε φορά που θέλουμε να το συμπεριλάβουμε στα οικονομικά ζητήματα ή στην πολιτική συνοχής ε, ε, οι περισσότεροι ρωτούν μα τι σχέση έχει τέλος πάντων το θέμα αυτό έχει να κάνει με την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Θεωρεί δηλαδή, θεωρούν δηλαδή και όντω. Αυτό τελικά καταλήγει να τοποθετείται σε, μια, σε περιθωριακά έγγραφα ε, γύρω από το βασικό θέμα που συζητείτε. Και να, είναι γεγονός ότι πρέπει να συζητήσουμε αυτό το θέμα, δημιουργεί επιπρόσθετα κονδύλια, επιπρόσθετο κόστος και δεδομένων των δημοσιονομικών περικοπών, αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Βάσει των δεδομένων του 2006, 7% του κοινωνικού ταμείου αποδόθηκε στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και αυτό συμπεριλαμβάνει τις δαπάνες για τη συμφιλίωση οικογενειακού ε, και, και επαγγελματικού βίου. Τι γίνεται σήμερα, αν δει κανείς ε, την οικονομική θέση των γυναικών, ε, ε, είναι το λιγότερα χρησιμοποιημένο δυναμικό ε, σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Ε, συνάδελφοί μου θα παρουσιάσουν την εμπειρία των βαλτικών χωρών. Σε επίπεδο απασχόλησης υπάρχει το σημαντικότερο πρόβλημα και αυτό αναφέρεται. Αυτό που δεν αναφέρεται είναι ο ρόλος και συνεισφορά των γυναικών από ποιοτική απόψεως. Τι προσφέρουν δηλαδή από απόψη ω ποικιλία ταλέντων, ε, ειδών διαχείρισης, προτεραιοτήτων, παραγωγής, ε, ε, μεθόδους ανάπτυξη και παραγωγής και επίσης την αντίληψή τους για το εισόδημα. Ε, οι γυναίκες δηλαδή ε, ως χρήστες ή ως ε, υπεύθυνοι λήψη αποφάσεων θα βοηθούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταγωνίζεται καλύτερα και σε τοπικά και σε περιφερειακά και σε, και σε τοπικό και σε περιφερειακό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι όταν βλέπει κανείς κάποια από τα ανέκδοτα που αναφέρονται. Αν οι Lehman Brothers ήταν ε, Lehman Sisters και Brothers, ενδεχομένως ε, η ανάληψη και η διαχείριση του κινδύνου όλης ε, ε της εταιρεία θα ήταν εντελώς διαφορετική. Αυτό είναι ένα ανέκδοτο που θέλει κάτι να πει. Ένα ακόμη παράδειγμα, όταν οι γυναίκες έχουν την πλειοψηφία του μεριδίου στην εκπαίδευση, για παράδειγμα, σε πολλές χώρες μέχρι και 60%, ε, μόνο 20-30% είναι ηγετικές θέσεις. Ε, ε, άρα αυτό που πιστεύω είναι ότι μια βασική πρόκληση για το θέμα αυτό είναι η ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των γυναικών ε, με, στην οικονομική, στον οικονομικό βίο μετά το 2013 και θα ήθελα τρεις καλές πρακτικές να ε, σας αναφέρω που κατά τη γνώμη μου θα μπορούσαν ε, να εγκριθούν σε επίπεδο πολιτικής συνοχής και να υιοθετηθούν. Πρώτον, καινοτομία οργάνωσης ε, θερινών σχολείων για την μακροοικονομία ε, μια ιδέα που, υπήρξε από το, που υπήρχε από το 1994 για την προαγωγή της συμμετοχής της γυναίκας ε, στην ε, λήψη αποφάσεων, στη χάραξη πολιτικών και στους μη κυβερνητικούς και στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Κάποια από τα προγράμματα έχουν ήδη εφαρμοστεί το 2011 και 2012 έχουμε ένα μακροπεριφερειακό πρόγραμμα το οποίο βασίζεται σε δύο ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Πολωνία, ε, στην Οικονομική Σχολή, αλλά και στο ε, ε, οικονομικό, στην οικονομική σχολή της Κωνσταντινούπολης και το λέω αυτό στο πλαίσιο της μακροπεριφερειακής πολιτικής ε, σε συνεργασία με τις ε, κοντινές, με τις γειτονικές χώρες του Καυκάσου με σκοπό τη συζήτηση του κατά πόσο οι γυναίκες μπορούν να βοηθήσουν ε, στην χάραξη της οικονομικής πολιτικής. Αυτό εμείς στην Πολωνία το έχουμε ήδη δρομολογήσει και σε περιφερειακό και σε παγκόσμιο επίπεδο σε συνεργασία με τον WIPO, τον Οργανισμό για την Πνευματική Διοκτησία στη Γενέβη. Ο σημαντικός ρόλος διαδραματίζεται από τα κέντρα καινοτομίας που συμμετέχουν ενεργά σε αυτήν την πλατφόρμα και ένα από τα ζητήματα που συζητήσαμε συζητήθηκαν ε, ήταν ποιο είναι ο όρο καινοτομία γιατί έχουν διαφορετική άποψη για την καινοτομία οι γυναίκε. Η καινοτομία χρηματοδοτείται από, το Ευρωπαϊκό, ε, από τα Ευρωπαϊκά Διαδροτικά Ταμεία ως ε, πρόγραμμα καινοτομίας. Και θα ήθελα εν τέλει να πω ορισμένα πράγματα για την επιτυχία των γυναικών σε περιφερειακό επίπεδο, μία προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή ε, εκλέγονται γυναίκες ε, σε ηγετικές θέσεις και για κοινωνικά θέματα αλλά και για περιφερειακά πολιτικά ζητήματα. Τώρα, ποια είναι τα συμπεράσματα για την αναθεώρηση της πολιτικής συνοχής. Ε, νομίζω ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να ξοδεύουμε τον γυναικείο δυναμικό, ούτε μπορούμε να είμαστε απλώς ουδέτεροι, να θεωρούμε τις οικονομικές πολιτικές ουδέτερες από απόψεις, από φύλου. Υπάρχει ο κίνδυνος όταν μιλάμε για μια θεματική συγκέντρωση που αναφέρεται και στην έκθεση, μπορεί να χάσουμε τις πτυχές της διάστασης του φύλου που από κοινωνικής απόψεως θα είχε πολύ μεγάλο κόστος ε, στο πολιτικό μας πρόγραμμα. Και το τρίτο μου συμπέρασμα είναι συνεπώς ότι η αναθεώρηση ε, του δημοσιονομικού πλαισίου της πολιτικής συνοχής μετά το 2013 θα έπρεπε να χρησιμεύσει ε, και για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου ε, και την κάλυψη των κενών που υπάρχουν ε, στην πολιτική αυτή. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπόδειγμα στα ζητήματα αυτά για τις ίσες ευκαιρίες σε παγκόσμιο επίπεδο και πρέπει να πρωτοστατήσει τώρα για την αναγνώριση του οικονομικού, δυναμικού των γυναικών. Και αυτό σημαίνει τουλάχιστον τρία πράγματα και θα ολοκληρώσω με αυτά. Πρώτον, αλλάξουμε τον τρόπο σκέψη μας ε, που, μας δίνουν, ε, που θα μας δώσουν τη δυνατότητα την ισότητα των ευκαιριών να τα συνδέσουμε με την οικονομία. Δεύτερον, εφαρμογή ε, πολιτικών επόμενη γενεάς, όπω για παράδειγμα διαπραγματεύσεις και τρίτον η μεγαλύτερη συμβολή των γυναικών ε, ε, στη διαδικασία εφαρμογή σε επίπεδο λήψη αποφάσεων. Διαφορετικά δεν έχει κανένα νόημα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή Thank Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ρουμίνη Καζίμνη. Και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην Αν Σαρλότ Κάλεστιγκ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Εγώ εδώ εκπροσωπώ σήμερα τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν σε ένα δίκτυο εκμάθησης ε, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, γιατί ε, εγώ εργάζομαι ε, σε αυτό ως εμπειρογνώμων. Άκουσα πολλά από την προλαλή για τις προοπτικές, για τις μελλοντικές πολιτικές και θα εξακολουθήσω κι εγώ να συζητώ το θέμα αυτό. Θα σας πω δύο πιθανά μελλοντικά σενάρια, ε, κατά τη γνώμη μου. Επόμενη διαφάνεια. Θα μιλήσω και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, το Ευρωπαϊκό ε, Κοινωνικό Ταμείο, αλλά και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη. Η περίπτωση λοιπόν της εφιούς ανάπτυξης και της καινοτομίας δείχνει ακριβώς τη συμπληρωματική φύση των δύο ε, ταμείων όταν μιλάμε για ζητήματα ε, ίσων ευκαιριών. Ε, έχει σχέση με το πώς ε, θεωρείται, πώς εκλαμβάνεται αυτή ε, η έννοια, γιατί ε, η συμμετοχή των γυναικών θα δώσει τη δυνατότητα μεγαλύτερης οικονομικής ανάπτυξης, περισσότερων πληροφοριών ε, και μιας κοινωνίας πιο ίσης σε τομείς όπως για παράδειγμα θαλάσσιες μεταφορές, οπτικές σύνες, όπως δείχνουν τα νορβηγικά και σουηδικά παραδείγματα, αν θέλετε μπορείτε να πάρετε και ένα αντίγραφο αυτών των φυλαδίων από μένα στο τέλος της συνεδρίασης. Ε, θα ήθελα επίσης να πω ότι το, η ενσωμάτωση των φύλων δεν είναι μόνο το σωστό, αλλά είναι και το ευφυές ε, πράγμα να γίνει. Όσον αφορά τώρα την εκμάθηση και την αλλαγή, γνωρίζουμε ότι ανεξαρτήτως πολιτικής Χρειαζόμαστε και εκπαίδευση και αφοσίωση. Χρειαζόμαστε υποστήριξη και καθοδήγηση για να είμαστε αποτελεσματικοί. Χρειαζόμαστε πόρους, γνώσεις, καθοδήγηση και παρακολούθηση. Επόμενη διαφάνεια. Ε, σύμφωνα με τις εμπειρίες μας λοιπόν ε, χρειαζόμαστε ε, τους στόχους που μερικές φορές χάνονται στη μετάφραση ε, από, τον, ε, από τον ορισμό τους μέχρι την εφαρμογή τους στα κράτη-μέλη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό ε, γιατί είναι εγκάρσια ε, η σημασία της ενσωμάτωσης διάστασης του φύλου. Αυτό που θα γίνει το 2000, ε, μετά το 2013 είναι αυτό που πρέπει να συμπεριλάβουμε και στις, στα εθνικά προγράμματα αναθεώρησης. Τι έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας, ποια στοιχεία έχουμε στη διάθεσή σας. Ε, τα διαρθρωτικά ταμεία και ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ήταν πάρα πολύ δραστήρια όσον αφορά το θέμα της ενσωμάτωσης διάστασης του φύλου. Γι' αυτό πρέπει να τονιστεί. Όμως, ε, βάσει πολλών αξιολογήσεων που έγιναν στην πλειονότητά τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και από άλλες ε, έρευνες, είναι σαφές ότι έχει γίνει πολλή δουλειά στα κρατημέλη, αλλά δεν υπάρχει συνοχή στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται ε, η ενσωμάτωση τη διάσταση του φύλου. Υπάρχει ένα χάσμα εφαρμογής, λοιπόν, και τον τρόπο με τον οποίο... Ε, εφαρμόζεται σε πολλές χώρες, ε, αναγνωρίζεται στη θεωρία, αλλά δεν εφαρμόζεται στην πράξη, σε τομείς όπως για παράδειγμα οι πολιτικές καινοτομία. Η σχέση πολιτικής και πόρων ε, δεν υπάρχει δεν υπάρχει βιωσιμότητα και επομένως σε μερικές περιπτώσεις δεν υπάρχουν μόνιμες δομές ε, για να εφαρμοστεί ε, μια σχετική προσπάθεια. Πολλά κράτη-μέλη έχουν εφαρμόσει μια πολιτική που ε, μόνο στα τελικά στάδια ενός προγράμματος η προτεραιότητα που τίθεται στην ενσωμάτωση διάσταση του φύλου από την Ευρωπαϊκή, την Επιτροπή είναι ένα βασικό παράγοντα που καθορίζει το πώ θα εφαρμοστούν οι πολιτικές αυτέ από τα κράτη-μέλη. Σε ένα πιο ομαδοποιημένο επίπεδο είναι επίση σαφέ ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ισότητα ε, ε, των Φύλων δεν έχει προπολογισμό και εξαρτάται για την εφαρμογή τη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Δεν υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο προπολογισμό για την ισότητα των φύλων. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ε, δεν έχει ε, συγκεκριμένη καθοδήγηση για την εφαρμογή των πολιτικών αυτών και επαφίεται στα κράτη-μέλη να διαλέξουν κάποιους από τους στόχους ε, ή κανέναν από αυτούς. Περνάμε λοιπόν τώρα στο τελευταίο θέμα που είναι και το βασικό θέμα για το μέλλον. Εσμελωτικές εξελίξεις. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο. Δύο σενάρια είναι πιθανά. Επόμενη διαφάνεια. Πρώτο σενάριο. Ε, το να είναι το θέμα αυτό ένα στρατηγικό τμήμα της πολιτικής συνοχής και ανάπτυξης Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ συγκεκριμένη στόχη και μάλιστα υπάρχει και προπολογισμό. Ε, είναι ένα ορατό τμήμα όλων των στόχων ε, πολιτικής. Η εφαρμογή ε, τυχαίνει καθοδήγησης και υποστήριξης και το αποτέλεσμα είναι μια πιο αποτελεσματική προσέγγιση πολιτικής και εντάσσεται σε έναν ευρύτερο ολοκληρωμένο στόχο. Η άλλη επιλογή είναι να μην υπάρχει καμία ρύθμιση, οι πολιτικές να είναι κατακαιρματισμένες, να περιλαμβάνουν μόνο μερικά στοιχεία των, ε, στόχων, κάτι το οποίο μπορεί να είναι αντιπαραγωγικό. Υπάρχουν πολλές χαμένες ευκαιρίες ε, για ε, ε, καινοτομία και οικονομική ανάπτυξη μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, να εξασφαλίσουμε ότι ο προπολογισμό θα υποστηρίξει εφαρμογή των στρατηγικών ενσωμάτων διάσταση του φύλου με απλά βήματα. Το υπόλοιπο της παρουσίασής μου θα πρέπει να το διαβάσετε όλοι, μόνοι σας. Και επίσης αν θέλετε μπορείτε να έρθετε και στην ε, ε, σχετική διάσκεψη που θα λάβει η χώρα στις Βρυξέλλες στις 26 Μαΐου. Αν ενδιαφέρεστε και θέλετε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ να μου δώσετε την κάρτα σας, το email σας ή μπορείτε να πάτε στο www.gendercoxeup.eu. Εκεί θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Και η τελευταία διαφάνεια Αυτά είναι που θα πρέπει να διαβάσετε μόνοι σας, οι διαφάνειε που περνούν. Ευχαριστώ πολύ για την ε, προσοχή σας. Και αυτό είναι ο τρόπος για να υποβάλλετε συμμετοχή στην ε, ε, διάσκεψη. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μίκαελ Λανταμπάζο, επικεφαλής του Τμήματος Θεματικό Συντονισμό και Ενοτομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μου ζητήθηκε να μελετήσω και να απαντήσω στις ε, ε, παρουσιάσεις που έκαναν οι εξαιρετές συνάδελφοι. Αυτό και θα πράξω. Πρώτη μου αντίδραση λοιπόν από τα όσα ακούσα είναι ότι όχι μόνο είναι θεμελιώδες δικαίωμα, θεμελιώδες αξία μάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προτεραιότητα ως στόχος οριζόντιος για, το, για τα ερωτικά ταμεία, όπως ορίστηκε στο άρθρο 16 του κανονισμού. Το ερώτημα όμως είναι το, η ενσωμάτωση της του φύλου έχει σχέση με την περιφερειακή ή με μια προσέγγιση εδαφική, χωρική. Και εμείς, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα ερωτικά ταμεία, κάνουμε αυτό που πρέπει. Η απάντησή μας στα δύο αυτά ερωτήματα είναι σαφώς ναι. Και θα ήθελα από τα όσα άκουσα από την Πρίτη Μαρία και τη Σαρλότ ως προς την περιφερειακή προσέγγιση να επισημάνω ότι το gender mainstreaming δεν είναι ουδέτερο ως προς το χώρο. Υπάρχει η περιφερειακή διάσταση δηλαδή στο gender mainstreaming και θα ήθελα να φερθώ στην πιο πρόσφατη μελέτη που συστήσαμε και με τα κράτη-μέλη για την ε, περιφερειακή διάσταση του gender mainstreaming που αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι οι διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών επιχειρηματιών στην επιχειρηματική δραστηριότητα ε, είναι πολύ, διαφορετική, πολύ μεγάλες ανάλογα με την περιφέρεια. Δηλαδή οι προηγουμένες περιφέρειες παρουσιάζουν διαφορές ως προς την επιχειρηματική δραστηριότητα ανδρών και γυναικών πολύ μικρότερες και μάλιστα στηριζόμενες σε δύο κυρίως ε, κρίσιμες μεταβλητέ. Το χρόνο που μπορεί να αφιερώσει η γυναίκα στην οικογένειά της και τον αριθμό του προσωπικού που μπορεί να προσλάβει, που είναι υψηλότερο στην περίπτωση των γυναικών μελών του προσωπικού. Για τις λοιπές μεταβλητές ε, βλέπουμε κάποια σχέση της διαφοράς μεταξύ ανδρών και γυναικών μόνο στις λιγότερο προηγμένες περιφέρειες. Και εδώ δεν έχει νόημα να κάνουμε κάποιες προσπάθειες. Τώρα θα ήθελα να πω για τα ε, κέντρα γυναικείων πόρων που ανέφερε η Μπριθ ότι πρέπει να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση στο πεδίο αυτό και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει η περιφερειακή διάσταση, η χωρική διάσταση στην ε, διαδικασία ενσωμάτωση του, του, των των φύλων να έχει σημασία. Και έτσι οι συνάδελφοι μελετούν στην υπηρεσία μας, ιδιαίτερα τις περιοχές της υπαίθρου, αν θέλουμε να διαφυλάξουμε την παρουσία και την οικονομική δραστηριότητα της γυναίκας στην υπαίθρο, πρέπει να προαγάγουμε τη δημιουργία της θέσης εργασίας εκείνης που θα κρατήσουν τις γυναίκες στην υπαίθρο. Και αυτό είναι σημαντικό καθήκον, πιστεύω, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το δεύτερο πράγμα στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι ο συσχετισμός μεταξύ του, της ενσωμάτωσης διάστασης του φύλου και της στρατηγικής 2020, την οικονομική διάσταση δηλαδή, της ενσωμάτωσης του, της διάστασης των φύλων. Θα λέγαμε ότι εν τέλει ο στόχος του 2020 είναι στόχος που σημαίνει ότι για να επιτευχθεί πρέπει να αυξηθεί από το 62-63% που έχουμε τώρα σε υψηλότερα ποσοστά η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία. Γιατί λοιπόν είναι ζήτημα φύλου η στρατηγική του 2020, διότι αν δούμε τι στατιστικές μας και τις πιο πρόσφατες από το Eurostat, διαπιστώνουμε ότι η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία είναι αντιστρόφως ανάλογη με τον αριθμό των παιδιών που κάνουν οι γυναίκες και αντιστρόφως ανάλογη με την κατάσταση των ανδρών. Άρα, εάν θέλουμε να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των γυναικών στον αγορά, στην αγορά εργασίας, θα πρέπει κάπως να βρούμε τη λύση για τη συμφιλίωση επαγγελματικού και οικογενειακού βίου. Και επανέρχομαι στο επιχείρημα στην αρχή της παρέμβασής μου. Άρα, η ε, υποδομές για υποδοχή παιδιών δεν είναι μια μεμονωμένη, μια αποκομμένη από την πραγματικότητα διάσταση ή κριτήριο. Έχει σημασία αν θέλουμε να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας για να φτάσουμε στους στόχους του 2020. Τώρα χρηματοδοτούμε μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, τέτοιου είδους ε, υποδομές υποδοχής παιδιών, παιδικούς κτλ. με πάνω από 500 500 εκατομμύρια. Και στις διαπραγματεύσεις, παλαιότερες διαπραγματεύσεις των προγραμμάτων μας, με πολλές από τις χώρες, Ισπανία, αν προκειμένου, ε, η παρουσία τέτοιων υποδομών υποδοχής παιδιών θεωρούνταν ως ε, επένδυση στοχευμένα που επιδίωκε την υλοποίηση των στόχων της Λισαβόνας. Αυτό κάναμε σκημένα βέβαια, δεν ήταν τυχαίο. Γιατί είχαμε αντιληφθεί σε επιτροπή ότι αν δεν μπορέσουμε να συγκεράσουμε τον οικογενειακό βίο με τις προοπτικές για πρόοδο επαγγελματική ανέλυξη των γυναικών, δεν θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει, να υλοποιήσει τους στόχους του το ευρωπαϊκό στρατηγικό πλαίσιο το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο της Ισπανίας. Παρουσία λοιπόν των γυναικών στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Και δεν μπορούμε από τις στατιστικέ που έχουμε σήμερα δυστυχώς να ε, διακρίνουμε πώς ε, οι 500.000 ευρώ που έχουμε διαθέσει ή ποιο μερίδιο αυτών που διαθέτουμε για την εκκίνηση μιας επαγγελματικής δραστηριότητας πάνε σε γυναίκες. Ξέρουμε όμως ότι φέρνουν συνολικά αποτελέσματα και γι' αυτό και το κύριο μας ε, βραβείο το δώσαμε πέρσι σε μια σουηδική ε, πρωτοβουλία που προήγαγε την ανάπτυξη επιχειρήσεων από γυναικές στην Σουηδία και τη στήριζε με μικροπιστώσεις. Κυρίως μόλις απευθυνόταν σε γυναίκες από διαφορετικές εθνοτικές προελεύσεις, ε, από περιθωριοποιημένες ομάδες κτλ. Ήταν ένα κέντρο ανθρωπίνων πόρων, γυναικείων τι κάνουμε λοιπόν και τι μπορεί να γίνει επιπλέον. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω καταρχάς ότι η Επιτροπή στην υπόθεση αυτή βρίσκεται σε ε, διαδικασία μικτής διαχείρισης, shared management, δηλαδή θα πρέπει για να τα καταφέρουμε αυτά στα, ε, από τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουμε τα εξής τρία πράγματα την αναγνώριση σημασίας της ανάγκης να επενδύσουμε ε, στην προαγωγή της ενσωμάτωσης των φύλων, της ισότητας των φύλων. Δεύτερον, θα πρέπει να γίνουν κάποιε επιλογέ δύσκολε μερικέ φορέ και ω προ τα χρήματα που θα διαθέσουμε, το, τη στόχευση των χρημάτων, τι προτεραιότητες. Και τρίτον, σημείο στήριξη πάλι στην Επιτροπή και λόγω αυτού του shared management που έχουμε, είναι να βρούμε ιδέες για το πώς θα υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Το πώς λοιπόν σημαίνει ευαισθητοποίηση, διάδοση βέλτιστων πρακτικών, γιατί σε αυτά επικεντρωνόμαστε, και επιτρέψτε μου πολύ γρήγορα να αναφέρω έναν ε, σύντομο κατάλογο ιδεών που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν για να σας δείξω τι προσπαθούμε να επιτύχουμε. Έχουμε επί παραδείγματι μια ομάδα το επίπεδου για την ενσωμάτωση της έσωσης του φύλου που ήδη λειτουργεί εδώ και μερικά χρόνια και όπου ζητάμε από τα κράτη-μέλη να καθίσουν, να παρουσιάσουν το καθένα τις πρακτικές του, να εμπνευστούν το ένα από τα άλλα και βέβαια πόσα μπορεί να προσφέρει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από πλευρά τη για, τους, ε, για τις επενδύσεις στον τομέα αυτών. γιατί μπορούμε να δεχτούμε στην πράξη και θα ήθελα να υπογραμμίσω στο άρθρο 16 ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε ίσες ε, ευκαιρίες με το σχεδιασμό ενός προγράμματος, με την ε, επιλογή των ορθών έργων μέσα σε ένα πρόγραμμα ή μέχρι και την τελευταία, ε, το τελευταίο στάδιο, δηλαδή την αξιολόγηση ενός έργου. Εκεί είναι η δυσκολία. Αυτή λοιπόν ε, η ομάδα ανώτατου επίπεδου που δραστηριοποιείται σε τέτοιο επίπεδο προσπαθεί να λειτουργήσει και ως πλατφόρμα για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Και έτσι προσπαθήσαμε και τελευταία φορά που συναντηθήκαμε και με τις συναδέλφους που ήρθαν να σας μιλήσουν σήμερα εδώ να διαδώσουμε στο βαθμό του δυνατού τι πληροφορίε, τι γνώσει που μπορούμε εμεί να αποκομίσουμε και από τη δική μα εμπειρία. Παραδείγμα, τελευταία χρόνια ε, έχουμε ε, επικοινωνήσει με τα κρατημέλη και του έχουμε μεταδώσει τις εμπειρίες που έχουμε από την περίοδο μέχρι το 2006. Αντίστοιχα και οι άλλες υπηρεσίες. Αντίστοιχα και η εξάντια αξιολόγηση του άρθρου 16 που πάλι μοιραστήκαμε με τα κρατημέλη. Σε αυτές τις συνεδριάσεις επίσης παρουσιάζουμε ε, παραδείγματα των πρακτικών και η Επιτροπή είναι παρούσα με στόχο την πρόταση της εναρμόνισης των βέλτιστων πρακτικών που υπενθυμίζουμε. Θέλω να επισημάνω, επισημάνω επίση ότι θεωρούμε ότι είναι πολύ καλή η δουλειά αυτή. Η Ισπανία, η Πολωνία, η Φιλανδία και τώρα και η Πορτογαλία έχουν ε, ξεκινήσει τις αξιολογήσεις, εθνικές αξιολογήσεις για την ενσωμάτωση των φίλων. Άρα προσπαθούμε να δώσουμε μια ευκαιρία για συμμετοχή των ανθρώπων, ε, των πιο έμπειρων σε αυτή τη διαδικασία. Να δαχθούμε, να μεταδώσουμε τις γνώσεις αυτές στα κρατημέλη, τα οποία βλέπουν στη γενική, στο γενικό κανονισμό πρόσκληση μέσω του άρθρου 66 παράγραφο σημείο 2 να ενσωματώσετε τις δικές και τους δείκτες τους όπου είναι δυνατόν. Όπου είναι δυνατόν, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, έτσι λέει το κείμενο, τις στατιστικές σε κατανομή φύλου. Αυτό είναι μια απέτηση. Δυστυχώς όμως αυτό δεν ε, γίνεται σε όλες τις επενδύσεις και σε όλα τα μέτρα σε όλα τα σχέδια καλύτερα. Όμως κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διαδώσουμε αυτή τη βέλτιστη πρακτική, για να ενσωματώσουμε τα εργαλεία μάθησης, ε, για να δώσουμε το λόγο σε αυτούς, σε αυτές τους ενδιαφέροντες ομιλητές ομιλήτριες, για να δώσουμε και τεχνική στήριξη στα κράτη-μέλη, ώστε να δημιουργήσουν τη δική τους εσωτερική πλατφόρμα. Γιατί κάθε χώρα έχει δική της δικές ιδιαιτερότητες, διαφορετική κατάσταση. Και με τεχνική μας στηρίξη ορισμένες φορές τα κράτη-μέλη μπόρεσαν να ιδρύσουν μια εθνική πλατφόρμα με ε, επαφή, συνεδρίαση για την αντιμετώπιση του ζητήματος της ενσωμάτωση των δύο φύλων, με τακτικές επικοινωνίες και με τις εθνικές κυβερνήσεις, με τα ιστοτοτών των Γυναικών τα κέντρα γυναικείων πόρων που εξετάζουν πώς προχωρεί η κατάσταση, πώς υλοποιείται αυτό το σύνολο καλών προθέσεων που έχουμε καταγράψει στους κανονισμούς. Και για να τελειώσω τώρα, θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να επισημάνω ότι από τα τρία πράγματα τα οποία καταγράφονται εδώ για την αλλαγή στις νοοτροπίες, ενσωμάτωσης της θέσης του φύλου στην υλοποίηση και την ενσωμάτωση των γυναικών σε δικασίες λήψη αποφάσεων, έχουμε νομίζω να λάβει δραστηριότητα, κάνουμε ό,τι μπορούμε και τι φαίνεται ότι δεν αρκεί, στους δύο πρώτους στόχους, με τα εργαλεία, με τα μέσα που σας ανέφερα, και Πολύ σημαντικό επίσης βρίσκω όταν γίνεται λόγος για θεματική θεατρολογική συγκέντρωση, δεν βλέπω αντίφαση μεταξύ θεματολογικής προσέγγισης και ενσωμάτωσης θέσης του φύλου, mainstreaming δηλαδή. Θα έπρεπε να υπάρχει αυτό ούτως ή άλλως. Το mainstreaming θα έπρεπε να είναι παντού, δεν θα πρέπει να είναι ένα χωριστό θέμα, δεν είναι θέμα το mainstreaming. Φερρυπίν τελευταία συνεδρίαση της ομάδας ψηλού επίπεδου για την σωματοζήτηση των φύλων δόθηκε ένα εξαίρετο παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο ε, σωματώθηκε η διάσταση του φύλου στην κατασκευή υπόγειου συνδρόδρομου. μετρό. Αντίστοιχα, παραδείγματα έχουμε δει από εκπαιδευτικέ ή ε, κοινωνικέ υποδομέ. Άρα θεωρούμε ότι το mainstreaming είναι, το gender mainstreaming είναι οριζόντιο θέμα, δεν είναι χωριστό θέμα, πρέπει να υφίσταται παντού, πρέπει να το βλέπουμε παντού, είναι θέμα αποτελεσματικότητας κιόλας. Και πιστεύουμε ότι υπάρχουν στην πράξη τρόποι για να επιτευχθεί αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά και ελπίζω να έχω δώσει απαντήσεις μου στις, ε, στους προβληματισμούς σας. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Λανταβάζο, θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Η κυρία Ρίζεπεθ Σρέτερ πρώτη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και πάνω απ' όλα ευχαριστώ για τη συμπερίληψη του σημείου αυτού στην ομιλία ένταξη σε μια χρονική στιγμή που ίσω να μην έχει τόσο μεγάλη προβολή. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχει εκεί πρόβλημα, στο ότι δεν θεωρείται τόσο σημαντικό το θέμα αυτό. Είναι σαφέ από τα όσα υπόθηκαν στι παρουσιάσει ότι πολλά λέγονται, λίγα γίνονται. Καθίσατε επίση σαφέ ότι από ό,τι φαίνεται αυτή η ρήτρα για την οποία είχαμε αγωνιστεί πολύ σκληρά για τις αρχικές προτάσεις, μην θυμίζω δεν υπήρχε και αγωνιστήκαμε σκληρά για να μπει το gender mainstreaming επιπλέον μέσα στις διατάξεις. Την ίστατη στιγμή των διαπραγματεύσεων, σκληρή λοιπόν διαπραγμάτευση όπως είπα, τη συμπεριέλαβε στο κείμενο. Αλλά όπως φαίνεται δεν αρκεί, δεν υπάρχει αρκετή στράτευση στην υπόθεση αυτή. Πάντω χαίρομαι διότι με την ομάδα αυτή επίπεδου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταφέρει να βρει ένα εργαλείο ένα μέσον ε, που κάνει καλή δουλειά, που επιτρέπει τουλάχιστον την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, γιατί νομίζω ότι είναι καλό να βλέπουμε αυτά τα καλά παραδείγματα. Τα έργα επίσης, τα σχέδια τα οποία υποστηρίζονται είναι πιλωτικά και δείχνουν τι δυνατότητες υπάρχουν και πόσο σημαντικό είναι αυτό που γίνεται. Τώρα πια βέβαια πρέπει να αναλογιστούμε τι κάνουμε στο μέλλον. Και ποια είναι τα στοιχεία κλειδιά, όπως αποδεικνύεται και από τις παρεμβάσεις. Από τις ομάδες εργασίας λοιπόν, τις οποίες έχω εγώ παρακολουθήσει και από όλα τα έγγραφα που έχω διαβάσει, βλέπω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται, αλλά πρέπει να ληφθεί πιο σοβαρά υπόψη. Δεν υπάρχει αρκετή σοβαρότητα στην αντιμετώπιση του. Αφενό από την Επιτροπή, γιατί βλέπω ότι η Επιτροπή δεν κάνει προγράμματα συγκεκριμένα που να πει να πρέπει να κάνουμε κάτι να βελτιώσουμε την υλοποίηση ή, και αν τα κάνει δεν γίνεται τίποτα ουσιαστικά. Ένα γερμανικό πρόγραμμα που έχω υπόψη μου εγώ. Ακριβώ αυτό έγινε. Ωραία λόγια και δεν έγινε τίποτα. Ίσως να μην ήταν τόσο λαϊκή η γλώσσα όπως σας τα περιέγραψα εγώ, ήταν κάπως πιο κόσμια ε, υπηρεσιακή ορολογία, αλλά το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Σε άλλε χώρε όμω βλέπουμε τα πράγματα να προχωρούν διαφορετικά. Και η Επιτροπή ανέφερε την Ισπανία ω παράδειγμα. Υπήρξε μια task force για την ε, ενσωμάτωση σα των φύλων στις τοπικές αρχές και μάλιστα αυτή φάνηκε χρήσιμη όχι μόνο για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και για τα εθνικά προγράμματα. Αξιοποιήθηκε δηλαδή και για τα εθνικά προγράμματα. Πράγμα το οποίο αποδεικνύει την προσθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει κυρίες και κύριοι συναδελφοί ένα ε, κείμενο επιστολής το οποίο είχα διατυπώσει ως συμπεράσματα αυτής της δουλειάς και της παρακολούθησης αυτών που γίνονται, που είχα αναλάβει εγώ και που δείχνει πιστεύω ότι όταν αυτά τα μέτρα, όταν αυτές οι προτάσεις ε, υλοποιούνται με σοβαρότητα, μπορούν να φέρουν σαστικά αποτελέσματα. Και υποστηρίζω βέβαια κάθε τέτοια σοβαρή προσπάθεια. Και βέβαια είναι σαφές ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει την ε, πρωτοβουλία και να πει ότι δεν δέχεται καμία στατιστική αν δεν έχει διάκριση μεταξύ των φύλων, εάν δεν έχει ταξινόμηση καλύτερα μεταξύ των φύλων, ότι δεν θεωρεί δηλαδή ικανοποιητικέ στατιστικέ αυτέ. Εάν αυτή τη διάσταση τη ε, ενσωμάτωση των φύλων δεν την λάβει στα σοβαρά υπόψη η Επιτροπή, δεν πρόκειται κανεί να το κάνει. Άρα, εδώ βλέπω μια συγκεκριμένη απέτηση για το mainstreaming στην πράξη και επίσης θα ήθελα να δούμε πόση χρησιμότητα αποδεικνύεται πως έχει και σε ποιο βαθμό τα κράτη-μέλη αφήνουν το θέμα αυτό και το θεωρούν μόνο αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ταμείου και λένε ότι δεν έχει το καμιά σχέση με αυτά. Νομίζω ότι το παράδειγμα της Πολωνίας είναι χρήσιμο γιατί δείχνει ότι μπορούν οι γυναίκες επιχειρηματίες να κερδίσουν ε, τη θέση τους στον επιχειρηματικό κόσμο. Έχω αντίστοιχο ένα παράδειγμα από τη Βρέμη και νομίζω ότι μπορώ να σας στείλω τον ε, σύνδεσμο στο διαδίκτυο. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε δηλαδή από εκεί το τι γίνεται στην πράξη και πώς μπορούν οι γυναίκες να συμμετάσχουν στην αγορά εργασίας. Και μάλιστα πρακτικά δόθηκε μια πρημοδότηση σε επιχειρήσεις, στη Βρέμη αυτό, ε, που ε, προσλάμβαναν γυναίκες. Και έτσι βελτιώθηκε πολύ σημαντικά και πολύ γρήγορα η κατάσταση. Για την ανάλυση τώρα στην οποία καταλήξαμε σε επίπεδο βρέμη, θα πρέπει να πω ότι το πρόβλημα τουλάχιστον για τη Γερμανία δεν ήταν τόσο πολύ χώρων ή υποδομών υποδοχή παιδιών, παιδικών σταθμών και ούτω καθεξής, αλλά περισσότερο ε, η παγωγή των γυναικών, η προτίμηση των γυναικών σε ορισμένες συγκεκριμένες ε, κατηγορίες επαγγελμάτων κατά 90% σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελμάτων που είναι και κακοπληρωμένες και αποτελούν ε, την ε, πόρτα για την φτώχεια των γυναικών, την πύλη μάλλον για την φτώχεια των γυναικών και εκεί θα πρέπει να κοιτάξουμε να ρίξουμε τους φραγμούς που ξεχωρίζουν άνδρες και γυναίκες. Αυτή λοιπόν ε, η γνώση την οποία συλλέγουμε από τις πολύ ενδιαφέρουσες ε, ε, παρουσιάσεις και ελπίζω να μας στείλετε και τις διαφάνειές σας, το αντίγραφο δηλαδή, γιατί ήταν εξαιρετικές οι παρουσιάσεις σας. Δεν θα για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω. Ήταν πραγματικά πολύ καλά και σημαντικά τα αποτελέσματα και για μας. Και θα πρέπει να σημειώσουμε ότι και η Επιτροπή στη δουλειά της και τις προτάσεις της και στη διατύπωση των προτάσεων, όχι δηλαδή στην ουσία μόνο, αλλά και στη διατύπωση, θα πρέπει να δείξει θάρρος και να πει ότι η διάσταση του φίλου θα πρέπει να ενσηματώνεται υποχρεωτικά, γιατί είναι υποχρέωση των κρατών μελών στην κάθε πολιτική. Πρέπει να αξιοποιείται κάθε δυνατότητα τεχνικής υποστήριξη από τον έναν προς τον άλλον για τη βελτίωση αυτής της διάστασης ε, σε όλα τα κράτη-μέλη για την οικονομική υποστήριξη. 100% τεχνική βοήθεια σημαίνει ότι αρχεί να έχει κανείς μια ιδέα. Άμα έχουμε την ιδέα υπάρχει πολιτική βούληση από πίσω και προχωρούμε στην υλοποίηση. Η δε ομάδα εργασίας θα πρέπει να έχει στο δυνατόν μεγαλύτερη, μεγαλύτερο απόϊχο της εργασίας της, περισσότερα αποτελέσματα δηλαδή. Και θα ήθελα για άλλη μια φορά να πω ότι κατέστη φέσαι από την παρουσίαση για την ομάδα εργασία ότι προσθέτει ακριβώς αυτή, προσφέρει ακριβώ αυτή την προσθέμενη αξία η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τον κανονισμό. Ζητάει από τα κράτη-μέλη να δίνουν στατιστικέ για τη διάσταση των φύλων στον χώρο εργασία, στην επιχειρηματική δραστηριότητα κτλ. Με βάση τα οποία μπορούν να μπορούμε να καταλήξουμε σε αποτελέσματα που θα μα επιτρέψουν να χαράξουμε πολιτική και σε άλλου τομεί, δηλαδή πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Δηλαδή δίνουμε αυτό το πουσάρισμα στην γυναίκα γυναίκα έτσι ώστε και να ξεφύγει από τη φτώχεια και να βγει από την ανεργία. Δηλαδή όλα αυτά ε, τα πολλαπλά αποτελέσματα που αποτελούν την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία και που πιστεύω αξίζει τον κόπο για να τα εξασφαλίσουμε να είμαστε πιο αυστηροί. Μέσω αυτή τη προσπάθεια θα διευκολυνθεί ακόμη περισσότερο η υλοποίηση των στόχων του 2020, θα κερδίσουμε τα μάλα. Υπάρχουν ζητήματα βέβαια και τεχνικά ε, κατάρτισης, ενημέρωσης, διοικητικά, γραφειοκρατικά, αλλά πάνω απ' όλα η πολιτική βούληση. Ευχαριστώ. Okay, Mr. Ε, Kelly, please. Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομο. With... Συμφωνώ απόλυτα με όλη αυτή την ε, ιδέα της ενσωμάτωσης διάστασης του φύλου και ε, πράγματι, αν θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους ε, για το 2020 και αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στον κόσμο, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλο μας το δυναμικό, όχι μόνο των πόρων ε, των οικονομικών αλλά και των ανθρώπινων πόρων, γυναικείων και ανδρικών. Οπότε πρέπει να ενισχύσουμε τις γυναίκες ακόμη περισσότερο και ειδικότερα σε ε, συγκεκριμένες περιφέρειες. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να υπάρχουν, ε, να ενισχυθούν οι γυναίκες εκεί που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, όχι γενικώ και αορίστιος. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο, ας πούμε, στον κατασκευαστικό τομέα οι γυναίκες θέλουν να έχουν ίσες ευκαιρίες με τους άντρες και να σηκώνουν βάρη, να χρησιμοποιούν φτιάρια ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν ε, άλλοι τομείς όπου υπάρχει τεράστια ανάγκη για παράδειγμα στις επιχειρήσεις, επιχειρηματικότητα. Αναφέρθηκαν μάλιστα, αναφέρθηκαν οι, αναφέρθηκε η Lehman Brothers ε, ως ε, ανέκδοτο. Γιατί νομίζω ότι στις επιχειρήσεις Υπάρχει ένα τελάς, τεράστιο κενό και το έχω δει και στην Ιρλανδία. Αν δεν είχαμε τόσο πολλούς ε, άνδρες ε, στα διοικητικά συμβούλια δεν θα είχαμε τόσο μεγάλο πρόβλημα. Και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει μεγάλη προσπάθεια περισσότερες γυναίκες ε, να αναλάβουν αυτές τις θέσεις και ειδικότερα να συμμετέχουν στο επιχειρήν. Ε, η, εκείνη, η, βραβευμένη με το ε, Ιρλανδικό βραβείο καινοτομία, ε, μου έστειλε χτες ένα email και μου έκανε κάποιες συστάσεις. Είναι κάτι που θα μπορούσαμε να το δούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ισότητα των φύλων προσπαθούμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερε γυναίκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διαφορετικά, αν ε, κυριαρχούσαν οι άντρε, θα ήταν τελείω διαφορετικά τα πράγματα. Αυτό πρέπει να ισχύει και στι πολιτικέ και σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο. Και αν το κάνουμε αυτό, νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια κανονική κοινωνία στην οποία άνδρες και γυναίκες ε, συμμετέχουν εξίσου ε, στην επίτευξη των στόχων ε, για την της Ευρώπης 2020. Ε, έτσι μόνο μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει μια πραγματική ισότητα μεταξύ των φίλων. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λούκα Σεγεύσκια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ χαίρομαι για αυτήν την συζήτηση τη σημερινή βλέπουμε καθαρά ότι υπάρχει το πρόβλημα σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και όλα όσα λέμε εδώ είναι πολύ σημαντικά τώρα. Δεν εμφανίζεται τόσο στην αγορά εργασίας οι γυναίκες, δεν εκμεταλλευόμαστε τις δυνατότητες τους. Ε, ακόμα και στις πιο φτωχές περιοχές υπάρχουν λιγότερες δραστηριότητες από πλευράς γυναικών. Αλλά για να δούμε. Το παράδειγμα Τώρα, αυτά τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε βέβαια μία βελτίωση της όλης καταστάσεως. Οι γυναίκες δεν είναι ότι είναι λιγότερο ή χειρότερα εκπαιδευμένες από τις γυναίκες με λιγότερα προσόντα, αλλά πολλές φορές ας πούμε έχουν κλασικής κατεύθυνσης σπουδές παραπρακτικής και γι' αυτό ίσως πληρώνονται λιγότερο. Χωρίς αυτό οι δραστηριότητες των γυναικών θα μπορούσαν να αλλάξουν μπορούμε να πούμε γιατί ακολουθούν ορισμένα στερεότυπα βέβαια όχι παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σκέφτεται παντού ότι η γυναίκα είναι στις, στο σπίτι της παραμένει αλλά ίσως αυτό συμβαίνει μάλλον συμβαίνει περισσότερο στις αγροτικές περιοχές και τώρα πώς θα συνδυαστεί μετά η επαγγελματική με την ιδιωτική ζωή μιας γυναίκας. Όσες γυναίκες έχουν παιδιά θα πρέπει να ασχοληθούν και με τα παιδιά αυτά, να τα μεγαλώσουν και αναρωτιούνται όλοι και οι ίδιες βέβαια πού θα μείνουν τα παιδιά όταν πάνε στη δουλειά εκείνες. Ε, σε αυτό δεν αναφερόμαστε και τόσο πολύ δυστυχώς. Και οι εργοδότες δεν ρωτάνε τις γυναίκες, τους ε, άνδρες ε, τι γίνεται εσείς θα τα φροντίσετε. Εδώ λοιπόν ε, αυτές οι ερωτήσεις σαν αποτελούν ένα ταμπού κοινωνικό ακόμα και το επίπεδο αμοιβών μισθών. Δεν υπάρχουν χώρες όπου για τις ίδιες εργασίες, για την ίδια εργασία ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες να αμείβονται το ίδιο και εκεί το δέχονται κοινωνικά και πολιτικά έτσι απλά. Αντίθετα θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Χωρίς αυτή την ευαισθητοποίηση δεν μπορούμε να καταστήσουμε ενέργειες περισσότερο. Τι ζάζεται να, τους, να τις λάβουμε υπόψη μας και κοινωνικά ε, και σε κάθε τομέα στην καθημερινή του ζωή. Και ακόμα να προσθέσω ένα παράδειγμα που δεν αφέρθηκε σήμερα, αλλά είναι ουσιαστικό βάσει της πείρας που διαθέτω εγώ. Οι γυναίκες θα έπρεπε να υποστηρίζονται περισσότερο μεταξύ τους. Εάν μια γυναίκα είναι διευθυντικός τέλεχος, βλέπουμε τελικά ότι της αρέσει, προτιμάει δηλαδή να συνεργάζεται με άνδρες. Τι γίνεται και σε ένα διαγωνισμό αν πετύχουν, αν έχουν την ίδια στο πούμε έτσι βαθμολογία άνδρες και γυναίκες προτιμούν να προσλάβουν τον άνδρα. Δεν έχω συγκεκριμένες στατιστικές αλλά βλέπουμε ότι και το ποσοστό που λαμβάνουν ας πούμε που βοηθούνται Επιχωρητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι άνδρες υπερισχύων χωρίς λοιπόν να έχουμε μια πολιτική βούληση δεν θα έχουμε στη διάθεσή μας το δυναμικό το γυναικείο θα πάει χαμένο και αυτό είναι κρίμα διάφορες συζητήσεις τώρα πολιτικές πιέσεις Όλα αυτά θα πρέπει να συνεχίσουν, αλλά ταυτόχρονα να ασκηθεί και πίεση, όπως είπαμε, για υπέρ των γυναικών. και υπάρχει δυσκολία στην κατανομή εξίσου των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μεταξύ ανδρών και γυναικών βέβαια γιατί πάνε τα χρήματα αυτά στα καλύτερα προγράμματα. Αλλά όπως είπε η κυρία Σρέντερ θα πρέπει να δούμε πού θα πάνε αυτά τα κονδύλια όπως στη Βρέμη ε, που ορισμένες εταιρείε ανταμείφθηκαν ακριβώς επειδή προτιμούσαν τη γενική εργασία. Θα πρέπει να τα ε, εκμεταλλευτούμε αυτά. Ευχαριστώ. Ε, thank you very much. Frau Krell, bitte. Ευχαριστώ κύριε Κρέλ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα συνεχίσω βεβαίως τα όσα είπε η Ελίζαμπετ Σρόντερ νωρίτερα. Ομολογώ ότι 22 χρόνια έχουμε στο Κοινοβούλιο δεν βλέπω να έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα. Κάθε δύο-τρία χρόνια η Επιτροπή των Περιφερειακών Υποθέσεων συζητάει την κατάσταση τη ενσωμάτωση των φίλων, τη ισότητα των ευκαιριών για άνδρε και γυναίκε. Και όταν έρχεται η ώρα για συγκεκριμένα παραδείγματα, μάλλον συγκεκριμένα μέτρα, η πλειοψηφία συνήθω αποτραβιέται και δεν τα υποστηρίζει. Έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Έχουμε πολλούς αγώνες ήδη διεξαγάγει για την ενσωμάτωση της διάστασης των φύλων στην περιφερειακή πολιτική, την πολιτική συνοχής. Εγώ έχω αναλάβει ήδη στο παρελθόν τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συγγήτρια ε, και είχαμε πολύ μεγάλη, μεγάλο κόπο να εξασφαλίσουμε αρμοδιότητες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απορρίπτει λειτουργικά προγράμματα όταν δεν ήταν επαρκής η ε, λήψη υπόψη τη διάσταση των φύλων ε, στα προγράμματα αυτά. Αλλά βέβαια η Επιτροπή δεν το έκανε ποτέ αυτό. Τώρα μα λέτε ότι να, υπάρχουν καλά παραδείγματα. Η Ισπανία. Ωραία. Πολύ καλά. Ωραίο παράδειγμα. Αλλά που δεν πάνε καλά τα πράγματα δεν μα λέτε. Μόνο το θετικά πρώτα προθέτε να μα προβάλλετε. Βλέπουμε ότι στη Γερμανία Φερρυπίν δεν λειτουργεί καθόλου η διάσταση των φύλων και φαντάζομαι ότι και αλλού υπάρχουν προβλήματα. Εάν δεν τα συζητήσουμε αυτά, θα πάμε πουθενά. Και ε, βλέπω ότι δεν υπάρχει και ζήτημα απόρριψης των λειτουργικών προγραμμάτων. Άρα, εάν ε, τώρα από το 2011 φτάσουμε στο 2015 για να συστούμε τα ίδια πράγματα και να ακούμε κάποια θετικά παραδείγματα, ε, επειδή κάποιοι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι και συνειδητοποιημένοι και με προσοχή ε, και σεβασμό ε, ενσωματώνουν τη διάσταση των φίλων στα προγράμματά τους, δεν νομίζω ότι έχουμε κάνει τίποτα. Θα πρέπει να επιδείξουμε έξω από τη σκιά μας, όπως λέμε, να χτυπήσουμε, το, να θέσουμε το δάχτυλο επί το τύπο των ύλων και να δούμε οι αρμοδιότητες αυτές που έχει η Επιτροπή να σταματήσουν να είναι απλώς ωραία λόγια και να μεταφραστούν σε πράξεις. Γιατί έτσι πια δεν πάει άλλο. Vielen Dank. Δυστυχώς... δεν έχω το λόγο να δώσω πάλι, δεν έχω το χρόνο να δώσω πάλι το λόγο στους ε, εμπειρογνώμονες μας. Ίσως για ένα λεπτό αν έχετε να κάνετε μια σύντομη δήλωση, μια σύντομη παρατήρηση. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με όλους όσοι έλαβαν το λόγο και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε ιδιαίτερα ε, την ε, εφαρμογή της διάστασης του φύλου, δηλαδή να δούμε με μεγαλύτερη σοβαρότητα την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου για να υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση και στα, και στα 27 κράτη-μέλη με αυτή την αυτό παράγοντα. Πλέον έχει έρθει η ώρα και γι' αυτό ακριβώς έχουμε εμείς ξεκινήσει με το σχέδιο αυτό Winner 8 δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στη δεκαετία του 80 να κάνουμε συζητήσει, συστήσει έχουν γίνει. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε εμπειρογνώμονες, μπορούμε να σα στηρίξουμε. Να παρακαλώ κι εσείς. Ναι, συμμερίζομαι απόλυτο στα όσα είπε η συνάδελφο και ήρθε πια η ώρα, πιστεύω, τώρα που θα γίνει αναθεώρηση πολιτική συνοχή ε, για την υλοποίηση μετά το 2013. Είναι η στιγμή, όπω έλεγα, να συμπεριληφθεί τυπικά, επισήμω δηλαδή μέσα στη διαδικασία, και είμαι βεβαία ότι και ο μηχανισμός και ο χώρος είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν. Χρειάζεται να υπάρχουν σαφείς θέσει στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων γιατί θέλουμε να κάνουμε τη διαδικασία αυτή. Υπάρχει μεγάλο πλούτο εμπειρία, γνώσει, βέλτιστε πρακτικέ από άλλα σχέδια και ελπίζω ότι θα ληφθούν υπόψη. Σα ευχαριστώ, λέει Εκ μέρους της Επιτροπής μας ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, παρισταμένους για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα περάσω τώρα στο τελευταίο σημείο της ημερησίας διάταξης που αφορά τα διάφορα και θα ήθελα να σας ενημερώσω για κάποιες αποφάσεις που έλαβαν ε, οι συντονιστές των πολιτικών ομάδων όσον αφορά την ανάθεση εκθέσεων και γνωμοδοτήσεων. Η γνωμοδοτήση για την κινητοποίηση του Ταμείου Φυσικών Καταστροφών Σλοβενία Τσεχική Δημοκρατία του 2010. Πρέπει να ψηφίσει, το αναλαμβάνει η Πρόεδρο θα πρέπει να γίνει ψηφοφορία τον Ιούνιο. Αμοιβαία, διαδικασία αμοιβαία αξιολόγηση. Η ομάδα θα ενημερώσει τη γραμματεία εάν ενδιαφέρεται. Εκθέσεις είναι. Οι συντονιστέ αντέλαξαν ε, απόψεις προς την ανάγκη για μια στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μεσογειακή, ε, στη Μεσογειακή ε, Λεκάνη. Επίση, δεν υπήρξαν προτάσει συγκεκριμένε. Οι πράσινοι θα αναδιατυπώσουν τι προτάσει του για μελλοντική συνεδρία. Στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα διατύπωσε μία πρόταση για τις άκρως απομακρυσμένε περιφέρειες, πολιτική συνοχής, δημόσιες προμήθειες που θα, θα εξετάσουν οι συντονιστέ. Το ίδιο που θα, επιβάλλουν θα υποβάλουν τις προτάσεις στη Γραμματεία για η έγκριση της προσεχής συνεδρίας. Νομοθετικό πακέτο για την πολιτική συνοχή μετά το 2012 θα ληφθεί απόφαση στην προσεχή συνεδρίαση της προσεχούς εβδομάδας. Συντονιστές θα συνεδριάσουν την επόμενη φορά στις 9 Μαΐου, 7 το βράδυ στο Στρασβούργο. Ευχαριστώ πολύ. Πέρα στη συνεδρία σας.